We start the meeting. Πάμε. Ξεκινάμε τη συνεδρίασή μας. Έγκριση μέλησης διάταξης πρώτα. Το θέμα της ε, αίτησης Μωρή Δικρού θα αναβληθεί η Επιτροφή Προϋπολογισμών θα ψηφίσει στις 31 Μαρτίου για το θέμα αυτό και επομένως δεν θα υπάρξει επίπτωση από την, την ε, αναβολή. Μπορούμε να δεχτούμε λοιπόν την μέση διαδάξη με αυτή την τροποποίηση. Για τις διερμηνευτικές διευκολύνσεις όλες τις γλώσσες τις έχουμε, αλλά τα κροατικά και τα μαλτέζικα Και σε σχέση με την πρόταση τροποποίηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων με τη δυνατότητα να υπάρξει προχρηματοδότηση με την πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων. Ναι, θα πρέπει να φέρουμε την ε, προθεσμία της τροπολογίας την 5η 12 Μαρτίου ώστε να έχουμε επαρκή χρόνο για την μετάφραση των τροπολογιών και για τις συναντήσεις των σκιωδών εισηγητών. Βέβαια, 16 Απριλίου θα πρέπει να ψηφίσουμε ούτως ή άλλως. Πάμε τώρα στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων, σημείο 3 της ημερησίας διάταξης. Και δίνω το λόγο στην κυρία Γιάσλοβιέσκα. Καλημέρα σας, σας ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, μετά από την κρίση υπήρξε σημαντική πτώση επενδύσεων στην Ευρώπη έναντι του 2007. Το 2007 ήταν έτος κορύφωσης για τις επενδύσεις. Το χάσμα επενδύσεων έχει οδηγήσει και σε μείωση απασχόλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση. και γι' αυτό το λόγο είναι πολύ δύσκολο να επιτύχουμε τους στόχους του, της Ευρώπης 2020 όταν υποτίθεται ότι η απασχολησιμότητα θα φτάσει στο 75%. Οι νέοι είναι τα κύρια θύματα των υψηλών επίπεδων ανεργίας. Επιζητούμε να βρούμε λύσεις σε αυτό το πρόβλημα. Δυστυχώς, τα διάφορα εργαλεία τα οποία έχουν προταθεί μέχρι στιγμής για τον στόχο αυτό είναι ελλειπή σε ό,τι αφορά την αποτελεσματικότητά τους. Εξακολουθεί να είναι υψηλή λοιπόν η ανεργία. Εξακολουθούμε να έχουμε ανάγκη να ενισχύσουμε τις επιχειρήσεις ώστε να μπορέσει να υπάρξει περισσότερη επένδυση και περισσότερη απασχόληση. Τα υψηλά επίπεδα ανεργίας είναι το άμεσο αποτέλεσμα της έλλειψης επενδύσεων. Γι' αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατηγικών Επενδύσεων είναι απαραίτητο. 315 δισεκατομμύρια ευρώ στα επόμενα τρία χρόνια, μέσα σε τρία χρόνια, που υπολογίζεται ότι θα δημιουργήσουν 1,3 εκατομμύρια νέες θέσεις απασχόλησης. Και επομένως θα υπάρξει ένα θετικό άμεσο αποτέλεσμα στα επίπεδα απασχόλησης. Ο κύριος στόχος μας εδώ είναι να δώσουμε μια ε, ισχυρή όθηση στην οικονομία ώστε να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και να διατηρηθούν αυτές οι οποίες ήδη υφίστανται. Το Ταμείο Επενδύσεων, το EFSI, θα λειτουργήσει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι επιχειρήσεις θα δείξουν ενδιαφέρον για να χρησιμοποιήσουν τα κονδύλια του Ταμείου και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμβάλλουν στο εγχείρημα αυτό. Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να δείξουν και μία πολιτική η οποία είναι προδραστική και να εξασφαλίσουν ότι οι δυνητικά εργαζόμενοι έχουν τις απαραίτητες δεξιώσεις τις οποίες απαιτούν οι επιχείρησεις που θα μπορούσαν να τους προσλάβουν. Θα εστιάσει ιδιαίτερα <clears throat> αυτό το νέο ταμείο στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση που γνωρίζουμε είναι το 95% όλων των επιχειρήσεων και δίνουν απασχόληση σε πάνω από 90 εκατομμύρια ατόμων. Τα τελευταία χρόνια 85% των νέων θέσεων απασχόλησης έχουν δημιουργηθεί από τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχουν πραγματικοί κίνητρα για τα κράτη-μέλη για να λάβουν υπόψη τους τη δυνατότητα χρηματοδότησης από το EFSI, από το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Όταν όμως η Κομισιόν εξετάζει την ικανότητα των κρατών μελών να ικανοποιήσουν τις προϋποθέσεις του Συμφώνου Σταθερότητος και Ανάπτυξης, οι επενδύσει οι οποίε εμπίπτουν στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων θα πρέπει να ξερούνται από τον υπολογισμό. Θα πρέπει λοιπόν ο στόχο να είναι να βελτιώσουμε την οικονομική κατάσταση στα κράτη-μέλη, να δημιουργηθούν θέσει απασχόληση σε μακροχρόνιο επίπεδο. Και όπω τόνισα, το κριτήριο για την επιλογή σχεδίων και προγραμμάτων θα πρέπει να περιλαμβάνει την δυνατότητα, την ικανότητα αυτών των σχεδίων μάλλον να δημιουργήσουν μόνιμες θέσεις εργασίας βιώσιμες θέσεις εργασίας και η δημιουργία θέσεων εργασίας από, το, από τη χρηματοδότηση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων θα πρέπει να τη χάνει συνεχούς εποπτείας σε, ιδιαίτερα για τις περιοχές που έχουν το υψηλότερο επίπεδο Ανεργία, Θα έρθω σε επαφή με τους εισηγητές και οδηγητέ στο Στρασβούργο και προσβλέπω στην ανταλλαγή απόψεων μαζί τους. Και φυσικά και στη σημερινή συζήτηση. Ελπίζω ότι όλα αυτά θα οδηγήσουν σε μια καλή έκθεση. Και απλώ θέλω να πω ότι θα εξετάσουμε την έκθεση αυτή μονάχα από την οπτική γωνία της δικής μας αρμοδιότητας, γιατί είμαστε Επιτροπή Απασχόλησης και μόνο με αυτό το πρίσμα θα δούμε αυτή την έκθεση. Η Μαρία Χαρδεζίκης από το SND, από Σοσιαλιστές. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα συγχαρητήρια στον εισηγητή γιατί πράγματι έκανε πολύ καλή δουλειά. Φυσικά και θα συνεργαστούμε μαζί σας, θα χτίσουμε και εμείς πάνω στη δικιά σας ε, τη δουλειά, Δανούτα. Αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων πρέπει να σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε τα μέσα αυτά να γίνουν ένα ισχυρό εργαλείο για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και μάλιστα ποιότητας. Αυτό είναι βασικός στόχος για τη δικιά μας την ομάδα. Πιστεύουμε ότι ο τρόπος για να γίνει αυτό εφικτό απαιτεί να πούμε με σαφήνεια ότι η δημιουργία απασχόλησης και μάλιστα τα αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα για το Ταμείο αυτό. Και αυτό πρέπει να φανεί στις κατευθυντήριες γραμμές που θα καθορίσει το steering board ε, του Ταμείου αυτού. Πρέπει επίσης να φανεί και στα κριτήρια επιλογής των έργων από την Επιτροπή Επενδύσεων. Γι' αυτό και πιστεύουμε ότι οι εμπειρογνώμονες πρέπει να επιλεγούν με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι εμπειρογνώμονες όχι μόνο στα οικονομικά των έργων, αλλά και όσον αφορά την πραγματικότητα των κλάδων τα οράματα που έχει ο κλάδος και τις ε, δυνατότητες που έχει να προσφέρει νέες θέσεις απασχόλησης. Για τις επενδυτικές πλατφόρμες τώρα αποτελεί ένα νέο εργαλείο αυτό που αναφέρεται στον κανονισμό και πιστεύουμε ότι αυτές οι επενδυτικές πλατφόρμες μπορεί να είναι βέβαια από πολλές χώρες και διαφορετικές, αλλά μπορεί να είναι και θεματικές πλατφόρμες. Όπως πάντως και να έχει το πράγμα, πιστεύω ότι οι πλατφόρμες αυτές πρέπει να σχεδιαστούν με τέτοιο τρόπο ώστε να αποτελέσουν το χώρο όπου επενδυτικές εταιρείες να μπορούν να συναντιούνται με όλους τους υπόλοιπους θεσμούς και παράγοντες ώστε να συζητούν τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης από κοινού. Μπορεί να αποτελέσει δηλαδή μια τέτοια πλατφόρμα ένα πολύ καλό κέντρο για καινοτομία και για δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Όλα αυτές οι ε, ενέργειες, οι δράσεις είναι επιλέξιμες από ό,τι φαίνεται. Και μπορώ να σας δώσω και ένα παράδειγμα. Αν έχουμε επενδυτική πλατφόρμα για την ε, απόδοση ενέργειας, μπορούμε να βάλουμε μαζί τις επιχειρήσεις, ερευνητικά κέντρα και την κατάρτιση. Οπότε η καινοτομία να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης ποιότητας. Δεύτερον, όπως γνωρίζετε, το επενδυτικό αυτό ταμείο πρέπει να κάνει και κοινωνικές επενδύσεις και είναι σημαντικό γιατί πρέπει να επενδύσουμε στην εκπαίδευση, στη μόρφωση, δηλαδή στην κατάρτιση και να δημιουργήσουμε και κοινωνικές διευκολύνσεις, κοινωνικό εξοπλισμό για την ε, παιδική μέρημνα, την οικογενειακή μέρημνα, κάτι που έχει να κάνει όλος ιδιαίτερως με τις γυναίκες αλλά και με τους άντρες για να συμφιλιώσουν την ε, οικογενειακή με την επαγγελματική ζωή. Τέλος πιστεύουμε ότι το επενδυτικό αυτό ταμείο πρέπει να δώσει ιδιαίτερη προσοχή στις περιφέρειες και τις χώρες εκείνες που έχουν περισσότερο πληγή από την κρίση. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σας ευχαριστώ. Γερικέ, από το ECR. Ja, <laughs> ich möchte im Namen von Ulrike Εξ ονόματος της Ουλίκη Τρεμπίσιους θέλω να λάβω το λόγο, δυστυχώς δεν μπόρεσε να είναι παρούσα η Ουλρίκε. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο για το έργο του σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων, το οποίο είναι ιδιαίτερα πλήρε. Εμεί θέλουμε να τονίσουμε ιδιαίτερα τη σημασία των διαρθρωτικών αλλαγών και του ελέγχου ποιότητα των ε, εγχειρημάτων. Υπάρχουν όμω περιπτώσει που δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε από, απόλυτα, όπως τη χάρη η εστίαση σε επιχειρήσεις οι οποίες βασίζονται σε ενέργεια συνδικαλιστικών οργανώσεων. Δεν θέλουμε να έχουμε ε, επιλογή προγραμμάτων τα οποία δεν θα συνάδουν με τους στόχους του ε, Ταμείου. Θεωρούμε ότι θα πρέπει να περιορίσουμε την γνωμοδότησή μας, όπως ζητήθηκε και από την ΕΚΟΝ και από την Επιτροπή Προϋπολογισμών, να περιορίσουμε την ε, ε, παρέμβασή μας με τη γνωμοδότησή μας και να τονίσουμε ιδιαίτερα ότι ιδίω για την αγορά εργασίας είναι απαραίτητε μεταρρυθμίσεις ιδίω στη Νότια Ευρώπη αλλά επίση και μεταρρυθμίσει στον τραπεζικό τομέα, ο οποίο αντιμετωπίζει μεγάλη δυσκολία στην παροχή χρηματοδότηση. Θα πρέπει η συζήτησή μα λοιπόν να εστιάσει στα θέματα αυτά. Ευχαριστώ. Okay. Σα ευχαριστώ, Λεπρόεδρο, και τώρα δώσουμε το λόγο στην Άλντε. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, πρώτα πρώτα να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το έργο της. Έχουμε πάρα πολλά κοινά μέσα στο ίδιο μικρό οπότε και μπορούμε να συμφωνήσουμε όσον αφορά το ότι πρέπει να εστιαστεί η προσοχή ε, στην υπόθεση της ε, απασχόλησης και ότι θα πρέπει να είναι θέμα προτεραιότητας επίσης ε, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και για την αποσύνδεση των πόρων αυτών όσον αφορά την υπολογή, τον υπολογισμό των ελλημάτων και των κενών στον προϋπολογισμό επί της ουσίας τώρα από πλευράς απασχόλησης και κοινωνικών υποθέσεων. Θεωρούμε ότι έχουμε δύο δυνατές ερμηνείες του προγράμματος Juncker. Πρώτα-πρώτα, πρόκειται να υπάρχουν για άλλε χρηματοδοτήσει, ώστε να εξοικονομήσουμε την Ευρώπη, να την κάνουμε πιο ανταγωνιστική, πιο παραγωγική. Και υπάρχει άλλη μια ερμηνεία που υποστηρίζουμε εμεί ότι έχουμε αυτού του είδους το κατεπήγον πρόγραμμα των τριών ετών γιατί θα πρέπει να δούμε ε, το πώς θα αντιμετωπίσουμε ε, αυτή την, την τρομερή ανεργία, την ε, τρομερή διάλυση της κοινωνικής συνοχής που υποφέρει ένα μέρος της Ευρώπης. Επομένως, θεωρούμε ότι αυτό είναι ένα ηλεκτροσόκο το και δεν είναι ακόμα ένα ταμείο, ακόμα κάποια χρήματα. Αυτό είναι το σχέδιο Juncker. Αλλιώ νομίζω ότι θα χάσουμε την αξιοπιστία έναντι ε, του κόσμου. Επομένως πρόκειται για σχέδιο εκτάκτου ανάγκης και γι' αυτό και εγκρίθηκε αυτό το σχέδιο Juncker. Οπότε δεν μπορούμε να συμφωνήσουμε με όσα είπε η συγγήτρια και θέλω να σταθώ σε κάποια σημεία. Ας μην διευθυνθεί ότι την επικρίνω. Απλώς θέλω να βελτιώσω το ήδη αξιολογοκείμενο. κείμενο. Πρώτα-πρώτα θα πρέπει να γίνει κάποια αξιολόγηση και με κριτήρια αξιολόγησης κοινωνικής πολιτικής να δούμε τι θα γίνει με την Τράπεζα Επενδύσεων και με τα λοιπά ταμεία. να επικεντρώσουμε την προσοχή μας στις ΜΜΕ και επίσης περισσότερο κατά περιφέρειες και λιγότερο κατά χώρες να δούμε πώς θα κατευθύνουμε επενδύσεις εκεί σε κάποιους θύλακες ανεργίες που πολλές φορές ξεπερνούν τα σύνορα. Επομένως, εκεί θα πρέπει να κεντρώσουμε την προσοχή μας. Εκεί είναι το διακύβευμα δεν είναι το να έχουμε περισσότερες ανισότητες και ανισορροπίες. Επίσης θα πρέπει το Κοινοβούλιο να τοποθετηθεί με ε, κάποιο είδου τελική έγκριση ε, συνεργασία όσον αφορά τα βασικά κριτήρια, τα εφαρμοστικά, τα οποία ξέρουμε ότι θα πρετανεύσουν για το EFSI. Γιατί το θέμα δεν είναι μόνο το κοινοβούλιο το κοινοβούλιο το οποίο θα πρέπει να μην αναλώνεται σε λαϊκισμούς και δημαγωγίες ούτε είναι κάποιο είδους ε, dealing room κάποιες τράπεζες. Είμαστε εδώ για να δούμε το πώς θα πιάσουν τόπο αυτές οι επενδύσεις όσον αφορά την κοινωνική συνοχή και την ε, ανεργία, για την απασχόληση. Άρα το Κοινοβούλιο θα πρέπει να συμμεταξει θα πρέπει να εμπλακεί σε αυτήν όλη την προβληματική για στο ευρύτερο πλαίσιο ενίσχυσης. Επομένως θα πρέπει να βοηθήσουμε για να δούμε πώς θα προχωρήσει ε, αυτή η υπόθεση στα πλαίσια του προγράμματος ε, Juncker για την παιδεία, για τις κοινωνικές υποδομές, γιατί θα πρέπει να πιάσουν τόπο αυτά τα χρήματα. Και έτσι νομίζω ότι σε τρία χρόνια θα μπορέσουμε να πετύχουμε τους κοινωνικο-οικονομικούς στόχους αυτού του είδους του κατεπίδοντος προγράμματος. Ευχαριστώ. Η ε, Πρόεδρος. Για την ΚΟΕ, ο Πατρίκ Λιερίκ. Αλλά όμως δεν είναι εδώ. Δεν θέλετε το λόγο, ε. Καλώς. Εντάξει ούτε κάποιος άλλος από την ομάδα σας. Ωραία. Τζιν Λάμπερτ. Από τους πράσινους. Παρακαλώ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Μιλάω εκ μέρους της Μόνικα Βάνα, της Κιόδους, συγκητριάς μας, που δεν μπορεί δυστυχώς να είναι εδώ σήμερα. Θα σας μεταφέρω τις απόψεις της, δηλαδή, αλλά και τις απόψεις της ομάδας μας. Πρώτα απ' όλα ευχαριστούμε πολύ την εισηγήτρια έκανε πολλή δουλειά που αποτελεί μια πολύ καλή βάση για να προχωρήσουμε σε αυτό το θέμα. Στον κανονισμό εμείς θέλουμε να δούμε κάτι δεσμευτικό σε σχέση με τους στόχους του 2020, δηλαδή μείωση της στόχιας, ισότητα μεταξύ των δύο φύλων, κλιματική αλλαγή, αντιμετώπιση της δηλαδή, διαφορετικά ταμεία κλπ. κλπ που τα διευθυντικά ταμεία πρέπει να αποτελούν εργαλείο για επενδύσεις. Συμφωνούμε ότι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης ποιότητας πρέπει να έχει πρωταρχική θέση επίσης. Θέλουμε επίσης όλα αυτά να συνδυαστούν και με περιφέρειες που έχουν πολύ ψηλά επίπεδα ανεργίας και φτώχειας. Στην αρχική μελέτη του ILO είχε αναφερθεί αυτό, ότι δηλαδή η επιτυχία του επενδυτικού αυτού ταμείου θα εξαρτηθεί από το αν τελικά θα δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης ποιότητας στις περιφέρειες που πλήττονται περισσότερο από την κρίση και από την φτώχεια. Το Διεθνές Γραφείο Εργασίας το είπε αυτό δηλαδή. Και πριν από λίγο κατά είπε και ο συνάδελφος από το Άλντε, από τους Φιλεύθερους. Κάτι τώρα για τη δημοκρατική λογοδοσία όμως του ταμείου αυτού, των επενδύσεων δεν αναφέρεται συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών, των κοινωνικών εταίρων. Δεν υπάρχει τίποτα τέτοιο που να προβλέπετε. Μιλάμε για πλατφόρμες. Πρέπει να υπάρξει μια πλατφόρμα για την κοινωνία των πολιτών. Άκουσα και τα σχόλια για την ευρεία ε, εκπροσώπηση στην, στην Επενδυτική Επιτροπή αυτή δηλαδή που θα αποφασίζει. Όντως πρέπει όπως είπε και κάποιος νωρίτερα να υπάρξει και κοινωνική διάσταση, δηλαδή οι επενδύσεις να είναι και κοινωνικές. Μόνο τότε θα πάμε προς τη σωστή κατεύθυνση. Φυσικά και θέλουμε και εμείς τις επόμενες εβδομάδες να συνεργαστούμε ώστε το επενδυτικό αυτό πρόγραμμα να πάει προς τη σωστή κατεύθυνση και ότι οι στόχοι 2020 θα συμπεριληφθούν στο επενδυτικό αυτό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Πρέπει να υπάρχει και δημοκρατική νομιμότητα. Χωρίς αυτήν δεν θα γίνει το Ταμείο αυτό που θέλουμε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Λάουρα Άγκια από το EFDD. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ευχαριστούμε για την ε, εισηγήτρια. Να σας πω κάποιες ε, σκέψεις μου. Εδώ κάποια χρόνια έχουμε στις ε, χώρες μας αυτού του είδους την ανθρωποθεσία της κρίσης και οπότε για αυτό το οποίο θέλουμε είναι να γίνει κάτι με αυτό το ταμείο, ούτω ώστε να μπορέσουμε να ανασχέσουμε τα αποτελέσματα αυτή τη κρίση. Οπότε δεν καταλαβαίνω γιατί πάντοτε μιλούμε για κάποια προγράμματα που είναι πάντοτε τόσο μακροπρόθεσμα, τόσο μακρόπνοα. Γιατί έλεγε η συνάδελφος ότι πρόκειται εδώ για ένα πρόγραμμα που έχει χαρακτήρα κατεπήγοντος. Αλλά εγώ θεωρώ ότι θα πρέπει το timing να είναι πολύ πιο άμεσο. Γιατί εδώ πέρα πάμε για αποτελέσματα μετά από μια δεκαετία. Επομένω, θέλω να σα προτείνω ότι θα πρέπει να ζητήσουμε να υπάρχει ένα άλλο timing για τις δράσεις αυτού του προγράμματο. Πάντως, ε, πάρα πολύ σωστό το ότι δίνεται η σημασία στι επενδύσει που χρησιμοποιούν απασχόληση και κατόπιν ε, θα λυθούν κάποια προβλήματα σε σχέση με την ανεργία. Επίση, θα πρέπει να δούμε τι γίνεται για κάποιε επιχειρήσει κάτω των 3.000 εργαζομένων. Θα πρέπει να συγκεκριμενοποιήσουμε περισσότερο ε, τι ισχύει για αυτέ τι επιχειρήσει οι οποίε θα είναι οι δικαιούχοι αυτών των ε, επενδύσεις και μιλούμε για τις νεοφυείς, τις ΜΜΕ, για κάποιες επιχείρησεις που ξεκινούν κάποιοι νέοι που έχουν καινοτομές ιδέες. Γιατί εγώ άκουσα να μιλούμε για υποδομές και για μεγάλα έργα και προγράμματα, μα το ενδυμικό αυτό πρόβλημα της ε, κρίσης δεν ε, λύνεται έτσι. Ε, στην πραγματική οικονομία. Δεν παρεμβαίνουμε έτσι. Γιατί μιλούμε τώρα για κάποια επιμέρους ε, κράτη εκεί όπου η οικονομία στηρίζεται στις μικρές επιχειρήσεις. Όμως αυτές οι μικρές επιχειρήσεις δεν έχουν 3 και 4 χιλιάδες ε, εργαζόμενους, έχουν 40-50 εργαζόμενους σε πάρα πολλές χώρες. Ε, αυτή είναι η πραγματικότητα και άρα εκείνη θα πρέπει να είναι κυρίως οι δικαιούχοι από αυτό το πρόγραμμα. Επίσης, διορθωτικές μεταρρυθμίσεις. Αυτό κυρίως για τις χώρες που έχουν στριμωχτεί. γιατί ζητούμε για μεταρρυθμίσεις, αλλά από την άλλη μεριά, για τις χώρες που βρίσκονται σε δυσκολία, θα πρέπει να υπάρξει κάποια όθηση στην ανασυγκρότηση της οικονομίας και στην καινοτομία. Άρα μην μας ζητάτε μόνο διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Μην κάνετε περικοπές εκεί που υπάρχουν κάποιες χρηματοδοτήσεις. Έτσι δεν είναι δυνατόν να δοθεί αυτή η ουσιαστική όθηση για αναθέρμανση της οικονομίας. Κάτι άλλο τώρα. Μιλούμε εδώ πέρα για κάποιες επενδύσεις υψηλού κινδύνου. Θα πρέπει να καταλάβουμε ότι πάρα πολύ συχνά αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να γίνει το άλμα στο κενό, να δίνεται ευκαιρία σε κάποιο ε, καλό πρόγραμμα, αλλά εδώ έχουμε και το θέμα του υψηλού κινδύνου. Οπότε θα πρέπει να δούμε πώς θα υλοποιούνται αυτά τα προγράμματα. Είπαμε για Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων, οι οποίοι θα ε, πρέπει να κάνουν την επιλογή των επιλεξίμων ε, σχεδίων και προγραμμάτων. Αλλά να μην βάλουμε τίποτα καθηγητάδες της οικονομίας, να βάλουμε κάποιους που ξέρουν την πραγματική οικονομία, την πραγματική απασχόληση. Οπότε να ε, υπάρχει βέβαια διαφάνεια, αλλά από την άλλη μεριά να μπορούν να ξέρουν την πραγματικότητα και να υπάρχουν κάποιες διακλαδώσεις, κάποιες συνέπειες τέλος πάντων όπως πρέπει αυτή της υπόθεσης. Δώστε λοιπόν τους πόρους στα κράτη-μέλη και έτσι να τροφοδοτηθεί η υπόθεση αυτού του ταμείου. Αλλά πώς θα γίνει αυτό. ας δοθούν οι εγγύησει ούτως ώστε να υπάρξει συγχρηματοδότηση και στα πλαίσια αυτού του ταμείου να έχουμε τους πόρους οι οποίοι θα βοηθήσουν τα επιλεκθέντα προγράμματα. Γιατί αλλιώς δεν μπορεί να συνεισφέρει ένα κράτος. Δεν θα υπάρξουν οι αναγκαίες εγγύησεις. Και τα πιο αξιόλογα προγράμματα τελικά είναι αυτά τα οποία είναι τα πιο απλά, τα οποία, τα οποία είναι πιο πολύ ριζωμένα στην πραγματικότητα των περιοχών του, τόπου. Ευχαριστώ κύριο Στόμας Μαν. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την εισηγήτρια για την ποιότητα της έκθεσής της. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να κάνουμε σαφές με την έκθεση αυτή ότι έχουμε μια πολύ καλή ευκαιρία να δώσουμε στην Ευρώπη μια, ένα κοινωνικό πρόσωπο όπως ε, αναφέρθηκε με επενδύσεις οι οποίες θα είναι αποτελεσματικές ε, σε κοινωνικό επίπεδο. Έχουμε δει εκπροσώπους από χώρες όπως είναι η Πορτογαλία και η Ισπανία που ξεπέρασαν το στάδιο των μεταρρυθμίσεων και μπορούν να προχωρήσουν σε ανάπτυξη. Όταν υπάρχουν οι προϋποθέσεις λοιπόν μπορεί να γίνει αυτό το πράγμα. Δεν πρέπει όμως να ε, δώσουμε και πάλι υποστήριξη σε εγχειρήματα τα οποία δεν έχουν καμία δυνατότητα να λειτουργήσουν και μονάχα ζητούν να καταναλώσουν χρήματα. Θα πρέπει να προωθήσουμε ανθρώπους οι οποίοι είναι πολιτικά ανεξάρτητοι, οι οποίοι έχουν τις απαραίτητες δεξιότητες, σχέδια, τα οποία δεν θα είναι σπατάλη χρημάτων, αλλά θα είναι ένας τρόπος με τον οποίο θα, μπορέσουν να, να, θα μπορέσουμε να επιτύχουμε οικονομική ανάπτυξη. Θα πρέπει φυσικά να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στην ε, απασχόληση. Εδώ μπορεί να έχει κανείς διαφορετικές αντιμετωπίσεις στο θέμα αυτό. Για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις όμως υπάρχουν πάρα πολλές οι οποίοι δεν έχουν πενταετή ή δεκαετή αιτήματα. Δεν ξέρουν πώς θα τα βγάλουν πέρα την επόμενη εβδομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν και το βρίσκω πολύ θετικό που βρίσκεται σε αυτή την έκθεση ότι θα πρέπει να διατηρηθούν οι υφιστάμενες θέσεις εργασίας. Είναι απαραίτητο να έχουμε ένα πλέγμα ε, μέτρο για να διατηρηθούν αυτές τις θέσεις εργασίας. Επίσης, είπε κανείς ότι θα πρέπει να δώσουμε έμφαση στις χώρες οι οποίες έχουν μεγαλύτερη ανεργία. Αλλά θα πρέπει ακόμα και σε ισχυρές οικονομικά χώρες να υποστηρίξουμε τις περιφέρειες, τις περιοχές που έχουν προβλήματα ανεργίας. Θα πρέπει λοιπόν γενικά να υπάρξει μια προτεραιοποίηση αυτών των χωρών. Στην ε, βόρεια ε, στην ε, Βόρεια Δυνανία Βεσφαλία υπάρχουν σε ορισμένε περιοχές τεράστια επίπεδα ανεργίας. Ο κόσμος πηγαίνει να δει τα μάτια ποδοσφαίρου αλλά δεν έχει τίποτα άλλο να κάνει στη ζωή του. Πρέπει λοιπόν να δώσουμε ιδιαίτερη έμφαση στις περιοχές που έχουν υψηλή ανεργία. Αυτό το συμμερίζομαι απόλυτα. Και θεωρώ επίσης σημαντικό να εμπλέξουμε και την κοινωνία των πολιτών και τους κοινωνικούς εταίρους. Είναι ένας τομέας, όπως τόνισε και η Τζιν Λάμπερτ, δεν θέλουμε να εφεύρουμε από την αρχή κάτι καινούριο, αλλά θα πρέπει να διατηρήσουμε αυτό το οποίο ισχύει ήδη. Θα πρέπει οι κοινωνικοί εταίροι να είναι αυτοί οι οποίοι θα μας δώσουν τα φώτα τους για την πολιτική απασχόληση. Νομίζω λοιπόν ότι έχουμε γενικά πολύ καλές προϋποθέσεις που πιστεύω ότι θα μπορέσει να μας οδηγήσει, παρά τις επικριτικές πρώτα φράσεις ορισμένων, θα μας οδηγήσει σε ένα κείμενο το οποίο θα είναι γενικά αποδεκτό. Ευχαριστώ, λέει πρώτο. Ο κύριος Χαμελόπες. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα θέλω να ευχαριστήσω και εγώ την εισηγήτρια για το έργο της. Έχω κάποια σχόλια. Πρώτον, το πιο σημαντικό για το επενδυτικό ταμείο είναι η αλλαγή πορείας μετά από πέντε χρόνια. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μετά από πέντε χρόνια που ακούγαμε ότι έπρεπε να έχουμε λιτότητα κτλ. Τώρα οι μακροοικονομικές πολιτικές παίρνουν το πάνω χέρι μετά από αυτή την τόσο σοβαρή κρίση που ήταν και κοινωνική αλλά και πολιτική σε κάποιες χώρες. Αυτή λοιπόν η μικρή αλλαγή πορείας, αυτό το μικρό βήμα που γίνεται και πάνω στο οποίο πολλοί από εμά βάζουμε πολλές ελπίδες, είναι ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλαγή λόγου. Τώρα στη συνέχεια βέβαια βλέπουμε και τους περιορισμούς, τους αντικειμενικούς περιορισμούς που θα έχουμε και τους οποίους πρέπει να υπογραμμίζουμε. Και ποιοι είναι αυτοί οι περιορισμοί, ναι, έχουν να κάνουν με το σχεδιασμό του επενδυτικού ταμείου και με τις δυσκολίες που έχει η ίδια η Ευρωπαϊκή Ένωση επειδή δεν διαθέτει τους κατάλληλους μηχανισμούς εξαιτία της δομής της που δεν μπορεί να έχει φρέσκο χρήμα. Επειδή οι χώρες μέλη δεν είναι διατεθειμένες μπορούν να επενδύσουν, αλλά αν δεν μπορούμε να έχουμε νέα έσοδα και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν βοηθάει, τότε πρέπει να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Με αναλογία αρκετά γενναιόδορη, με 21 δισεκατομμύρια εμείς τουλάχιστον ελπίζουμε να καταφέρουμε να έχουμε μόχλευση αλλά θα παρακολουθήσουμε τι θα γίνει στην πραγματικότητα τα επόμενα χρόνια. Έρχομαι τώρα στην επιλογή των έργων. Εκτός από τους αντικειμενικούς περιορισμούς, τι αποφασίσαμε. Τρία σχόλια έχω εδώ. Πρώτον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και όλοι συμφωνούν ότι πρέπει να υπογραμμιστεί όλος ιδιαιτέρως το θέμα έργων που έχουν να κάνουν με περιφέρειες που αντιμετωπίζουν μεγαλύτερα προβλήματα απασχόλησης και να φροντίσουμε να υπάρξουν θέσεις απασχόλησης ποιότητας μακροπρόθεσμα. Όμως με την επιλογή των έργων, εγώ βλέπω δύο πράγματα που πρέπει να έχουμε υπόψη μας. Πρώτον, το ταμείο αυτό δεν μπορεί να χρησιμεύσει για να γίνουν έργα τα οποία είχαν ήδη σχεδιαστεί από πριν. Είναι προφανές. Αν συμβεί, γιατί μπορεί να, υπάρξει, να υπάρξουν επενδύσεις από το δημόσιο ή από τον ιδιωτικό τομέα που είχαν σχεδιαστεί, είναι μία περίπτωση και άλλη είναι ε, με τα χρήματα αυτά να μην μπορούν να πετύχουν τον στόχο που αρχικά είχαν θέσει. Υπάρχει ο κίνδυνος αυτός λοιπόν να ζητηθεί συμμετοχή αυτού του ταμείου. Προσοχή. Και δεύτερον, να θυμόμαστε τους διαρθρωτικούς περιορισμούς που έχει ένα τέτοιο επενδυτικό ταμείο που θέλει κυρίως να έχει ιδιωτικά κεφάλαια. Για να χρησιμεύσει όχι για κοινά αγαθά, γιατί όπως ξέρετε είναι διαφορετική η λογική αυτών της απόδοσης, του κέρδους. Εδώ ένα τέτοιο ταμείο που έχει ιδιωτικό κεφάλαιο εννοείται ότι θα απαιτήσει επιστροφή κερδών. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό να μπορούμε να ελέγχουμε την κατάσταση, τα έργα, να ξέρουμε πώς προχωρούν τα έργα και να είμαστε πολύ προσεκτικοί στην εφαρμογή. Το είπαν και άλλοι πριν, ότι πρέπει να υπάρχει αυτός ο έλεγχος. Έγιναν πριν και κάποια σχόλια για την Ισπανία και τις διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις στην Ισπανία. Αν η Ισπανία βγει από την κρίση αλλά όχι η Ισπανή, καταλαβαίνετε ότι δεν κάνουμε κάτι καλό. Ε, και αυτό ακριβώς συμβαίνει στη χώρα μου και όχι μόνο στη δικιά μου χώρα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η Ισπανία βγαίνει από την κρίση, οι Ισπανοί όμως δεν βγαίνουν από την κρίση. Άρα εδώ έχουμε μεγάλο πρόβλημα αν αυτό συνεχίσει. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. μπάλας. Ευχαριστώ. Δεν θα μακρηγορήσω τόσο πολύ γιατί ο Πανλόπες με κάλυψε σε πολλά από αυτά που ήθελα να πω Η εισηγήτρια έχει κάνει καλή δουλειά και αποτελεί καλή βάση, όντω. Και θεωρώ ότι με ικανοποιεί. Υπάρχει μια συνένεση όσον αφορά τις επενδύσεις με μια βάση από το δημόσιο. Πριν από λίγο καιρό το είχαμε συζητήσει και όντως πιστεύω και εγώ ότι υπάρχει μια αλλαγή στον οικονομικό τρόπο σκέψης και αυτό είναι θετικό. Τώρα, ποιος κάνει την επιλογή των έργων. Αυτό είναι το σημαντικό. Ποιος έχει αυτή την αρμοδιότητα. Ποια κριτήρια χρησιμοποιούνται και πώς ελέγχεται αυτή η αρχή που προβαίνει στην επιλογή των ε, έργων. Το ακούσαμε και πριν. Η επιλογή της Επιτροπής Επενδύσεων, αν εκείνη είναι η αρχή που αποφασίζει, έτσι είναι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Αν πάντως είναι η Επιτροπή Εμπειρογνωμένων, δεν μπορεί να είναι μονόχρωμη όσον αφορά τις αρμοδιότητε, της. Και τι εννοώ με αυτό. Μην έχουμε μόνο οικονομολόγους, μην έχουμε μόνο ειδικού στην καινοτομία, χωρίς να έχουμε καθόλου ανθρώπους που να γνωρίζουν το χώρο. Ή αν δεν υπάρχει κάποιος που να είναι για την ε, οικολογία, ε, κάποιος που να είναι δικός για την απασχόληση. Δεν φτάνει. Γι' αυτό λοιπόν εμείς θα επιμείνουμε στην Επιτροπή αυτή οι να εκπροσωπούνται τα συμφέροντα και του κόσμου της εργασίας. Πολύ σημαντικό. Και το τελευταίο που θέλω να πω είναι το εξή. Σήμερα δεν έχω ιδιαίτερο πρόβλημα με αυτά τα οποία προτείνουμε στην αιτιολογική σκέψη. Υπάρχει όμως μία λογική απίστευτη που πιστεύω ότι είναι λάθος. Όταν λέμε ότι η προϋπόθεση για τις επενδύσεις είναι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις, πρώτα απ' όλα δεν ορίζονται αυτές. Τι είναι αυτές οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις. Και λέμε ότι συγχρόνως χρειάζεται δημοσιονομική ευθύνη, δηλαδή λιτότητα, ε, αυτό ακριβώς είναι το πρόβλημα. Πώς θέλετε να προχωρήσετε σε μεταρρυθμίσεις αν δεν έχετε χρήματα να τις χρηματοδοτήσετε. Και όλη η οικονομική ιστορία μας δείχνει ακριβώς το αντίθετο. Ότι δηλαδή όταν πρέπει να κάνουμε μεταρρυθμίσεις στις χώρες μας, να συμφωνήσουμε βέβαια ποιες είναι αυτές, ε, τότε ακριβώς είναι που χρειάζεται μια ευφυής οικονομική πολιτική και όχι περιοριστική. Άρα λοιπόν υπάρχει τροπολογία 1 στην σκέψη 2 που πιστεύω ότι επιδεινώνει αυτή τη λογική πρώτα λιτότητα και ε, μεταρρυθμίσεις, ευελιξία δηλαδή στην αγορά εργασίας, γιατί αυτό εννοούμε συνήθω, και μετά επενδύσεις. Μα αν αυτό λειτουργούσε, σήμερα η Ευρωζώνη και το ευρώ θα είχε υγείας. Χωρί κανένα πρόβλημα. Το πρόβλημα όμω τη Ευρώπη είναι ακριβώ ότι μέχρι τώρα ακριβώ αυτή την λογική ακολουθήσαμε που πρέπει να την αναστρέψουμε. Πρέπει να υπάρξει μείγμα των δύο και να πούμε ότι χρειάζεται μια πολιτική επενδύσεων που να βοηθάει μια πολιτική μεταρρυθμίσεων. Αλλιώ δεν βλέπω πώ θα τα καταφέρουμε. Γι' αυτό και με ενοχλεί αυτή ακριβώ η τροπολογία που σα είπα. Ευχαριστώ λέει Έχετε κάτι να προσθέσετε, αναφέρετε στη στην εισηγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ για τα καλά σας λόγια, για τα σχόλιά σας, για τη γνώμη σας. Πρώτα απ' όλα συγχωρήστε με γιατί δεν θα αναφερθώ συγκεκριμένα σε καθένα που έλεγε το λόγο, αλλά έχουμε υπερβεί το χρονικό όριο για τη συζήτηση του θρήσου υποσημείου αυτού. Πάντως όσον αφορά ε, αυτού του είδους την επενδυτική πλατφόρμα και κυρία Ροντρίγκε, είναι τα πράγματα όπω τα είπατε, πολύ σημαντικά. Έρευνα και ανάπτυξη. Εγώ θα, θα προσθέτω ότι αυτό θα πρέπει να γίνει μέσω ε, των ε, τοπικών και περιφερειακών αρχών και όλοι θα πρέπει να συνδυάσουν τις δυνάμεις τους τόσο ώστε να δημιουργήσουν νέες θέσεις απασχόλησης. Κύριε Γκύρικ, το γεωγραφικό κριτήριο ίσως δεν είναι το πιο ενδεδειγμένο. Νομίζω ότι η ECR θα έπρεπε κατά κάποιο τρόπο να αναθεωρήσει. Θέλετε οι προβληματικές περιοχές να εξαιρεθούν. Μα εγώ πιστεύω ότι εκείνες είναι οι περιοχές όπου μπορούμε να έχουμε πετυχημένη φορμή του προγράμματος και προς το παρόν δεν υπάρχουν εκεί επενδύσεις γιατί υπάρχει κάποιο είδους αγωνία σε σχέση με αυτές τις περιοχές αλλά δεν θα πρέπει να τις αφήσουμε απ' έξω. Επίσης, να με συγχωρούν όλοι ε, τον οποίο το όνομα ξεχνώ δεν το προφέρω καλά, αλλά ε, κάποια συνάδελφος αναφέρθηκε σε κάποια μακροπρόθεσμα προγράμματα. Μα εξορισμού αυτά τα προγράμματα θα είναι βράχη πρόθεσμα. Μιλούμε για τριετή περίοδο. Και πρέπει να σας πω ότι δεν συμφωνώ ότι πρέπει να δοθούν πόροι για κάποια προγράμματα μικρού κινδύνου. Με αυτά θα πραγματοποιηθούν έτσι καλώς. Λέμε και αυτά τα οποία ε, δεν θα μπορούσαν να γίνουν χωρίς την ενίσχυση. Ο κύριος Μπαλάς και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι αναφέρθηκαν στους ε, οι οποίοι πρόκειται να κάνουν αυτό το screening, τέλο πάντων τον έλεγχο αυτών των προγραμμάτων, μα αυτός ο έλεγχος, αυτό το φιλτράρισμα θα γίνει από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Εκείνοι θα τσεκάρουν τις, τις αιτήσεις. Οι οποίοι είναι ικανότατοι, έχουν όλες τις απαραίτητες ε, δεξιότητες και έχουμε όλους αυτούς τους συμβούλους οι οποίοι συμβουλεύουν τις επιχειρήσεις τους ώστε να προετοιμάζονται και να ε, υλοποιούνται τα έργα αυτά. Αλλά δεν ξέρουμε κατά πόσον αυτό θα ισχύσει παντού. Αυτό είναι το σημαντικό να δούμε τι θα γίνει, γιατί η Επιτροπή και η Τράπεζα Επενδύσεων μπορούν να φροντίσουν ε, αυτό το φιλτράρισμα, αυτό τον έλεγχο. Εμείς ασχολούμαι με τα υπόλοιπα και α εξασφαλίσουμε το να έχουν πρόσβαση ε, σε πολύ καλέ ε, συμβουλές οι επιχειρήσει και παντού στην Ευρώπη. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ και περιμένω τη συνέχεια τη συνεργασίας μας με προσμονή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Ευχαριστώ. Όταν ξεκινήσαμε αυτή τη συνεδρίαση, είχα θέσει το ερώτημα του κατά πόσο θα μπορούσαμε να καθυστερήσουμε τις ψηφοφορίες για μία από τις ε, αιτήσει χρήσης του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης και την αίτηση Μωρή Μικρό συγκεκριμένα και είπατε ναι θα την βάλουμε. Αλλά τότε δεν ήταν και πολλά μέλη παρόντα. Τώρα έχει αυξηθεί ο αριθμό των μελών και κάποιοι έχουν εγείρη αντίρρηση για την ε, αναβολή της ψηφοφορίας. Θέλουν να υπάρξει ψηφοφορία και για τις δύο αιτήσει του Ταμείου Παγκοσμιοποίησης είναι πάρα πολλοί λοιπόν οι οποίοι ήταν έτοιμοι για να ψηφίσουν. Το πρόβλημα είναι ότι το ΕΛΚ όμως ζήτησε την αναβολή για την δεύτερη αίτηση, όχι για την Lufthansa, αλλά για το Μωρί Ντικρό. Υπάρχει λοιπόν μια πρόταση. Πόσοι θέλουν να ψηφίσουμε και τις δύο αιτήσεις σήμερα. Και πώς θέλουν να αναβάλουμε τη δεύτερη. Λοιπόν, ψηφίζουμε και τις δύο ομούς σήμερα. Και όπως γίνεται πάντα με το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης θα πρέπει να είναι ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ξεκινάμε λοιπόν με την ε, αίτηση από την Lufthansa Technik. Άρχεται η ψηφοφορία. And the vote is closed. Πέρα της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται και πάμε στην αίτηση Μόλι Ντικρό. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και αυτή εγκρίνεται. Ευχαριστώ πολύ. Uh, Uh, Τώρα, ερχόμαστε στο σημείο 5. Δραστηριότητε και υποπτία των Ιδρυμάτων που προσφέρουν υπηρεσίε υπηρεσίες επαγγελματικών συνταξιοδοτικών παροχών. Και θα δώσω το λόγο στον εισηγητή, τον κύριο Λένα Αρς. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Ο τίτλος βέβαια είναι αρκετά μακρύς και περίπλοκος. Αυτό που είναι σημαντικό είναι να καθορίσουμε εδώ τα ιδρύματα αυτά επαγγελματικώ ταξιδιωτικών παροχών, τι ακριβώς είναι και τι κάνουν, γιατί μας αφορούν και να ξέρουμε τι δουλειά έχει γίνει μέχρι τώρα για τις συντάξεις στην Πράσινη και στη Λευκή Βίβλο. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό εδώ να πούμε ότι αυτά τα ιδρύματα έχουν κοινωνικό σκοπό καταρχήν και την ευθύνη συνταξιοδοτικών παροχών. Τα μέλη και οι δικαιούχοι τους δηλαδή πρέπει όταν σταματήσουν την εργασία τους να μπορούν να έχουν μια καλή σύνταξη. Υπάρχει συνεργασία επίσης μεταξύ των Ιδρυμάτων των ε, εργοδοτών και των εργαζομένων. Είναι πολύ βασική και αυτή και είναι μια βασική αρχή της οδηγίας η καλή αυτή συνεργασία. Γενικό σκόπος λοιπόν τώρα είναι να διευκολύνει τις αποταμιεύσεις για επαγγελματικές συντάξεις. Και τώρα με την οικονομική κρίση, όπως καταλαβαίνετε, οι συνταξιοδότη, οι συντάξεις μάλλον πιέζονται σε πολλές χώρες μέλη. Και ξέρετε ότι έχει δημιουργηθεί ένα τοπίο όχι και τόσο καλό όσον αφορά την αναλογία των ατόμων που εργάζονται και εκείνων που συνταξιοδοτούνται, δηλαδή που ζουν από τις συντάξεις τους. Αυτοί οι οποίοι χρηματοδοτούν τις συντάξεις, δηλαδή αναλογικά, είναι όλο και λιγότεροι. Κυρίως στον πρώτο πυλώνα. Για να αποφύγουμε λοιπόν την πίεση αυτή στον προπολογισμό των χωρών μελών μακροπρόθεσμα, είναι πολύ σημαντικό να βρούμε τρόπους να ενισχύσουμε τι συντάξει δεύτερου πυλώνα, δηλαδή ακριβώς αυτά τα ιδρύματα επαγγελματικών ταξιδιωτικών παροχών, τα IOPRs. Για να γίνει αυτό, να εννοείται πως είναι σημαντικό τα ιδρύματα αυτά να έχουν υψηλέ προδιαγραφές. Όσον αφορά την ασφαλειά τους, όσον αφορά την εποπτεία, τη διαφάνεια και αυτά ακριβώς είναι και τα πράγματα τα οποία προσπαθεί να πετύχει η πρόταση που εξετάζουμε. Και είναι όντω σημαντικό να υπάρξει εμπιστοσύνη σε αυτά τα συστήματα. Οι άνθρωποι πρέπει να εμπιστεύονται τα ιδρύματα επαγγελματικών ταξιδιωτικών παροχών και να νιώθουν ότι μπορούν να επενδύσουν σε τέτοια συστήματα. Αλλά χρειάζεται και κάτι άλλο. Προτεραιότητα της Ευρώπης πρέπει να είναι οι χώρες μέλη να οθούνται να αναπτύσσουν περισσότερα τέτοια ιδρύματα. Αλλά πρέπει να κάνουμε και κάτι παραπάνω. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει να παίξει σημαντικό ρόλο όσον αφορά τη συνεργασία κυβερνήσεων και κοινωνικών εταίρων προκειμένου να συζητούν για τη δημιουργία αυτών των ιδρυμάτων. Σε αυτή τη γνωμοδότηση λοιπόν προσπαθούμε να εντοπίσουμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν με τη λειτουργία των ιδρυμάτων αυτών και να δούμε πώς μπορούμε να οθήσουμε τις χώρες μέλη να κάνουν ακόμα περισσότερα προς αυτή την κατεύθυνση. Η Επιτροπή προτείνει τέσσερις συγκεκριμένους στόχους. Την άρση των υποπτικών εμποδίων για τα διασυνοριακά τέτοια δρήματα, τη διασφάλιση χρηστής διακυβέρνηση και διαχείριση των κινδύνων, την παροχή σαφών και σχετικών προφορών σε μέλη και δικαιούχου και την εξασφάλιση των αναγκαίων εργαλείων στι υποπτικέ αρχέ για την αποτελεσματική εποπτεία των ιδρυμάτων αυτών. Είναι όντω πολύ σημαντικά όλα αυτά. Και πρέπει να δούμε τι κάνουμε σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Το Κοινοβούλιο μας και η Επιτροπή μας πάντα τονίζει ότι τα συνταξιδοτικά συστήματα είναι άρρητα συνδεδεμένα με την οτροπία, τις συνήθειε τον τρόπο λειτουργίας των χωρών μελών. Έχουν ε, να κάνουν και με φορολογικές συνήθειες, με κοινωνικούς κανόνες που ισχύουν. Οπότε και εγώ πιστεύω ότι αν έχουμε το one size fit all στην Ευρώπη, δηλαδή ένα είδος μόνο τέτοιων ιδρυμάτων, δεν θα πετύχουμε αυτό που θέλουμε. Είναι σημαντικό δηλαδή οι χώρες μέλη να διατηρούν ένα βαθμό ευελιξίας, ώστε αυτό που κάνουμε, ο κοινό μας στόχος, να επιτευχθεί βάσει των εθνικών συστημάτων και των νοοτροπιών που επικρατούν σε κάθε χώρα. Πρέπει δηλαδή οι χώρες μέλη να αποφασίζουν τον καλύτερο τρόπο με τον οποίο θα το πετύχουν, να έχουν το περιθώριο να προχωρήσουν σε καινοτόμες διαδικασίες που ήδη ισχύουν σε κάποιες χώρες μέλη. Και βάσει της αρχής της επικουρικότητας επίσης οι χώρες μέλη έχουν την πλήρη ευθύνη για την οργάνωση των συνταξιδοτικών τους συστημάτων. Πιστεύω συνεπώς ότι η πρόταση αυτή πηγαίνει κάπως μακριά όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Επιτροπής που πλήττει τις εθνικές αρμοδιότητες για τον καθορισμό του κινδύνου ή των ωφελών από τα επαγγελματικά αυτά ιδρύματα συντάξεων. Πρέπει να προσέξουμε επίσης να μην δημιουργήσουμε υπερβολικές ρυθμίσεις με υπερβολικές λεπτομέρειες. Πρέπει να δείξουμε εμπιστοσύνη στις χώρες μέλη. Όταν υπάρχουν τέτοια ιδρύματα, να αντιμετωπίσονται όχι οι άσπρο-μαύρο, αλλά να λαμβάνονται υπόψη και όλες οι αποχρώσεις. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε έξι για να εξηγήσουμε τι πρέπει να είναι μέσα σε ένα ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιδοτικών παροχών. Πρέπει να δείξουμε ευελιξία, γιατί υπάρχουν χώρες που έχουν πολύ καλές εξελίξεις όσον αφορά αυτά τα ιδρύματα. Δεν πρέπει να δυσκολεύουμε τη δουλειά τους λοιπόν. Εν κατακλείδη, αυτό που προσπαθώ να κάνω στο σχέδιο γνωμοδότησής μου είναι να διασφαλίσω μια καλή ισορροπία. Από τη μια μεριά δηλαδή να έχουμε υψηλές προδιαγραφές σε ευρωπαϊκό επίπεδο, ώστε οι άνθρωποι και οι χώρες να μπορούν να εμπιστευθούν τα συστήματα αυτά και όταν συμμετέχουν σε ένα τέτοιο ίδρυμα επαγγελματικών συνταξιδοτικών παροχών να ξέρουν ότι θα πάρουν μια καλή σύνταξη όταν έρθει η ώρα, αλλά αυτό να το συνδυάσουμε και με ένα βαθμό ευελιξίας στις χώρες μέλη ώστε να μπορούν να προσαρμόσουν τους κανόνες έτσι ώστε αυτοί να συνάδουν με τις εθνικές παραδόσεις και τις εργασιακές επίσης παραδόσεις. Ευχαριστώ. Πρόεδρος. Ιωκίμ Σούστε από τους Σοσιαλιστές και Δημοκράτες. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Μπορώ να συμφωνήσω σε πολλά σημεία με τον ε, προλαλήσαντε. Νομίζω ότι υπάρχουν πολλά θετικά στοιχεία τα οποία περιλαμβάνονται σε αυτή την πρόταση. Εγώ θα ήθελα να σταθώ σε ένα πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο, το οποίο είναι θέμα ουσίας. Όταν υπάρχει σαν συνταξιοδοτική παροχή, αυτή δεν είναι παροχή υπηρεσίας, είναι μια κοινωνική παροχή υπηρεσίας. Θα πρέπει λοιπόν αυτό να παραμείνει μέσα στην κοινωνική οικονομική παράδοση. Επομένως θα πρέπει να υπάρχουν όρια στις ε, ευρωπαϊκές ρυθμίσεις για τα θέματα αυτά. Αν δούμε την πρόταση της Κομισιόν, βλέπω πολλά θετικά στοιχεία σε σχέση με την προηγούμενη κατάσταση. Από την άλλη πλευρά όμως υπάρχει μια προσπάθεια να υπάρξει απλώς και μόνο η συμπλήρωση της εσωτερικής αγοράς. Αυτό σημαίνει όμως για μας και μας φαίνει κάποιες ανησυχίες ότι η, χρήση του πυλώνα 2 στις επιχειρήσεις δεν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Τίθεται εδώ το θέμα της καλύτερης πληροφόρησης των εργασομένων και των ε, συστημάτων διακυβέρνησης που θα πρέπει να μας οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι εδώ δεν μπορούμε να έχουμε μια συνολική ευρωπαϊκή ρύθμιση όπως γίνεται παραδείγματος στο χρηματοπιστωτικό τομέα και γίνονται εκεί οι απαραίτητες ενέργειες. Στην περίπτωση της σύνταξης που παίρνει ένας εργαζόμενος από την επιχείρηση πρέπει να έχουμε μια διαφορετική αντιμετώπιση για να μην αποδυναμώσουμε το καθεστώς αυτό. Η Κομισιόν έχει αφαιρέσει πολλά στοιχεία από την αρχική της ιδέα, αλλά παραμένουν κάποιες κερκόπορτες ακόμα που συνδέονται με την ε, οδηγία για την ε, αφαιρεγγιότητα, το, ε, την αφαιρεγγιότητα 2. Υπάρχει λοιπόν ένα σύνολο προτάσεων από, από την Κομισιόν στον τομέα αυτό, ίσως κάτι ακόμα το οποίο θα πρέπει να λάβουμε υπόψη ως προβληματικό είναι εδώ πέρα η πρόταση στην, στο έγγραφο της Κομισιόν να μην υπάρξει, να πάψει να υπάρχει πλέον η κρατική εποπτεία στα θέματα αυτά. Αυτό είναι κάτι το οποίο εμείς το βρίσκουμε ιδιαίτερα σαφές στην πρόταση της Κομισιόν. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς θέλει να επιτύχει η Κομισιόν και εδώ φυσικά βρισκόμαστε σε ένα τομέα ο οποίος μπορεί να δημιουργήσει κινδύνους για τις ε, εισφορές των εργαζομένων εάν δεν υπάρξουν επαρκή ε, όρια σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο θα χρησιμοποιούνται αυτές οι εισφορές παραγωγός χάρη σε τοποθετήσει στο χρηματιστήριο που μπορούν να είναι κερδοσκοπικές. Υπάρχουν λοιπόν, όπως είπε και ο εισηγητής, ε, υπάρχει ανάγκη να έχουμε πολλές τροποποιήσεις τροπολογίες που θα καταθέσουμε για το θέμα αυτό και ελπίζω ότι θα μπορέσουμε με περαιτέρω συζήτηση να καταλήξουμε σε μια σωστή γνώμοδότηση και να επιτύχουμε αυτό το οποίο είναι ο πραγματικός μας στόχος και αρμοδιότητάς μας να μην αντιμετωπίσουμε σαν μια καθαρά οικονομική παροχή υπηρεσιών την ε, συνταξιοδοτική παροχή, αλλά να, κανονίσουμε ότι, να καθορίσουμε ότι είναι ένα θέμα που υπόκειται στην επικουρικότητα, ότι είναι μια κοινωνική παροχή και πρέπει να τύχουν σεβασμού οι εθνικές προδιαγραφές στον τομέα αυτό. Ευχαριστώ κύριο Γκέρικε από την ομάδα των συντηρητικών. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή τη στιγμή είναι σημαντικό να έχουμε εξασφάλιση των ε, παροχών σύνταξης για τους εργαζομένους και τις οικογένειές της. Θα πρέπει να ενισχύσουμε το σύστημα που ισχύει στη Γερμανία, στην Αγγλία, στην κάτω, στις κάτω χώρες κτλ. Και εδώ θα πρέπει να είμαστε σαφείς. Εγώ χαιρετίζω ιδιαίτερα την έκθεση του κυρίου Λέναρτς. Θέτει ένα, ενώπιον μας ένα σαφή δρόμο ο οποίος ακολουθεί αυτά τα οποία έχει προτείνει η Κομισιόν. Η σύνταξη δεν είναι ένα χρηματοπιστωτικό προϊόν. Είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να οδηγεί σε μια ασφαλή κοινωνική παροχή για όλους τους εργαζόμενους. Οι, σύνταξη, συντάξεις είναι κάτι το οποίο θα πρέπει, όπως λέει και η Λευκή Βίβλος, να έχουν βιώσιμο χαρακτήρα και να εξασφαλίσουν μια αξιοπρεπή διαβίωση μετά τη συνταξιοδότηση. Και επομένως οι συντάξεις που προέρχονται από τα ταμεία των επιχειρήσεων παίζουν ένα σημαντικό τομέα, ένα σημαντικό ρόλο. Είναι απαραίτητο λοιπόν εμείς να μην μπλοκάρουμε την χρήση αυτών των συνταξιοδοτικών ταμείων, αλλά να τα ενισχύσουμε. Εγώ με εναντίον κάθε μορφής γραφειοκρατίας η οποία προωθείται. Όποιος δει τα, ε, τα υποδείγματα για τη σύνταξη στην Ευρώπη βλέπει ότι είναι μορφά αυτά τα μοντέλα και διαφορετικά. Δεν μπορεί να υπάρξει μία ενιαία λύση για όλα αυτά. Είναι απαραίτητο λοιπόν να μην επιβαρύνουμε τους εργαζομένους. Κανείς δεν μπορεί να καταλάβει όλα αυτά τα ψηλά τα οποία γράφουν οι προδιαγραφές για τις ε, συντάξεις. Θα πρέπει να είναι σαφή και εύληπτα αυτά τα οποία προβλέπονται. Και προβλέπω σε, προσβλέπω σε μια καλή συνεργασία με τον εισηγητή και τους σκιώδεις εισηγητές και μια καλή έκβαση για τους συνταξιοδοτημένους και τις οικογένειές τους. Thank you, ε, from the... Η κυρία Χάρκιν από την Άλντε. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Δυστυχώς τώρα δεν μπορώ να πω τίποτα. Γιατί ασχολούμαι 24 ώρες την ημέρα με το TTIP. Ε, συμπαθάτε με, θα τα πούμε αργότερα με τον εισηγητή. Από την ΚΟΕ κάποιος, κύριε Γκονσάλες, για το λόγο. Γεια σας. Καλημέρα, σας ευχαριστούμε Νομίζω ότι όλοι συμφωνούμε ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να βελτιωθεί ο πλευρά διαφάνεια η διαχείριση των ε, συντεκτικών ταμείων. Γιατί αυτό υπάρχει μια παρεμβολή πολύ ενοχλητική στο μικρόφωνο της ομιλήτριας. sí. <laughs> Καλημέρα σα και πάλι έλεγα ότι συμφωνούμε πως θα πρέπει να υπάρχει περισσότερη διαφάνεια στην διακυβέρνηση, στη διαχείριση των των ταμείων, αλλά αυτό να μην οδηγήσει σε κάποιο είδους ιδιωτικοποίηση από την πίσω πόρτα, γιατί κάποιοι συνάδελφοι εδώ εκεί το πάνε. Πρόκειται για το επιχείρημα ότι δηλαδή οι, τα κρατικά διευθυντικά ταμεία δεν, δεν αντέχουν και αυτό το ακούμε κάθε φορά που έχουμε ιδιωτικοποίηση κάποιες κρατικής υπηρεσίας. Ε, αυτό είναι αφόρητο, αυτό είναι έολο πλέον το επιχείρημα, οπότε και θα πρέπει να υπάρχει ε, ένα, άλλο επιχείρημα, όχι δηλαδή ότι δεν αντέχει το δημόσιο. Και να καταλήξουμε σε κάποιο ιδιωτικό φορέα που μόνο λίγοι μπορεί να καλυφθούν από αυτό. Μα μιλάμε για κάποιο αγαθό που αφορά το βιωτικό επίπεδο των ανθρώπων που ε, έχουν αποχωρήσει από τον ενεργό βίο. Να μην πάμε σε κεκαλυμμένη ιδιωτικοποίηση, λέει ξανά η Μιλήτρια. Και πολλές φορές ωφελούνται από τέτοιες προσπάθειες επομένως καπιδιωτικοί φορείς και εξαπατούν κάποιες οικογένειες οι οποίες πιστεύουν ότι έτσι θα βρουν μια λύση για το μέλλον. Εναρμόνιση να γίνει, αλλά για τις κρατικές συντάξεις, εκείνες ε, στις οποίες έχει όλος ο κόσμος πρόσβαση και μπορεί έτσι να διατηρήσει το βιωτικό του επίπεδο τα τελευταία χρόνια της διαδρομής του γιατί και στη χώρα μας έχουμε κάθε μέρα ολοένα και περισσότερους οι οποίοι ε, κρατιούνται από τις συντάξεις των παππούδων και των γιαγιάδων και ολόκληρη οικογένεια εξαρτάται από αυτούς μια που δεν έχουν δουλειά. Επομένως προσοχή γιατί εδώ πέρα διακυβεύεται η ευημερία της κοινωνίας μας. Thank you. Ε, ευχαριστούμε λέει η Πρόεδρος. Κύριε Τόμας για το λόγο. Ευχαριστώ πολύ και εγώ θέλω να ευχαριστήσω τον Ζερούν. Νομίζω ότι έχει κάνει μια πολύ καλή έκθεση η οποία εξισορροπεί τις διάφορες αιτήσει οι οποίες είναι απαραίτητε, οι οποίες διατυπώνται σε σχέση με την απαραίτητη συνταξιοδοτική προστασία. Εγώ δεν μπορώ να δεχθώ την έννοια του ότι η ρύθμιση για τις συντάξεις είναι μια συγκεκαλυμμένη ιδιωτικοποίηση. Όποιος δει προσεκτικά τι λέει η πρόταση καταλαβαίνει ότι δεν είναι αυτός ο στόχος μας. Είναι μια πάρα πολύ σημαντική περιοχή όπου θέλουμε να δώσουμε τη δυνατότητα να υπάρχει μια απόλυτη εξασφάλιση από την, ε, για τις συντάξεις αλλά αυτό το σύστημα δεν είναι ένα σύστημα το οποίο ισχύει σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε κάνει κάποιες εκθέσεις για τα θέματα αυτά στο παρελθόν στην Επιτροπή ΕΚΟΝ την τελευταία φορά και εκεί υπήρξε μια γενική συνένεση για μια τέτοια ρύθμιση. Το πιο σημαντικό σε σχέση με τη ρύθμιση αυτή των ε, συντάξεων σε χώρες όπως είναι η Ολλανδία, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο το δύσκολο εκεί είναι αυτό το οποίο αναφέρει ο Ζερούν. Δεν είναι δυνατόν το σύστημα αυτό να μεταλαμπαδευτεί σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα σύστημα το οποίο ισχύει παντού. Πάντως στη Γερμανία το σύστημα αυτό είναι κάτι το οποίο λειτουργεί. Αυτή τη στιγμή έχουμε φτάσει σε 460 δισεκατομμύρια ευρώ που είναι το σύνολο των ε, ε, ενεργητικών των ταμείων που δίνουν συντάξεις. Αυτό συνάδει με πολύ υψηλή όχι μόνο ποσότητα αλλά και ποιότητα παροχών. Θα ήθελα λοιπόν να γίνει σαφές ότι δεν, δεν θέλουμε να θεωρήσουμε τα συνδεδοτικά ταμεία ως παρόχους χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών και επομένως το Solvency 2 δεν θα πρέπει να εφαρμόζεται σε αυτά τα ταμεία. Οι επίτροποι, όπως ξέρετε, έχουν ένα χρονικό οριζόντα 5 ετών, αλλά η Κομισιόν συνεχίζει την επεξεργασία των θεμάτων αυτών και πολλές φορές επανέρχεται μία ε, εντύπωση ότι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν όχι σαν κοινωνικές συλλογικές παροχές οι συντάξεις αλλά μόνο ως ένα ε, χρηματοπιστωτικό προϊόν. Μα η Κομισιόν το τονίζει ότι είναι πρώτα απ' όλα ένα κοινωνικό προϊόν. Και νομίζω ότι πρέπει να υπάρξει και μια ολιστική εξισορρόπηση, ένα, ένα ολιστικού ισολογισμού για όλα αυτά τα θέματα όπου θα μπορέσουμε να δούμε ποια είναι τα θετικά και τα αρνητικά στοιχεία. Δεν θα πρέπει λοιπόν να δώσουμε μια τέτοια εικόνα χρηματοπιστωτικού προϊόντος για τις συντάξεις. Έχουμε αρκετές πληροφορίες και έχουμε και αρκετά στοιχεία που μας επιτρέπουν να έχουμε μια σωστή αντιμετώπιση και εγώ δεν καταλαβαίνω τους συναδέλφους που αναφέρονται σε γραφειοκρατία. Η γραφειοκρατία χρειάζεται να υπάρχει μια διαχείριση όλων αυτών. Θα πρέπει να μπορεί κανείς να παρακολουθήσει όλα αυτά τα πράγματα. Υπάρχουν πάρα πολλές πληροφορίες οι οποίες υπάρχουν πραγματικά όταν κατεβάζω ένα app από το διαδίκτυο. Θα διαβάζει αυτά κανείς. Λέει κανείς ότι α, θα τα διαβάσω όλα και θα πω ότι δεν δέχομαι αυτήν την, ε, την αλλαγή, την αναβάθμιση. Πρέπει λοιπόν να υπάρχει δυνατότητα σωστής πληροφόρησης για όλους. Οι συνταξιοδοτήσεις λοιπόν έχουν κάποιες ε, εξασφαλίσεις για την ε, παροχή τους. Πιστεύω λοιπόν ότι μέχρι στιγμής το μοντέλο αυτό το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε χώρες όπως η Γερμανία, η Ολλανδία και η Μεγάλη Βρετανία είναι μια πραγματική επιτυχία γιατί και οι εργαζόμενοι έχουν συμβάλει στη λειτουργία αυτού του στοιχείου και η Κομισιόν δεν θα πρέπει να προσπαθεί να τα ισοπεδώσει όλα σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αναφέρεται ο κύριο Σούστερ για τα κεφάλαια τα οποία ε, τοποθετούνται σε κατά κάποιο τρόπο ριψοκίνδυνες τοποθετήσεις. Όλες οι τοποθετήσεις όμως συνδέονται με κάποιο κίνδυνο. Μπορεί να, είναι κανείς, να έχει κανείς τοποθετήσει τα χρήματά του κάπου που να νομίζει ότι απλώς παίρνει μερίσματα, αλλά πάντα υπάρχει ένας κίνδυνος. Όλες οι επενδύσεις υπόκειται σε κάποιο κίνδυνο, ακόμα και αν είναι απόλυτα ασφαλής, όπως λέγεται. Αυτή τη δυνατότητα λοιπόν δεν μπορούμε να την απεμπολίσουμε. Και είναι σωστό να το κατανοήσουμε ακόμα και ο τομέας αυτός των επενδύσεων είναι ένα σημαντικός τομέας. Κανείς ο οποίος είναι επιτυχής δεν αντιμετωπίζει ελαφρά την καρδία την επένδυση αυτών των ε, κονδυλίων. Μίλησαμε προηγουμένως για τα 315 δισεκατομμύρια του σχεδίου Juncker. Μα θέλουμε να συμμετάσχει και ο ιδιωτικός τομέας δίνουμε δημόσια χρήματα, αλλά χρειάζεται και από τους παίκτες της αγοράς, από τον ιδιωτικό τομέα να συμμετάσχει. Δεν μπορούμε λοιπόν να αγνοήσουμε το γεγονός ότι η δυνατότητα κερδοφορίας συνδέεται πάντα με κάποιο κίνδυνο. Η πολιτική συντάξεων λοιπόν έχει να αντιμετωπίσει και τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν από την πολιτική χαμηλών επιτοκίων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτό θίγει τα συνταξιοδοτικά ταμεία. Εγώ έρχομαι από την περιοχή της Φραγκφούρτης και είναι πολύ κοντά μου η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, αλλά ο τομέας των συντάξεων πρέπει και αυτός να αντιμετωπιστεί από τον κύριο Ντράγη και την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Λέει η κυρία Γιαζλόφικα. Πολύ χαίρομαι που ο συνάδελφος ασχολήθηκε με το θέμα αυτό. Πριν από λίγο καιρό, όντως ήταν εκείνη που ασχολιόταν με αυτά, τώρα ο εισηγητής μας νομίζω ότι είναι αποφασισμένος να προχωρήσει. Η έκθεση αυτή λοιπόν δείχνει ότι όλη η δουλειά που έγινε, έγινε με μεγάλη σοβαρότητα. Συμφωνώ για το ότι πρέπει πραγματικά να ασχοληθούμε κυρίως με τη διασυνοριακή πτυχή. Εγώ είμαι πάντα υπέρ της κινητικότητας, ιδιαίτερα μάλιστα σήμερα που βρισκόμαστε σε οικονομική κρίση. Πρέπει λοιπόν σήμερα να βρούμε τις ιδανικές συνθήκες για τα άτομα εκείνα τα οποία δουλεύουν στο εξωτερικό προκειμένου να διασφαλιστούν οι συντάξεις τους. Μιλήσαμε επίσης για διαφορετικούς κινδύνους. Πρέπει να ενθαρρύνουμε τις χώρες μέλη να δημιουργήσουν τους τρεις πυλώνες, ώστε το σύστημα να είναι πιο σταθερό. Η ασφάλεια μπορεί να υπάρξει και να την εγγυηθούμε εφόσον έχουμε συντάξεις καλής ποιότητας. Και όσον αφορά τα διασυνοριακά ζητήματα, η ποιότητα αυτή είναι ζωτική σημασίας. Οι λύσεις αυτές που θα βρούμε πρέπει να είναι αξιόπιστες, γιατί μόνο τότε οι πολίτες μπορούν να μας εμπιστευτούν. και να μπορέσουν όλοι να εξυπηρετηθούν από ένα τέτοιο σύστημα. Ευχαριστούμε κυρία Μακιντάιρ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον κύριο Λέναρς για τη δουλειά του για αυτή την υπόθεση. Η Όμεν Ράιτεν πρέπει να το θυμίσω αυτό, στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία έκανε πάρα πολλή δουλειά για αυτά τα ιδρύματα. Ξέρουμε λοιπόν την Ολλανδική άποψη, τη Γερμανική άποψη και όλοι λίγο πολύ συμφωνήσαμε με αυτό το θέμα. Και εγώ το στήριξα πολύ και στηρίζω αυτά που είπε ο Τόμας Μαν. Εμείς αυτό που κάνουμε είναι ότι αμφισβητούμε την ε, ανάγκη για παρετέρω νομοθεσία. Θεωρούμε ότι δεν έχει αποδειχτεί ανάγκη για παρετέρω ρύθμιση. Όσον αφορά την ε, εκτίμηση αντικτύπου, αυτό είναι σημαντικό. Και φυσικά και θέλουμε εμείς καλύτερη ρύθμιση. Πρέπει λοιπόν να επιμείνουμε εδώ ότι θέλουμε μια αιτιολογημένη πρόταση. Να δούμε δηλαδή γιατί χρειάζεται. Θέλουμε να δούμε την εκτίμηση αντικτύπου, δηλαδή ποια θα είναι τα αποτελέσματα. Γιατί χρειάζεται. Εγώ δεν πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αντιμετωπίσει σωστά το θέμα της αναλογικότητας. Είναι πολύ ανησυχητικό το γεγονός ότι υπάρχουν κάποιες απαιτήσεις εδώ που θα επιβαρύνουν οικονομικά το σύστημα. Προσπαθούμε τις, ε, τα επαγγελματικά αυτά στα εξοδοτικά συστήματα να μην επιβαρύνουν περισσότερο διοικητικά το όλο σύστημα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επίσης βλέπω ότι θέλει και ένα θέμα αξιολόγησης. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, βλέπετε, είναι τραστ αυτοί που έχουν τα σταξιδιωτικά συστήματα και υπάρχουν ε, δικαιούχοι μέσα από τα συνδικάτα. Αν ήταν μόνο επαγγελματίες, τότε ένα καλό σύστημα με εκπροσώπους από τις δύο πλευρές θα μπορούσε να σταθεί. Όσον αφορά την επικουρικότητα τώρα. Και αυτό είναι ένα σημαντικό θέμα. Όπως ακούσαμε, υπάρχει διαφορετική νομοθεσία στις χώρες μέλη. Δεν μπορούμε να έχουμε μία ρύθμιση που να ταιριάζει σε όλους να πάμε από 30 άρθρα σε 80 για να συμπεριλάβουμε τα πάντα και να ρυθμίσουμε τα πάντα είναι εντελώς λάθος. Και σαν παράδειγμα θα σας πω το εξής. Στο Ηνωμένο Βασίλειο αρχίσαμε μια αυτόματη συμμετοχή σε κάποιο επαγγελματικό σύστημα. Δεν είναι ότι θέλουμε να κάνουμε περισσότερα, Αυτό που γίνεται μέχρι τώρα δηλαδή είναι πολύ καλό με αυτό το αυτόματο σύστημα. Οπότε εμένα πολύ με απασχολεί το να βάλουμε από την πίσω πόρτα τις απαιτήσει της οδηγίας Όλβανση 2. 2. Θα ήθελα να προσθέσω και κάτι ακόμα. Ή που είμαστε υπέρ του τρίτου πυλώνα που θεωρούμε ότι είναι κάτι σημαντικό, όπως συμβαίνει στο Ηνωμένο Βασίλειο, γιατί πιστεύουμε ότι έτσι χρησιμοποιούνται καλά οι επαγγελματικές συντάξεις, γιατί είναι συντάξεις οι οποίες ανήκουν σε άτομα. Όταν λοιπόν το άτομο αλλάξει δουλειά, αλλάξει χώρα, το συνταξιοδοτικό του πακέτο πρέπει να το συνοδεύει. Και οι εργοδότες επίσης πρέπει να συνεισφέρουν σε αυτό το σταξιδοτικό του πακέτο. Και όταν είχαμε συζητήσει για τις συντάξεις, το είχα αναφέρει και τότε. Είχα πει ότι έπρεπε να το σκεφτούμε και να το στηρίξουμε. Λοιπόν, ευχαριστώ και πάλι τον εισηγητή για το έργο του εδώ. Ευχαριστώ, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Σιγητά, θέλετε να προσθέσετε κάτι. Λένας. Ευχαριστώ πολύ στον Αντρέα που τον λόγο. Χαίρομαι πάρα πολύ που υπάρχει ευρεία συνένεση σε σχέση με το τι χρειάζεται να γίνει και τι γίνεται από πλευρά ε, κοινωνικών στόχων και ε, για αυτά τα ταμεία, αυτούς τους φορείς, ε, τι χρειάζεται ο κόσμος. Άκουσα κάποιο συναδέλφο την κυρία Μακεντάρ, τον κύριο Σούστερ και άλλους οι οποίοι μίλησαν για το νομοθέτημα για την των παραθμών 2 οπότε θα πρέπει και εμείς να εξασφαλίσουμε ότι οι προϋποθέσεις που τάσει αυτό το νομοθέτημα δεν θα ε, τις επικληθήκαν, δεν τις επικαλεστήκαν, ε, συγγνώμη, από την Κερκόπορτα να μπουν μέσα δηλαδή, στο παιχνίδι. Οπότε ε, και κάτι άλλο το οποίο άκουσα ότι ίσως δεν χρειάζεται επιπλέον νομοθεσία, όπως είπε ο κύριος ε, Σούστερ, αλλά να είμαστε προσεκτικοί, μην αυξήσουμε το κόστος το διοικητικό ή την γραφειοκρατία, γιατί ό,τι προσθέτουμε σαν κόστος τελικά μετακυλίεται στους ε, συνταξιούχους. Άρα, εμείς από τις θέσεις μας θα πρέπει να εξασφαλίσουμε το ότι θα υπάρχει ένα ευρωπαϊκό πλαίσιο το οποίο θα εξυπηρετεί τα συμφέροντα των ε, Ευρωπαίων. Συμφωνώ και με αυτό που ο κύριος ε, Μάν αλλά και η κυρία Γκονσάλες για την εξαπάτηση και για την κεκριμένη ιδιωτικοποίηση όχι, δεν έχει δίκιο. Γιατί εμείς θέλουμε να εξασφαλίσουμε το ότι η δίποτε στεξιωτικό πρόγραμμα θα είναι επικουρικό στις συντάξεις του πρώτου πυλώνα. Κάτι το οποίο έχει μεγάλη σημασία σε όλα τα κράτη-μέλη να συνεχιστεί και να υπάρχει μια επαρκή σύνταξη ε, για τον κόσμο όταν έρθει η ώρα. Πολύ σημαντικό αυτό για τους εργαζομένους για να μπορέσουν να έχουν καλύτερο βιωτικό επίπεδο από ότι με την απλή σύνταξη του πρώτου πυλώνα όταν συνταξιδοτηθούν. Να πιένει είναι η προσθεμένη αξία της υπόθεσης αυτής. Τέλος πάντων περιμένω πώς και πώς τη συνεργασία με τους συναδέλφους. Σας ευχαριστώ για τις προτάσεις σας και θα τα συζητήσουμε εντελεχέστερα. Πρόεδρος. Σας ευχαριστούμε. 19 Τρίτου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες και 16 Τετάρτο θα τα συζητήσουμε. Θα ψηφίσουμε 28 Πέμπτου εδώ και στην Οικονομική τον Νοέμβριο. Όπως γνωρίζετε, εδώ πρόκειται περί αναδιατύπωσης ε, προϊσχυσάσεις, οδηγίες. Επομένως, οι τροπολογίες θα αφορούν μόνο τα σημεία του κειμένου που ήδη τροποποίησε η Επιτροπή. Αυτά που είναι με έντονους χαρακτήρες στην πρόταση της Επιτροπής. Άρα εκεί θα τροπολογήσουμε μόνο να πρόκειται αναδιατύπωση. Σας ευχαριστώ. Και τώρα, πάμε στο σημείο 6 της μέσης διατάξεως. Το οποίο είναι το ίδιο σαρπαστικό όπως και οι συντάξεις. Είναι το TTIP, η Ατλαντική Σχέση Εμπορίου Επενδύσεων. Και θα δώσουμε τώρα το λόγο στην εισηγητριά μας, την κυρία Χάργεν. Έχεις το λόγο. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα ένα-δύο γενικότερα σχόλια ότι καταρχήν εγώ είμαι υπέρ μιας ε, εμπορικής συμφωνίας με τη ΣΥΠΑ από πλευράς ε, πολιτικής, από πλευράς στρατηγικής τουλάχιστον και ε, άλλωστε η χώρα από την οποία προέρχομαι έχουμε τέτοιου είδους οικονομία που αν δεν εμπορευτούμε δεν μπορούμε να επιβιώσουμε. Και έχουμε ήδη πολλές περισσότερο από όσο νομίζει κανεί εμπορικέ ροέ με τη ΣΥΠΑ. Πάντω το εμπόριο δεν είναι αυτό ο σκοπό. Οπότε θα πρέπει να υπάρξουν και άλλου είδου ωφέλη από το εμπόριο και όχι μόνο ε, οικονομικά. Να δούμε τι θα γίνει με αυτή την πρόταση όμω σε σχέση με αυτό. Γιατί έχουμε ένα σωρό εμπορικέ συμφωνίε και έχουμε κάποιε εξαιρέσει όπω ε, η συμφωνία με τον Καναδά, οι οποίε κυρίω συμφωνίε αφορούν την κατάργηση, τη μείωση τέλο πάντων των. Ε, δασμών ε, που είναι σημαντικές βέβαια και με τη ΣΥΠΑ αλλά τώρα εδώ πρόκειται περί άλλου πράγματος γιατί θα πρέπει να δούμε τι θα γίνει με πρόσβαση στην αγορά με τις ε, δημόσιες προμήθειες και με την ε, συνεργασία, συνεργασία των ρυθμιστικών αρχών. Θα και να δούμε πώς θα αρθούν οι τεχνικοί φραγμοί στο εμπόριο. Αλλά με τι εμπορικέ διατάξει να έχουμε βιώσιμη ανάπτυξη μέσω του εμπορίου. Και αυτό θα γίνει με την προστασία του περιβάλλοντος και των εργασιακών δικαιωμάτων. Να δούμε πώς θα έχουμε ελεύθερο ανταγωνισμό και να δούμε πώς θα βρούμε κάποιους τρόπους ώστε να επιλύσουμε τις ε, διαφορές στα πλαίσια της εμπορικής συμφωνίας. Χθε ήμουν ε, ε, η διευθύνουσα, τέλο πάντων πρόεδρο, σε κάποια εκδήλωση για το τίτλο εδώ στο Κοινοβούλιο και ο κόσμο έλεγε ότι υπάρχει περίεργο μεγάλο ενδιαφέρον για Εγώ δεν το θεωρώ κάτι το περίεργο αυτό αλλά λόγω της ε, συνθήκης της Αγώνα τώρα το Κοινοβούλιο έχει ευξημένε αρμοδιότητες ε, επί του προκειμένου. Πάντως ε, ακριβώς επειδή πρόκειται για τέτοιου συμφωνία για αυτό και ο κόσμος ενδιαφέρεται πολύ. Δηλαδή δεν είναι μόνο τα αγαθά, είναι το εργατικό δίκαιο, είναι η εξασφάλιση της απασχόλησης, είναι η επιβίωση του κοινωνικού μας μοντέλου ε, είναι και θέμα δυνατότητας νομοθεσίας των κρατών. Γι' αυτό νομίζω είναι σημαντική υπόθεση αυτή, αλλά υπάρχουν και σημαντική κίνδυνη πρώτα-πρώτα. Κάτι το οποίο πολλοί το κουβεντιάζουν. Το ISDS. Οι επενδύσεις. Για το ΣΕΤ Το 2011 είχαμε ένα ψήφισμα. Και το ψήφισμα αυτό έλεγε επιλέξει ότι υπάρχουν αναπτυγμένα νομικά συστήματα σε, σε Ένωση και Καναδά και παρά τον ε, μηχανισμό τον, ε, και, και μάλλον υπάρχει μηχανισμός όπου με επαρκή τρόπο επιλύονται οι διαφορές οι οποίες ανακύπτουν από τις επενδύσεις, από το ISDS δηλαδή. Αλλά είπε ο κύριος Γιούνκερ ότι υπάρχει πρόβλημα το ότι πάρα πολλοί δεν δέχονται τη δικαιοδοσία των ευρωπαϊκών δικαστηρίων, οι οποίοι, τα οποία άρα λίγα μπορούν να κάνουν όσον αφορά τι διαφορέ για τι επενδύσει. Άρα θα πρέπει για το ISDS να δούμε τι θα γίνει, θα πρέπει όλα αυτά να ληφθούν υπόψη σε ό,τι και αποφασίσουμε τυχόν. Τέλος πάντων, πριν δούμε τώρα τις ε, λεπτομέρειες, έχουμε εδώ πέρα ένα κείμενο 1500 λέξεων και θα πρέπει όλα αυτά να τα κοιτάξουμε καλύτερα, να, να τα βελτιώσουμε με τις τροπολογίες. Κάποια θέματα δεν τα έχω θίξει, τα οποία θα πρέπει να τα περιλάβουμε και η μεθοδολογία μου είναι να προσπαθώ να βρω λύσεις ούτως ώστε να αποδώσει η υπόθεση αυτή. Γιατί έχουμε συγκεκριμένες προκλήσεις να αντιμετωπίσουμε. Για να τώρα. Τι λέω εδώ στο κείμενο. Είπαμε για το TTIP, το οποίο θα πρέπει να βοηθήσει για να έχουμε περισσότερες, καλύτερες θέσεις απασχόλησης και όσον αφορά τις θέσεις απασχόλησης έχει κάνει μελέτη στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει κάποιες τεχνικές αξισορρόπησης. Τι να σας πω, δεν καταλαβαίνω πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα, αλλά τέλος πάντων νομίζω ότι ανάλογα με το τι στοιχεία δώσει κανείς σε αυτό το σύστημα θα πάρει άλλα αποτελέσματα. Ε, πρόκειται για τη ζήτηση της απασχόλησης και άλλα μεγέθη. Αλλά αυτό είναι και το πρόβλημα που έχουμε εδώ. Γιατί έχουμε εδώ διαφορετικές αναλύσεις. Το δε ερευνητικό μας κέντρο ασχολήθηκε με αξιόλογο τρόπο με την ε, έκθεση της Επιτροπής και την ανέλησα και νομίζω είναι πάρα πολύ χρήσιμα τα αποτελέσματα. Πάντως, όπως είπαμε, έχουμε ένα σωρό εκθέσεις, αναλύσεις, η καθεμία έχει διαφορετικά αποτελέσματα. Αλλά για να δούμε και άλλες εμπορικές συμφωνίες, όπως της ναύτα. Εκεί υπερεκτιμήθηκαν τα θετικά αποτελέσματα και εμείς ως νομοθέτες θα πρέπει να νιώθουμε κάποια βεβαιότητα θα πρέπει να νιώθουμε την ασφάλεια των ε, στεγανών στοιχείων πάνω στα οποία δουλεύουμε. Αλλά από ποιον να αυτά τα στοιχεία που έχουμε, ας τα θεωρήσουμε απλές εκτιμήσεις. Είτε καταλήγουν ότι θα έχουμε να κερδίσουμε, είτε ότι θα έχουμε να χάσουμε από τη συμφωνία. Επίσης, αναφέρονται, αναφέρεται και η απώλεια θέσεων εργασίας και χτες σε αυτό το συμπόσιο που προέδευσα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μίλησε για το Ταμείο Παγκοσμιοποίησης που είναι ένα από τα εργαλεία που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για να παρέμβει κανείς. Έχω, έχω να πω ότι μια που κατά τα δύο τρίτα συρρυκνώθηκε το Ταμείο μακάρι να μπορέσει να χειριστεί τα τρέχοντα. Πού να προφτάσει το Ταμείο να καλύψει για τις συνέπειες του TTIP. Είδατε τι έκανε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πάντω, αν θέλουμε κάτι να κάνουμε για την απόλυτη θέση εργασία, θα πρέπει να ζητήσουμε παλού βοήθεια και όχι από το Ταμείο Παγκοσμιοποίηση. Επίση, χτε συζητήθηκε το τι είδου θέσει εργασία θα πρέπει να προσδοκούμε. Η Κομισιόν επ' αυτού είπε ότι υπάρχουν κάποιοι κλάδοι όπως ο εξαγωγικός ε, και εκεί μπορεί να προκύψουν ποιοτικές θέσεις εργασίας. Εντάξει, συμφωνώ. Αλλά από την άλλη μεριά, πρόσφατα, από τα στοιχεία της Κομισιόν, δεν προκύπτει κάτι τέτοιο, ιδίω όσον αφορά θέσεις απασχόλησης για νέους. Επίσης, μιλούμε για φιλόδοξα εμπορικά στάνταρ τα οποία να αφορούν και την ανάπτυξη. Πολύ ωραίο, πολύ ωραίο. Και στρογγυλά τα λέει αυτή η διατύπωση όπως είπε και ο κύριος Μαν, αλλά θα πρέπει, θα πρέπει αυτά όλα να τα υλοποιήσουμε. Μην είναι απλώς κάτι που χαϊδεύει τα αυτιά. Είδαμε τις ε, συμβάσεις του ILO, το θεματολόγιο, τον είπα, δεν θα κάνουν καμία κύρωση των συμβάσεων των συμφωνίων του ILO οι Αμερικανοί. Θα πρέπει πάντως να δούμε εμείς πώς θα μπορούσαμε να τρυπώσουμε κάποιες τέτοιες διατάξεις εδώ στη συμφωνία. Επίσης, ε, να ακούσω τι έχουν να πούνε οι συνάδελφοι. Γιατί να δούμε τι θα γίνει με τα εργασιακά δικαιώματα. Εκεί ανακύπτουν πάντοτε διαφορές. μιλάμε για ίση μεταχείριση των επενδύσεων. Είναι θέματα στα οποία κολλάμε πολλές φορές. Πολλά θέματα, ιδίω για τα εργασιακά δικαιώματα. Τώρα, για να δούμε όσον αφορά τι κοινωνικέ διατάξει και τα εργασιακά, αυτά είναι οριζόντιου χαρακτήρα. Θα πρέπει όλα αυτά να ενταχθούν εδώ πέρα. Όλα αυτά θα είναι στο εκτελεστικό ούτω ή κομμάτι τη συμφωνία και έχουμε και το θέμα τη βιωσιμότητα, τη βιώσιμη ανάπτυξη τέλο πάντων, που και αυτό θα πρέπει να καλυφθεί η κοινωνία των πολιτών, κοινωνική εταίρη αυτοί θα πρέπει να εμπλακούν. Ξέρω, ξέρω πιέζει ο χρόνος, δεν θα με κρηγορήσω άλλο. Επίσης αναφέρομαι για το ότι θα πρέπει να περιφρουρήσουμε, λέω πλήρως, να περιφρουρήσουμε το δικαίωμα των κρατών μελών να ε, νομοθετούν για τις κρατικές υπηρεσίες όπως επίσης και για τις διατάξεις ασφαλείας. θα πρέπει πάνω απ' όλα να υπάρχει σαφήνεια στις ρυθμίσεις. Πρόκειται για εμπορική συμφωνία ιδιαίτερη σημασία και χρειάζεται να κάνουμε κάποιο είδου θετική απαρίθμηση το τι θέλουμε να μπει και αρνητική τι δεν θέλουμε να μπει. Πάντα υπάρχει μια φαιά ζώνη και ξέρετε τι σημαίνει με τις ε, φαιές ζώνες στο τέλος. Άρα, εγώ θεωρώ ότι όταν έχουμε μια θετική απαρίθμηση, αυτό θα άρει τις ασάφειες. Να δούμε τι θα γίνει με τις ρήτρες, με τις σταθερότητας, stand still, που βοηθούν και θα πρέπει και εμείς και οι συνομόδιες επιτροπέ όλε να βρουν λύσεις όπου χρειάζεται. Όπως σα είπα, μελέτησα τι είπε για το ISDS, η ερευνητική μα υπηρεσία. Και από το 1994 μέχρι το 2012 ε, ε, είχαμε τρομερή αύξηση. Το μεγαλύτερο μέρος της χώρας της Αμερικής αλλά και ένα μεγάλο μέρος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι πολύ ενδιαφέρον να δούμε ότι είναι 59 περιπτώσεις μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Οπότε έχουμε και τέτοια προβλήματα. 8 εκατομμύρια δολάρια κοστίζει η τυπική περίπτωση διαιτησίας και έχουμε φτάσει ένα σημείο που έχουμε και χρηματοδότηση από τρίτες πηγές. Δεν το πίστευα αυτό μέχρι να το διαβάσω στο έγγραφο του Κοινοβουλίου, όπου τράπεζες και επενδυτικά ταμεία και ταμεία αντισταθμίσματος ε, επενδύουν σε αυτές τις περιπτώσεις μεταξύ 15 20% από το τελικό αποτέλεσμα είναι το αντίτιμο της επένδυσής τους. Αυτό το οποίο συμβαίνει εδώ δεν είναι παραδεκτό πλέον και παρά το, πέρα από το γεγονός ότι το ISDS θα εμποδίσει τη ρύθμιση από τις κυβερνήσεις είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να το λύσουμε. Εγώ περιμένω να ακούσω τι έχουν να πούν οι συνάδελφοι για όλα αυτά τα θέματα λοιπόν και φυσικά να συνεργαστώ και με τους εισηγητές. Σας ευχαριστώ για την πάρα πολύ ενδιαφέρουσα εισαγωγή στη συζήτησή μας για το θέμα αυτό. Θα δώσω το λόγο στη Ρωμάνα Τόμψ από το EPP, από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ πολύ κύριε, κύριε Πρόεδρε. Πρώτα απ' όλα, να ευχαριστήσω την εισηγήτρια την κυρία Χάρκιν για το έργο που έχει φέρει σε πέρας. Προφανώς είναι ιδιαίτερα ευρύ θέμα το θέμα του, της TTIP, ένα πάρα πολύ σημαντικό ζήτημα το οποίο θα επηρεάσει τη ζωή και την εργασία των ανθρώπων μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα υπάρξουν επιπτώσεις σε όλα τα κρατημέλη. Και νομίζω σε Κοινωνική Επιτροπή και Επιτροπή Αναπασχόλησης θα πρέπει να επιληθούμε αυτού του θέματος και θα πρέπει να εξασφαλίσουμε φυσικά ότι τα ευρωπαϊκά πρότυπα δεν θα υποβαθμιστούν ή τουλάχιστον να μην υποβαθμιστούν ιδιαίτερα. Γιατί θεωρούμε ότι τα πρότυπά μας είναι ιδιαίτερα θετικά και κατάλληλα θα πρέπει όλοι να αγωνιστούμε για να εξασφαλίσουμε τη διατήρηση αυτών των προτύπων. Η Επιτροπή μας είναι από τις σημαντικότερες για τον τομέα αυτό και μπορούμε λοιπόν να βοηθήσουμε την αρμόδια επιτροπή στο θέμα αυτό, να δώσουμε μια σημαντική συνεισφορά στο θέμα αυτό για να αντιμετωπίσουμε λοιπόν αυτό το πρόβλημα με τις συστάσεις μας. Έρχομαι λοιπόν τώρα συγκεκριμένα στη γνωμότητα της κυρίας Χάρκη μας εξήγησε ποιο είναι το σημείο κίνησης της και συμφωνώ με αυτά τα οποία είπε. Θα είναι απαραίτητο στη συνέχεια να κάνουμε και κάποιες προσθήκες στη γνωμοδότησή της, να κάνουμε κάποιες διευκρινήσεις και πιστεύω ότι υπάρχουν και περαιτέρω σημεία τα οποία θα έπρεπε να ληφθούν υπόψη μέσα σε αυτή τη γνωμοδότηση. Η πολιτική μας ομάδα θα τα εξετάσει όλα αυτά ενδελεχέστερα, αλλά Θέλω να υπογραμμίσω ορισμένα σημεία ήδη τώρα, τα οποία εμείς χαιρετίζουμε στην έκθεση της κυρίας Χάρκιν. Είναι πάρα πολύ καλό πρώτα απ' όλα να αναφερθεί το γεγονός ότι η συμφωνία TTIP θα πρέπει να δημιουργήσει νέες θέσεις απασχόλησης. Εγώ Νομίζω ότι αυτό είναι έγκυρο. Άκουσα αυτά τα οποία είπε η κυρία Χάρκιν. Αλλά μας είπε η κυρία Χάρκιν ότι θα μειωθεί η απασχόληση ενδεχομένως στην περίπτωση της εφαρμογής του TTIP. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει εδώ να έχουμε μια πιο ε, αισιόδοξη αντιμετώπιση. Θα πρέπει να ε, ξάρουμε και τον θετικό ρόλο που μπορούν να διαδραματίσουν οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Όλοι θεωρούν ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις είναι σημαντικές για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Υπάρχει ήδη ένα μεγάλο ποσοστό της απασχόλησης στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και επομένως θα πρέπει να ληφθεί αυτό υπόψη. Επιπλέον θα πρέπει να σκεφτούμε και τι σημαίνουν τα πρότυπα του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας που εξασφαλίζουν την ε, υγεία, την ασφάλεια, την ε, μονιμότητα των θέσεων εργασίας και γι' αυτό το λόγο θα πρέπει και αυτό να ληφθεί υπόψη. Η εταιρική ευθύνη των επιχειρήσεων, η κοινωνική ευθύνη μάλλον των επιχειρήσεων θα πρέπει και αυτή να αναφερθεί καθώς και το δικαίωμα των κρατών μελών για τη διατήρηση υπηρεσιών κοινωνικού ωφέλους και την διατήρηση αυτονομίας της αποφάσης στον τομέα αυτό. Θα ήταν βέβαια πάντα δυνατόν να επιφέρουμε κάποιες βελτιώσεις και θα πρέπει να θέσουμε το ερώτημα του τι θέλουμε σε σχέση με την επίλυση διαφορών μεταξύ επενδυτών <clears throat> και κρατών. Να έχουμε ένα θετικό και αρνητικό κατάλογο για αυτές τις διαδικασίες. Και εγώ συμφωνώ με την κυρία Χάρκιν ότι είναι απαραίτητο να έχουμε ένα θετικό κατάλογο σε αυτή την περίπτωση. Η TTIP θα οδηγήσει σε μια απελευθέρωση των αγορών, σε ένα μεγαλύτερο άνοιγμα των αγορών, επομένως θα υπάρχουν θετικά αποτελέσματα από αυτή την άποψη. Από την άλλη πλευρά όμως θα κάνει πιο ευάλωτες τις ε, οικονομικές και κοινωνικές δομές. Θα πρέπει η Επιτροπή μας να εξασφαλίσει ότι τα δικαιώματα και τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ιδίως σε αφορά τις πιο ευε, και ευάλωτες ε, ομάδες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και συγκεκριμένα τα δικαιώματα των εργαζομένων, οι οποίοι βρίσκονται σε μεγάλες επιχειρήσεις, θα διατηρηθούν και επίσης το επίπεδο κοινωνικής προστασίας που έχουμε αυτή τη στιγμή θα επιβιώσει. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ ο κύριος. κύριος Σούστερ. Εγώ μπορώ να συμφωνήσω σε μεγάλο βαθμό με την προηγούμενη ομιλήτρια. Εμείς βλέπουμε πόσο αμφιλεγόμενο είναι το θέμα του TTIP στην κοινή γνώμη. Είναι η πρώτη συμφωνία εμπορικού χαρακτήρα που έχει ένα τόσο μεγάλο ε, πολιτικό αντίκτυπο και γι' αυτό πράγματι αξίζει τον κόπο να προσπαθήσουμε να καταλάβουμε τι σημαίνει, τι συμβαίνει αυτή η συμφωνία. Δεν είναι ότι θα αλλάξουν τόσο πολύ οι οικονομικές μας δοσοληψίες με τις Ηνωμένε Πολιτείε λόγω αυτής της συμφωνίας. Έχουμε ήδη σήμερα μια πολύ έντονη εμπορική σχέση και οι μελέτες που έχουμε δει είναι κάπως επιφυλακτικές σε σχέση με τα θετικά αποτελέσματα που θα προκύψουν σε επίπεδο οικονομικής ανάπτυξης και ε, απασχόλησης. Και υπάρχουν και μελέτες που δείχνουν ότι θα συμβεί το αντίθετο. Γι' αυτό λοιπόν είναι απαραίτητο να λάβουμε πάρα πολύ σοβαρά το θέμα του TTIP. Το, ουσια, το ουσιαστικό εδώ είναι, νομίζω, πέραν της εμπορικής φιλελευθερωποίησης το θέμα είναι να δημιουργήσουμε <clears throat> παγκόσμια πρότυπα. Εμείς θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε αυτήν την σχέση για να μπορέσουμε να έχουμε κοινά παγκόσμια πρότυπα για την παγκόσμια οικονομία. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχει μεγάλη ανησυχία στον πληθυσμό γιατί θέλουν και περιμένουν από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς αντίστοιχα οι Αμερικανοί από το Αμερικανικό Κοινοβούλιο να προστατευτούν τα πρότυπα τα οποία ισχύουν. Γι' αυτό πρέπει να κάνουμε κάθε προσπάθεια να βρούμε τα σωστά αυτά πρότυπα. Η εναλλακτική λύση δεν είναι να οχυρωθούμε στον μικρό και όμορφο κόσμο μας. Κινδυνεύουμε να βρεθούμε σε μια κατάσταση που δεν θα υπάρχουν καθόλου πρότυπα τα οποία θα ισχύουν εν γέννη και θα συνεχίσει ένας παγκόσμιος ανταγωνισμός χωρίς χαλινούς. Η κυρία Χάρκιν έχει λοιπόν προσπαθήσει να δώσει απάντηση σε πολλά από αυτά τα ερωτήματα και εγώ θα ήθελα να επανέλθω στα ζητήματα αυτά από τη δική μας πλευρά. Ποιε είναι οι κατευθύνσει που θα πρέπει να αντιμετωπιστούν. Το πιο σημαντικό θέμα θα πρέπει να είναι να διατηρήσουμε τη δυνατότητα πολιτικής ρύθμισης και εφαρμογής των δημοκρατικών δικαιωμάτων του κρατούς δικαίου. Όλα αυτά θα πρέπει να παραμείνουν και να υλοποιηθούν μέσα σε, στη συμφωνία αυτή. Όπως είπε η κυρία Χάρκεν, υπάρχουν κίνδυνοι για αυτά τα στοιχεία σε πάρα πολλού τομεί. Και εμεί θα πρέπει να δούμε πώ μπορούμε να εξασφαλίσουμε ότι θα διατηρηθούν αυτά τα στοιχεία. Δεν πρόκειται μονάχα για τα δικαιώματα των εργαζομένων, αλλά και για κοινωνικά και περιβαλλοντικά πρότυπα. Εμεί θα πρέπει να αποφύγουμε να υποβαθμιστούν αυτά τα πρότυπα. Και από την άλλη πλευρά ξέρουμε ότι από τις δύο χτες του Ατλαντικού διαφέρουν πάρα πολύ τα συστήματα αυτά και θα είναι δύσκολο να καταλήξουμε κατά 100% σε ένα κοινό σύστημα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα των εργαζομένων. Ξέρουμε ότι οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ακολουθήσει ένα ριζικά διαφορετικό ε, δρόμο και παραγωγικά σε ό,τι αφορά την δράση των εργατικών ενώσεων και των συνδικάτων δεν ισχύουν τα ίδια στην Αμερική από ό,τι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεύτερον, το θέμα της διαιτησίας είναι σαφές ότι θέλουμε να έχουμε προστασία των επενδυτών, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο πρέπει να οδηγήσει απαραίτητα σε ένα χωριστό μηχανισμό για την επίλυση διαφορών. Μας έχει αναφέρει πολλά παραδείγματα η κυρία Χάρκιν που δείχνουν ότι αυτή η ιδιωτική διαδικασία επίλυσης διαφορών δεν είναι πάντα ικανοποιητική και φύγεται η αρχή της ισότητας εναντί των δικαστηρίων, ενώπιον των δικαστηρίων, χάνεται η εγγύηση της ε, διαφάνειας, χάνεται η δυνατότητα να εξασφαλίσουμε ότι δεν θα υποσκάπτεται η νομολογία των εθνικών και ευρωπαϊκών δικαστηρίων από ιδιωτικές διαδικασίες διαιτησίας. Άλλοι τομείς που αναφέρθηκαν είναι όλος ο τομέας των ε, υπηρεσιών κοινωνικού ωφέλους, όπου πολύ σωστά είπε η κυρία Χάρκεν ότι εκεί πρέπει να διατηρήσουμε τη δυνατότητα αυτή, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε τις ε, ε, ρήτρες ε, σταθερότητος και γι' αυτό αναφέρθηκε επίσης και ο θετικός κατάλογος, ο οποίος νομίζω ότι είναι πολύ λογικός. Δεν πρέπει να μιλάμε για αρνητικούς καταλόγους, θα πρέπει να καθορίσουμε με θετικούς καταλόγους ποιοι είναι οι τομείς οι οποίοι θα πρέπει να περιλαμβάνονται στη φιλελευθερωποίηση και ποιοι όχι. Ένα άλλο στοιχείο λοιπόν το οποίο δεν έχει τονιστεί ιδιαίτερα είναι το εξής. Είναι φανερό ότι μια φιλελευθερωποίηση δεν φέρνει μονάχα πλέον εκτήματα. Το ξέρουμε και από την οικονομική θεωρία, το εμπόριο δημιουργεί μια μεγαλύτερη εξειδίκευση η οποία δίδει πλεονεκτήματα σε ορισμένου τομεί, αλλά άλλοι τομεί αναγκαστικά χάνουν από αυτή τη διαδικασία και αυτό σημαίνει και απώλεια θέσεων απασχόλησης. Θέλουμε λοιπόν μηχανισμούς οι οποίοι θα απαλύνουν αυτά τα μειονεκτήματα και γι' αυτό το Ταμείο ε, Παγκοσμιοποίηση θα πρέπει να παίξει ένα σημαντικό ρόλο και θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και την διάσταση αυτού του Ταμείου, τη δυνατότητα χρηματοδότησής του Εγώ επίσης θέλω να προτείνω το εξή, επειδή οι μελέτες που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι ιδιαίτερα ικανοποιητικές και φυσικά αυτό είναι αδύρυτο, γιατί κανείς δεν ξέρει τι ακριβώς τομείς θα καλύψει το TTIP και ποιες, ε, ποιοι, ποιοι κλάδοι της οικονομίας θα επηρεαστούν περισσότερο. Εγώ θα ήθελα στη στιγμή αυτή που δεν έχουμε επαρκείς ε, γνώσεις κάποια στιγμή να ζητήσουμε να γίνει μια μελέτη η οποία θα προσπαθήσει να αντιμετωπίσει το θέμα και κατά τομείς και κατά περιφέρειες στην Ευρώπη, δει ποιες περιοχές στην Ευρώπη θα θυγούν και ποιες όχι, ώστε να μπορέσουμε τελικά να μπορούμε να ε, ζυγίσουμε τα θετικά και τα αρνητικά αποτελέσματα. Δεν μπορούμε να εμποδίσουμε τις διαθετικές αλλαγές, αλλά θα πρέπει να τις διαχειριστούμε σωστά. Και εγώ νομίζω ότι Έχουμε πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση που θα πρέπει να διεξαγάγουμε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που έλαβαν το λόγο. Για να μπορέσουμε λοιπόν να πετύχουμε μια συμφωνία, κάτι το οποίο για μένα θα ήταν θετικό, θα πρέπει να εξασφαλίσουμε και το τονίζω και πάλι ότι θα τηρηθούν αυτά τα οποία απαιτούμε σε επίπεδο δημοκρατίας και κράτους δικαίου και προσβλέπω και εγώ στις περαιτέρω συζητήσεις με την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Κυρία Μακεντάιρ. ECR. Ευχαριστώ. Πρώτα απ' όλα ευχαριστώ τη Μαριάν Χάρκιν. Την ευχαριστώ πολύ για την έκθεσή της. Είναι δύσκολο καθήκον να βάλει κανείς σε 1500 γράμματα ένα τόσο περίπλοκο θέμα. Με τις τροπολογίες βέβαια θα το συμπληρώσουμε. Σίγουρα όμως είναι μια πολύ καλή βάση πάνω στην οποία να δουλέψουμε. Θέλω να σχολιάσω τέσσερις τομείς. Πρώτον, οι ρήτρε για το ISDS, το Μηχανισμό Επίλυσης Διαφορών. Φαντάζομαι, mail παίρνουν και οι άλλοι ευρωβουλευτές που λένε να μην έχουμε ένα τέτοιο μηχανισμό, αλλά δεν νομίζω ότι δεν καταλαβαίνει το κοινό ποιος είναι ο ρόλος αυτού του μηχανισμού. Οι ευρωπαϊκές χώρες έχουν 1.400 συμφωνίες που περιλαμβάνουν τέτοιες ρήτρε μηχανισμών επίλυσης διαφορών. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, από το 1975, το Ηνωμένο Βασίλειο έχει συνάψει 94 διμερείς συμφωνίες με τέτοιες ρήτρε ISDS. Αν δείτε πώς ε, κατανέμονται, ε, θα δείτε ότι το 2000 πιο πολύ. Πολλές προσφυγές έχουν γίνει, καμία δεν έχει πετύχει. Νομίζω λοιπόν ότι είναι λογικό να πούμε ότι χρειαζόμαστε μια ρήτρα μηχανισμού επίλυσης διαφορών μεταξύ επενδυτών χωρών. Δεν πρέπει να τον φοβόμαστε. Δεύτερον, Νομίζω ότι είναι στο σημείο 5. Η κυρία Χάρκιν σωστά αναφέρεται στις ε, διασφαλίσεις που πρέπει να υπάρχουν για τις δημόσιες υπηρεσίες. Η συμφωνία ήταν με τον Καναδά, από όσο ξέρω, περιλαμβάνει μία εξαίρεση για τις δημόσιες υπηρεσίες το σύστημα υγείας, για παράδειγμα, γιατί πολλοί αναφέρθηκαν στο Βρετανικό σύστημα υγείας. Θα μπορούσε λοιπόν να υπάρχει κάτι τέτοιο και για άλλες δημόσιες υπηρεσίες, έτσι ώστε οι δημόσιες υπηρεσίες στο 5, το βλέπω, να αναφέρονται σε κάτι το οποίο ελέγχουν οι χώρες μέλη. Επίσης, συμφωνώ που θέλουμε να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις. Υπάρχει ένα δυσανάλογο εφέ πάνω στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις των δασμολογικών και μη δασμολογικών ε, μέτρων. Εκεί που διαφωνώ είναι στην παράγραφο 9 Εγώ θα προτιμούσα μια αρνητική απαρίθμηση και όχι θετική απαρίθμηση. Στη ΣΥΤΑ με τον Καναδά για παράδειγμα έτσι είναι. Ευχαρίστως να το συζητήσουμε παρετέρω, αλλά προς το παρόν δεν συμφωνώ με αυτό που αναφέρεται εδώ στο νέο. Κατά τα άλλα, προσβλέπω και εγώ σε συνεργασία με την Μαριάν και ελπίζω να καταλήξουμε σε μια καλή γνωμοδότηση από της Επιτροπής μας. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Μην μακάρι δεν είναι εδώ. Από την ΚΟΕ. Κάντι Μαντέλη. Από τους Πρασίνους. Ούτε. Τιτσιάνα. Πέκερ λοιπόν από το EFTD. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να ευχαριστήσουμε πρώτα πρώτα την εισηγήτρια για το έργο της. Θα είμαι είναι πάρα πολύ σημαντικό ότι είμαστε εδώ πέρα ε, στην Επιτροπή αυτή, αλλά επίσης εργάζομαι και στην Επιτροπή για το τύπος ε, σκιώδης ηγητρία. Οπότε έχω επισέλθει στις λεπτομέρειες του θέματος, αλλά σήμερα ας ε, εστιάσουμε την προσοχή μας στα ζητήματα που αφορούν τη δική μας Επιτροπή. Να αρχίσω με ένα πραγματικό γεγονός. Η έκθεση επιπτώσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το TTIP λέει ότι θα υπάρξουν θετικά, αλλά υποτιμούνται τα αρνητικά σημεία τα οποία θα προέλθουν και θα αφορούν την οικονομία μας. Ξέρετε ε, ποια είναι η σκοτεινή πλευρά, αλλά ακούστε τι λέει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Λέει συχνά ότι θα υπάρξουν πολλά θετικά κέντρο ε, οικονομικής έρευνας προέρχονται αυτά τα στοιχεία, αλλά δεν αναφέρεται κάτι άλλο. Δεν αναφέρονται επομένω οι απώλειες θέσεων εργασίας. Και λέει επομένω αυτό το κέντρο οικονομικής έρευνας, λέει ότι θα έχουμε 1.300.000 θέσεων απασχόλησης που θα χαθούν λόγω του TTIP. Και ε, αυτό θα αφορά την κατάργηση του 80% των δασμών, κάτι το οποίο ε, βέβαια είναι πάρα πολύ φιλόδοξο. Και πώς θα βρουν δουλειά όλοι αυτοί. Αυτοί δεν θα μπουν στο περιθώριο. Δεν είναι να μάθουμε τις απαντήσεις γιατί το οικονομετρικό μοντέλο αυτής της ανάπτυξης προβλέπει μεταξύ των άλλων να υπάρξει σταθερή προσφορά εργασίας. Σύμφωνα με την οικονομική επιστήμη ε, λένε ότι πάντοτε θα υπάρξουν ε, μεσοπρόθεσμα αποτελέσματα προσαρμοστικά και μακροπρόθεσμα τα θετικά αποτελέσματα. Δηλαδή τι είναι. Είναι η αγοραστική δύναμη που θα μειωθεί των οικογενειών και το εισόδημα το οποίο θα απολυστεί. Το δέχθηκε αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα έχουμε πλήγμα στην απασχόληση θα χαθούν θέσεις εργασίας σε κάποιους κλάδους χωρίς αναγκαστικά να αυξηθούν θέσεις απασχόλησης σε άλλους κλάδους. Τι θα γίνει με τις ΜΜΕ. Εμείς ποντάρουμε σε αυτές να βγούμε από την κρίση. Θα τις εκπλήξει το TTIP και διάφορες ανεξάρτητες μελέτες λένε ότι θα πέσει το 40% ε, το ενδοκινοτικό εμπόριο και ανταυτού θα έχουμε αύξηση του εμπορίου στις Είπα, θα χάσουμε επομένω εμπόριο, ε, ας πούμε με, τη, με κάποια γαλλική εταιρεία, κάποιες ανταλλαγές, γιατί θα γίνονται αυτές τώρα πια με τους Αμερικανούς. Πού είναι αυτά τα κέρδη, μα δεν βλέπετε ότι το TTIP το θέλουν οι μεγάλες επιχειρήσεις. Οπότε λέμε ότι τώρα θα έχουμε πρόσβαση σε μεγάλους ε, τομείς της αμερικανικής οικονομίας. Μην πιστεύετε αυτά τα μεγάλα λόγια, λέω εγώ. Επομένως, πάρα πολλοί θα χάσουν τη δουλειά τους. Και άρα θα πρέπει εμείς εδώ να κάνουμε ό,τι μπορούμε όταν ψηφίζουμε και αποφασίζουμε για την ενίσχυση από το ε, Ταμείο Αποκλεισμοποίησης. Ναι, αλλά τι θα γίνει αν έχουμε κάποιο νομοθέτημα που δεν αρέσει σε κάποιον Αμερικανό, α πούμε, για την απασχόληση, θα πρέπει να τον αποζημιώσουμε. Άρα, να κοίταξτε τι γίνεται στον ναύτα. Αντί για 55.000 θέσει απασχόλησης που είχαν υποσχεθεί, χάθηκαν ένα εκατομμύριο και δύο εκατομμύρια ε, στο, στη, στη, στη Γεωργία, γιατί τώρα εκεί είναι οι μεγάλες εταιρείες που κυριαρχούν. Στη δική μας περίπτωση οι ΙΠΑ έχουν τελείως διαφορετικές διαστάσεις, ιδίως όσον αφορά τις συλλογικέ διαπραγματεύσεις. Η προστασία του εργαζομένου είναι πολύ μικρότερη, αυτό αφορά και την υγεία και τις συντάξεις. Επίσης για την θέμα του ανταγωνισμού θα έχουμε κοινωνικό dumping. Πώς θα εμποδίσουμε τους Αμερικανούς με αυτή τη συμφωνία πρόκειται να χαμηλώσει ο πύχης. Τι θα είναι εργαζομένου. Θα πρέπει να τα λάβει όλα αυτά υπόψη η, η Η Πρόεδρος, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε και την εισηγήτρια και τους κοιόδης εισηγητές. Τώρα, να δούμε ποιοι έχουν ζητήσει το λόγο. Είναι πολλοί και παρακαλώ να τηρήσετε ένα δίλεπτο έκαστος για να μπορέσουμε να τα καταφέρουμε. Η κυρία Αρένα έχει πρώτη λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Όπως και η προλαλήσασα και εγώ εργάζομαι στην ε, Επιτροπή ΙΝΤΑ. Εδώ όμως να δούμε τα θέματα απασχόλησης και ποιότητας απασχόλησης. Είναι αλήθεια ότι για το TTIP έχουμε κάποιες μελέτες επιπτώσεων. Τα έχει κάνει αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και Έχουμε κάποια μοντέλα μακροοικονομικά, κάποια μοντέλα τα οποία μας οδηγούν στο ότι θα υπάρξει κάποιο κέρδος για την Ευρώπη. Ε, έχουμε κάποιο απελευθέρωση στο εμπόριο με τη ΣΥΠΑ. Για να δούμε επίσης την ανάλυση των μοντέλων που χρησιμοποίησαν αυτές οι μελέτες. Η αφετηρία των μελετών είναι το ότι υπάρχει μια γεωγραφική, επαγγελματική και τομεακή κινητικότητα των εργαζομένων. Δηλαδή, μία χώρα πάει καλά και αναδέχεται στους ορισμένους χώρες που δεν τα πάει καλά. Δεν λέω ονόματα, φεύγουν επομένως από την α χώρα και μας στη β χώρα. Οπότε υπάρχει και επίση ένας τομέα που πάει καλά και δέχεται εργαζομένου από τομέα που δεν τα πάει καλά και κάποιοι που χάνουν τη δουλειά τους να πάνε σε κάποια άλλη ε, επιχείρηση. Όλα αυτά τα λέει η θεωρία. Πολύ ωραία. Αλλά στην πράξη δεν είναι έτσι τα πράγματα. Η γεωγραφική, η επαγγελματική και η τομιακή κινητικότητα δεν λειτουργούν τόσο απλά. Και έχουμε τις μελέτες, Αλένα, που βασίζαν στο ίδιο μοντέλο και κατέδειξαν στο ότι εκεί που βγήκε ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας, 20 χρόνια μετά Είχαμε άλλες μελέτες που λένε ότι έγινε απώλεια 700 θέσεις εργασίας. Άρα έχουμε τρομερή απώλεια θέσεων εργασίας λόγω της συμφωνίας. Όμως είχαμε ζημία και στην ποιότητα εργασίας δηλαδή οι, εργαζόμενοι μετακινήθηκαν προς το Μεξικό ε, με την Ελενά, με την Ναύτα πήγανε προς προς το Μεξικό, ας πούμε, εκεί που υπάρχει λιγότερο προστασία εργαζομένων. Επομένως, εμείς ε, ήδη έχουμε συναλλαγές με τις ε, είμαστε οι πρώτοι σε, αυτό, αλλά τι θα γίνει με τους εργαζομένους. Τώρα κάτι άλλο για τις επενδύσεις και το ISDS. Έχουν ε, διατυπώσει κάποιες ε, ε, επικρίσεις, αλλά μια που έχουμε εδώ δικαιοδοτικά όργανα, Μα έχουμε επενδύσει αμερικανικέ ήδη στην Ευρώπη και προσφεύγουν στη δικαιοδοσία την ευρωπαϊκή. Δεν είναι τίποτα τέλειο, αλλά αυτού του είδου την δημοσία κρατική δικαιοσύνη να την αντικαταστήσουμε με δικαστικά όργανα, διαιτητικά όργανα, ε, ιδιωτικά. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να μείνουμε αυτό το οποίο έχουμε και να μην μπει ο λύκος στο Μαντρί. Γιατί δεν θα υπάρχει ε, διαφάνεια, θα είναι ιδιωτική αυτή η φορής και θα υπάρχει φοβερή χειραγώγηση. Αλλά εγώ δεν θεωρώ ότι θα πρέπει ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών να μπει στο TTIP. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Κύριε Μάνου Ευχαριστώ. Δύο λεπτά είναι δύσκολο βέβαια να τα καλύψω αυτά που θέλω να πω. Εγώ νομίζω ότι μας δίνει τη δυνατότητα να κερδίσουμε κάτι η TTIP δεν είναι μονάχα μια συζήτηση που γίνεται και κλεισμένο των θυρών. Είναι πιο ανοιχτά πια τα πράγματα. Έχουμε κάνει και ακροάσεις στην Επιτροπή μας και είναι σαφές ότι και με την έκθεση Ταραμπέλα έχουμε και τη δυνατότητα να υπάρχουν και παρεμβάσεις όλων αυτών που ενδιαφέρονται για αυτό το θέμα. Χαίρομαι λοιπόν για αυτό το θέμα. Και εμείς έχουμε κάνει στην εκλογική μου περιφέρεια ε, εκδηλώσεις οι οποίες πληροφορούν τον πληθυσμό. Όλα αυτά είναι πάρα πολύ θετικά λοιπόν. Είναι επίσης και οι απόψεις των ε, ε, εργαζομένων και των περιβαλλοντολόγων οι οποίοι συμμετέχουν στο συμβούλιο το οποίο έχουμε δημιουργήσει για την TTIP. Επομένως, επιτέλους καταφέρουμε να έχουμε κάτι το οποίο είναι ουσιαστικό, να υπάρχει η γνώση για την κοινία των πολιτών. Θα θέλουμε και εμείς, πρέπει και εμείς λοιπόν να εξασφαλίσουμε ότι θα πρέπει να εστιάσουμε στα ουσιαστικά στοιχεία. Εμείς τονίζουμε καταρχήν την ανάγκη να διατηρηθεί η προστασία της εργασίας στην Ευρώπη. Πρέπει όμως όλες οι αιτήσει που έχουμε να γίνουν συγκεκριμένες. Είναι απαραίτητο να έχουμε τα σωστά πρότυπα τα οποία θα ε, διατηρηθούν. Εμείς μέχρι στιγμής δεν έχουμε κάνει όλα αυτά που κάνουμε για να πούμε όχι δεν θέλουμε φιλελευθερωποιημένη αγορά αλλά θέλουμε να έχουμε την προστασία των προϊόντων που είναι, που είναι σημαντικά για μας. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια στρατηγική η οποία θα είναι ουσιαστική και όχι μονάχα μια απόρριψη. Ε, έχει αναφερθεί πολλές φορές η κοινωνική εταιρική ευθύνη. Αυτά είναι θέματα τα οποία παραμένουν σε ένα θελοντικό επίπεδο αλλά θέλουμε να υπάρξει μια πραγματική δέσμευση και από την άλλη πλευρά των επιχειρήσεων. Νομίζω λοιπόν ότι με όλα αυτά τα μέτρα θα μπορέσουμε να προχωρήσουμε με θετικό τρόπο και η δική μας Επιτροπή βέβαια δεν είναι η επικεφαλής αλλά πρέπει οι συστάσεις μας να ληφθούν υπόψη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπαχ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Και εγώ θέλω να ευχαριστήσω εκ βάθους καρδίας τη Μαριάν Χάρκιν και να τη συγχαρώ για την έκθεσή της. Είναι πιστεύω μια έκθεση η οποία έχει ένα πολύ θετικό χαρακτήρα. Χαιρετίζω επίσης τις σαφείς δηλώσεις της σε σχέση με την ε, διαπραγμάτευση που λαμβάνει ε, χώρα αυτή τη στιγμή. Έχουμε ενώπιόν μας μια πολύ μεγάλη πρόκληση και είναι δύσκολο για πολλά κράτη-μέλη να έχουν μια θετική εικόνα για τις διαπραγματεύσεις της TTIP. Επίσης έχουν ε, λεχθεί πάρα πολλά και δεν χρειάζεται να τα καλύψω όλα για τον θετικό ή αρνητικό κατάλογο. Εγώ πιστεύω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπάρξει ένας τέτοιος κατάλογος Δεν μπορούμε εδώ να προσθέσουμε ένα νέο θέμα στις διαπραγματεύσεις γιατί οι διαπραγματεύσεις έχουν ήδη το θεματολόγιο τους. Και επομένως θα πρέπει να στραφούμε προς την Κομισιόν να μας δώσει μια μεγαλύτερη σαφήνεια στο θέμα αυτό. Και επίσης η αρχή της, ε, των υπηρεσιών κοινή ωφελία δεν έχουν λεχθεί πάρα πολλά εδώ θα πρέπει να γίνει κατανοητό και από τους Αμερικανούς ότι αυτό είναι μια επίτευξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης η οποία θα πρέπει να διατηρηθεί. Και τέλος κλείνοντας, πιστεύω ότι εμείς ως Ευρώπη να διατηρήσουμε τον παγκόσμιο ρόλο μας. Θα πρέπει λοιπόν να παίξουμε ένα ενεργό ρόλο στις διαπραγματεύσεις οι οποίες θα διαμορφώσουν πρότυπα. Με όλα τα προβλήματα τα οποία μπορεί να υπάρχουν, αλλά εμείς θα πρέπει να μην υποχρεωνόμαστε να τηρούμε πρότυπα, να πρέπει να, συνδιαμορφώσουμε κι εμείς πρότυπα για το παγκόσμιο εμπόριο, αλλιώς κινδυνεύουμε να αποκλειστούμε από το παιχνίδι. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πυρίνσκι, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Χάρκιν, παρουσιάζοντάς μας την θέση της, περιγράφει συνολικά τα ωφέλη, αλλά και τις αμφιβολίες που υπάρχουν. Χτες στην ακρόαση που είχαμε, ένα πράγμα κατέστη σαφές, ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει σκεφτεί τον αντίκτυπο της συμφωνίας σε διάφορες μεμονωμένες χώρες, κυρίως στην Νότια και Νοτιοανατολική Ευρώπη. Ερωτήθηκε και εκπρόσωπος της Επιτροπής από πρόσωπο της Ουγγαρίας και απάντηση ήταν ότι δεν έχουν σκεφτεί τον αντίκτυπο αυτό σε αυτές τις χώρες. Και αυτό με φέρνει σε κάτι γενικότερο, κύριε Πρόεδρε. Η συμφωνία αυτή άρχισε διμερός πριν από πολλά χρόνια από μία ομάδα εργασίας ως συμφωνία υπέρ της ανάπτυξης και της απασχόλησης για να βγούμε ακριβώς από την κρίση. Και σιγά σιγά κατέληξε σε κάτι μεγαλύτερο. Μία διάσταση ενισχύει την διατλαντική εταιρική σχέση μέσα σε έναν κόσμο που αλλάζει και συγχρόνως προσπαθεί να καθορίσει προδιαγραφές για την παγκοσμιοποίηση η ανησυχία που εκφράζεται στις χώρες μας έχει να κάνει ακριβώς με την αίσθηση των πολιτών μας ότι δεν πρόκειται μόνο για το εμπόριο και ότι είναι κάτι το οποίο απειλεί το βασικό κοινωνικό ευρωπαϊκό μοντέλο. Αν λοιπόν θέλουμε να ενισχύσουμε τις διαδραντικές σχέσεις, πιστεύω ότι πρέπει να πιέσουμε όσο γίνεται περισσότερο υπέρ επενδύσεων, απασχόλησης και να μην Είμαστε υπερβολικά φιλόδοξοι νομίζοντας ότι θα φτιάξουμε ένα σύστημα που θα αλλάξει τον κόσμο. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, εμείς σας ευχαριστούμε. Τζιν Λάμπερτς. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω εκ μέρους της σκιώδης μας, της Καρεντέλη. Ε, φυσικά και συμφωνούμε και εμείς με πολλές από τις ανησυχίες που ακούσαμε εδώ σήμερα. Το θέμα της ανάπτυξης και της απασχόλησης, για παράδειγμα δεν είναι αυτόματο και τι θα γίνει και με την ε, κατανομή. Επίσης, συμφωνούμε με τις ανησυχίες που εκφράζονται σε διάφορες μελέτες που έχουν γίνει μέχρι τώρα. Τα είπε και ο συνάδελφος πριν από λίγο για το τι μπορεί να σημαίνει μια τέτοια συμφωνία για κάποιες χώρες και για κάποιους κλάδους. Είναι κάτι που δεν το έχουμε προσέξει αρκετά ή και καθόλου. Συμμεριζόμαστε επίσης πολλές από τις ανησυχίες που εκφράστηκαν όσον αφορά τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών. Είναι κάτι το οποίο δημιουργείται μεταξύ δύο πλευρών που έχουν όμως πολύ ισχυρά δικαστικά συστήματα. Και από τη χώρα μου έχουμε ακούσει ότι Κάτι από αυτά που κρύβεται δεν είναι τόσο το τι θα κάνουν οι Ηνωμένες σε ομοσπονδιακό επίπεδο, αλλά σε επίπεδο <coughs> πολιτιών και δικαστηρίων στις πολιτείες των Ηνωμένων Πολιτειών. Τελικά θα βρεθούν σε δύσκολη θέση οι ευρωπαϊκές χώρες και γι' αυτό λένε να έχουμε ένα τέτοιο μηχανισμό χωρίς να λαμβάνεται υπόψη το νομικό καθεστώς κατά περίπτωση. Μη συμφωνήσουμε λοιπόν με κάτι το οποίο επιτρέπει ιδιωτικά συστήματα σε αντιπαράθεση με τα εθνικά. Γι' αυτό συμφωνούμε και εμείς με αυτούς που θέλουν και ζητούν περισσότερη ενημέρωση. Όσον αφορά τη θετική απαρίθμηση, θα έχουμε μία τροπολογία που θα επεκτείνει την ιδέα αυτή και συμφωνούμε και με όσα αναφέρονται για τον αποκλεισμό κάποιων δημοσίων υπηρεσιών. Υπάρχει και στην οδηγία τη δικιά μας για τις δημόσιες υπηρεσίες, αλλά δεν είχαμε ικανοποιητική λύση για τον τρόπο με τον οποίο θα προστατεύονται κάποιες δημόσιες υπηρεσίες και θα συμπεριλαμβάνονται συγχρόνως εδώ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση λοιπόν πρέπει να προσπαθήσει να κάνει κάτι αντίστοιχο και εδώ. για την ε, μετακίνηση των εργαζομένων. Εδώ βέβαια υπάρχουν ανάμεικτα συναισθήματα και απόψεις. Είναι πολύ δύσκολο να πεις σε κάποιον ότι δεν θα μπορέσει να μετακινηθεί σε άλλη χώρα επειδή απασχολείται σε ένα συγκεκριμένο τομέα. Επηρεάζονται τα επαγγελματικά και τα προσωπικά τους δικαιώματα. Αλλά αυτό βέβαια μας φέρνει στην αμοιβαία αναγνώριση προσόντων, το οποίο δεν έχει προχωρήσει αρκετά μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτές λοιπόν είναι κάποιες από τις ανησυχίες που έχουμε σε σχέση με την απασχόληση. Η Μάριαν Χάρκιν ίδια αναφέρεται στην εργασιακή νομοθεσία, στη γνωμοδότησή της. Πράγματι και εμείς θέλουμε περισσότερα αποτελέσματα εδώ και τις συστάσεις του Διεθνούς Γραφείου Εργασίας να συμπεριληφθούν εδώ στην περίπτωση που η συμφωνία αυτή ολοκληρωθεί κάποτε. Ευχαριστώ. Πρόεδρος, ευχαριστούμε πολύ. Τζιν Λάμπερτς που μιλήσατε εκ μέρους της σκιώδους εισηγήτριας των Πρασίνων, έτσι. Τώρα, επιστρέφουμε στα δύο λεπτά ο καθένας. Παρακαλώ, Άγκελε. Ευχαριστώ πολύ. Έχω κάποιες αμφιβολίες. Η συμφωνία αυτή υποτίθεται ότι θα μας δώσει περισσότερες θέσεις απασχόλησης. Αλλά οι εμπορικές συμφωνίες δεν υπογράφονται για να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας. Λογικά έχουν σαν στόχο να απλοποιήσουν το εμπόριο και να το διευκολύνουν και να δώσουν περισσότερα κέρδη στους εμπορευόμενους. Τα κέρδη μπορούν να αυξηθούν πολύ πιο εύκολα με το να μειωθεί ο αριθμό των εργαζομένων. Δεν κερδίζετε με το να αυξάνετε θέσεις απασχόλησης και με το να δίνετε περισσότερες αμοιβέ στους εργαζομένους. Λέγεται επίσης ότι θα αυξηθεί το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης από αυτή τη συμφωνία. Ακόμα και αν αυτό γίνει, και εδώ αμφιβάλλω, ακόμα και αν αυξανόταν το ΑΕΠ της Ευρωπαϊκής Ένωσης Καμία εμπορική συμφωνία δεν θα εξασφαλίσει ποτέ ότι ο αυξανόμενος πλούτος θα διανεμηθεί ισόρροπα σε όλο τον πληθυσμό. Δεν υπάρχει αναδιανεμητικός μηχανισμός ο οποίος να εμπεριέχεται σε μια συμφωνία εμπορικού χαρακτήρα. Ακόμα και να αυξηθεί το, ε, το ΑΕΠ δεν υπάρχει καμιά εγγύηση ότι τα κέρδη από αυτή τη συμφωνία δεν θα παραμείνουν στα στις τσέπες των μεγαλοκαρχαριών και των μεγαλοεπενδυτών. Αν αυτή η συμφωνία λοιπόν εγκριθεί, θα ισχύει για πάντα. Δεν θα μπορούμε να την ξεπεράσουμε. Αλλά τι θα γίνει αν αυτή η εμπορική συμφωνία δεν δώσει τα ωφέλη τα οποία υποτίθεται ότι θα δώσει. Τι θα γίνει αν δεν δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης. Τι θα γίνει αν δεν αυξηθεί η ευμάρεια. Τι θα γίνει αν θα δώσει μονάχα κέρδη στους μεγαλοεπενδυτές και στους μεγαλοκαρχαρίες. Ευχαριστώ λέει η Πρόεδρος ο Τανούτα Γιάσλοβιέσκα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω και εγώ, αλλά και να συγχαρώ την Μαρία Η έκθεσή της είναι κλήρης και μας παρουσίασε επίσης και πολύ ζωντανά τα πράγματα. Η Τζιν Λάμπερτ αναφέρθηκε στην αναγνώριση των δεξιοτήτων και των ε, διπλωμάτων και θέλω επ' αυτού να πω ότι θα πρέπει να έχουν ίση μεταχείριση όλοι οι πολίτες της ε, Ένωσης γιατί υπάρχουν κάποια κράτη-μέλη των οποίων οι πολίτες θα πρέπει να πάρουν βίζα για να πάνε στη ΣΥΠΑ. Όταν τεθεί σε ισχύ το TTIP αυτές οι χώρες, αυτοί οι άνθρωποι θα έχουν μεγάλο πρόβλημα. Παρακαλώ αυτόν τον λάβει υπόψη. Μάριον και έχω υποβάλει σχετική ε, τροπολογία. Ο κύριος Σούστερ. Σούλτσε, sorry. Σούλτσε, Σούλτσε, συγγνώμη. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Λίγα είναι δύο λεπτά είναι η πρώτη φορά που μέχρι τώρα δεν έχουν μιλήσει οι πράσινοι σε μια συνεδρίαση για το TTIP. Εγώ δεν θέλω να επαναλάβω όλα αυτά τα θετικά που ελέγχθηκαν, μόνο σε δύο σημεία να αναφερθώ. Εγώ ε, μπορώ να συμφωνήσω με πολλά από αυτά που ελέγχθηκαν. Θέλω να επαναλάβω ότι αυτό είναι ένα θέμα που συζητείται σε πάρα πολλές ε, επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και αυτό είναι σημαντικό για την ε, διαφάνεια. Δεν μπορούμε λοιπόν να έχουμε όλα τα στοιχεία και για τον ε, κύριο Σούστερ θα ήθελα να πω είναι μία από τις συμφωνίες για τις οποίες έχει γίνει η μεγαλύτερη συζήτηση. Είναι μία συμφωνία λοιπόν για την οποία όμως έχει υπάρξει μεγάλη παραπληροφόρηση στην ε, κοινή γνώμη από τα μέσα ενημέρωσης. Έχουν ελεγχθεί πράγματα τα οποία δεν ευσταθούν και το τονίζω και πάλι μετά από αυτά που είπα από τη συνάδελφο του FTD. Δεν νομίζω ότι μπορώ να συμφωνήσω με όλα αυτά τα πράγματα. Είναι αποτέλεσμα παραπληροφόρησης αυτά τα οποία λέγονται. Ένα σημείο τώρα θέλω να τονίσω πάντα για το TTIP. Το θέμα των θέσεων εργασία. Λέγεται ότι θα πρέπει να εξασφαλίσουμε να δημιουργηθούν περισσότερε θέσει εργασία και καλύτερε θέσει εργασία. Εγώ έρχομαι από τον οικονομικό χώρο. Κάθε επιχείρηση θα πρέπει να σκέφτεται πρώτα τη διατήρηση των θέσεων εργασία. Και εδώ ίσως θα πρέπει να καταθέσω μια τροπολογία για το θέμα αυτό, να τονίσω ότι το σημαντικότερο στοιχείο με το TTIP είναι να κρατήσουμε τις θέσεις εργασίας και να εξασφαλίσουμε ότι θα εξασφαλίσουμε καταρχήν τις καλές ευρωπαϊκές θέσεις εργασίας και αυτά για τα δύο λεπτά που μου δώσατε. Thank Σας ευχαριστώ. Ε, ε, ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ την εισηγήτρια και τους συναδέρφους που παρακολουθούν την υπόθεση αυτή. Θα είμαι πολύ σύντομος. Πρώτον, το κοινοβούλιο μας πρέπει να αξιολογήσει μια τέτοια πρόταση για την οποία το κοινό έχει πολλές αμφιβολίες, πολλούς δισταγμούς, οικονομικούς, μακροοικονομικούς, γεωπολιτικούς, αναφέρθηκαν από τους συναδέρφους, αλλά υπάρχουν και εντελώς προφανείς κίνδυνοι. Σε αυτούς θα αναφερθώ. Πρώτον, για τη δημιουργική καταστροφή της ελεύθερης αγοράς που ξέρουμε ότι υπάρχει, που γνωρίζουμε ότι μια τέτοια συμφωνία ελεύθερου εμπορίου θα ωφελήσει κάποιους τομείς και κάποιους άλλους όχι, γιατί ξέρουμε η παγκοσμιοποίηση πώς λειτουργεί. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, ώστε να ξέρουμε ποιοι κλάδοι θα πληγούν Καλά κάνουμε και μιλάμε για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Παγκοσμιοποίηση. Δεύτερον, είμαστε στην Επιτροπή Απασχόληση. Εννοείται ότι οι συλλογικέ συμβάσει είναι κάτι που πρέπει να προσέξουμε όλου ιδιαίτερω και τι εργασιακέ συνθήκε που διαφέρουν στην Ευρώπη και στι Ηνωμένε Πολιτείε. Είμαστε εντελώς διαφορετικά οργανωμένοι. Συνεπώς, πριν προχωρήσουμε στη συμφωνία, να ξέρουμε ότι δεν θα πάνε προς τα κάτω τα δικαιώματα αυτά. Έπειτα για τις δημόσιες υπηρεσίες αναφέρθηκε. Προφανώς και πρέπει να προστατεύσουμε τα δημόσια αγαθά. Τουλάχιστον μέχρι πρόσφατα στην Ευρώπη τα προσέχαμε πολύ αυτά. Επίσης, προστασία δεδομένων, δικαιώματα των καταναλωτών, αρχή προφύλαξης. Είναι πολύ διαφορετική η κατάσταση στην Ευρώπη από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Και τέλος, ο μηχανισμός επίλυσης διαφορών. Είναι πολύ απλό. Δεν μπορούμε να έχουμε ένα μηχανισμό ο οποίος να καλύπτει τους επενδυτές πάνω από τον νόμο. Έχουμε συστήματα εγγύσεων και στις Ηνωμένε Πολιτείες και στην Ευρώπη. Οπότε η ομάδα μας τουλάχιστον έχει αποφανθεί κατά ενό τέτοιου μηχανισμού ISDS που θεωρούμε ότι είναι περιττός. Σίγουρα υπάρχουν αβεβαιότητες. Η ερώτηση όμως είναι η κοινή γνώμη αν είναι παραπληροφορημένη ή δεν έχει όλες τις πληροφορίες στα χέρια της, ποιος φταίει. Εκείνη ή αυτοί που κάνουν τις διαπραγματεύσεις και δεν τους ενημερώνουν. Ο κύριος Το πετύχαμε. Είδα το λόγο. Ευχαριστώ πολύ. Άρα ένα λεπτό και 50 δευτερόλεπτα. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή σας. Σε αυτές τις ε, σκέψεις της κυρίας ε, Χάρκιν θα ήθελα να προσθέσω τρία βασικά. Πρώτα πρώτα όταν μιλούμε για τα μειονεκτήματα της εμπορικής συμφωνίας, θα πρέπει να σκεφτούμε από την άλλη μεριά ποια είναι τα μειονεκτήματα του προστατευτισμού, όπως αυτά που έχει αναδείξει η ίδια ιστορία. Μακρόπνο θα πρέπει να βλέπουν οι πολιτικοί και να εξασφαλίζουν ένα καλύτερο μέλλον για τον κόσμο. Όμως, ο κίνδυνος που διατρέχει το κοινωνικό μοντέλο το ευρωπαϊκό δεν είναι το άνοιγμα το εμπορικό. Είναι το να μην έχουμε αρκετά χρήματα για να τα καταφέρουμε. Δηλαδή, θα ανοίξει νέου δρόμου η εμπορική συμφωνία, αλλά δεν ξέρουμε αν θα έχουμε αρκετά χρήματα. Οπότε θα δούμε το ότι έχουμε μάθει να ελέγχουμε, έχουμε μάθει την ελληνική. οπότε σας ζητώ το εξή από αρχής πλευράς. Θα πρέπει να κάτσουμε και να ζυγίσουμε καλύτερα τα αποτελέσματα στην απασχόληση. Αυτό θα πρέπει να το προσέξει πάρα πολύ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και επίσης να λάβει υπόψη ότι η απασχόληση και η ανεργία είναι πολύ διαφορετικά σαν έννοιε εδώ από ό,τι στι είπα. Αυτό θα πρέπει να σκεφτείτε για να ξέρουμε γιατί πράγμα μιλάμε. Εδώ θα βάλω τελείω. Πρόεδρος. Ευχαριστούμε και τώρα δώσουμε το λόγο στους εκπροσώπους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η κυρία Μονίκα από τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου. Σύντομα μπορείτε να μας πείτε τις ε, παρατηρήσεις σας για το TTIP. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Πρώτα πρώτα να ευχαριστήσουμε την κυρία Χάρκιν για το σχέδιο γνωμοδότησης ε, το οποίο είναι πολύτιμο για μας όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις αλλά επίσης την ευχαριστούμε και για την εκδήλωση που χθε ε, διοργάνωσε. Θέλω να μιλήσω για τέσσερα. Την πρώτα πρώτα τα πλεονεκτήματα για την απασχόληση, δεύτερον για τις κρατικές υπηρεσίες, τρίτον για το ISDS και τέταρτον για τα εργασιακά δικαιώματα. Πρώτα πρώτα για την απασχόληση και την θέσει απασχόληση που για το εμπόριο. Έχουμε εδώ διάφορες μελέτες και υπάρχει υπο, ε, ε, υποτίμηση και υπερεκτίμηση. Αλλά ε, σήμερα έχουμε 30 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης που από το εμπόριο και η είναι ο μεγαλύτερος μας εταίρος. Επομένω, ε, περιμένουμε 5 εκατομμύρια θέσει ε, εργασίας να <clears throat> υπάρχουν ε, λόγω του εμπορίου με τη ΣΥΠΑ. Θα γίνουν και άλλες θέσει εργασίας, γιατί τώρα θα τονωθεί το εμπόριο, γιατί υπάρχουν, υπάρχει προσθέμενη αξία με τη, με τη διατλαντική εμπορία. Επίσης, η ΕΠΑ είναι βασικός επενδυτής ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μην ξεχνούμε ότι αφορά και τις επενδύσεις αυτή η συμφωνία. Και περισσότερε επενδύσει σημαίνει περισσότερε θέσει απασχόληση. Τώρα θα γίνει αύξηση των εισαγών και εκεί θα έχουμε ε, φτηνότερε εισαγωγέ, φτηνότερη ενέργεια, φτηνά ε, ανταλλακτικά, φτηνέ πρώτε ύλε. Άρα και εκεί θα έχουμε θέσει απασχόληση. Για τι ΜΜΕ τώρα το 80% που εξάγουν σήμερα είναι ε, τέτοιες εταιρείες, 600 και 6 εκατομμύρια εργαζόμενοι. Οπότε έχουμε τώρα ε, τα δύο τρίτα ε, των εξαγωγών από αυτέ τι απασχολήσει. Όπω είπε όμω και κάποιο ομιλητή οι φραγμοί στο εμπόριο ε, σημαίνουν άλλο πράγμα για τι μεγάλε εταιρείε από για τι μικρές. Οι μεγάλες μπορούν να πάνε να επενδύσουν σε κάποια χώρα, <clears throat> αλλά ανεξάρτητα από, τις, από τους φραγμούς. Ε, όμως η ΜΜΕ δεν έχει τέτοιες δυνατότητες. Πιο πολύ θέλει εξαγωγές και άρα αυτές θα ε, ωφεληθούν από τη συμφωνία. Και είναι αλήθεια ότι δεν έχουμε τόσο μεγάλους δασμούς, αλλά έχουμε τόσο πολύ εμπορίο και ακόμα και το 1 το 2% ε, για ας πούμε για τα μαχαιροπύρωνα, για τα για τις σοκολατίτσες ας πούμε, ε, και, και μετράνε αυτοί οι μικροί δασμοί. Βεβαίως θα πρέπει να γίνουν και προσαρμογές όπως με κάθε συμφωνία, αλλά τι γίνεται τώρα με το TTIP. Έχουμε τις εξαγωγές εταιρείε που είναι ενταγωνιστικές, οπότε θα απορροφηθεί η πίεση από το άνοιγμα της αγοράς. Και έχουμε βέβαια και τους συνήθεις μηχανισμούς των κρατών μελών για την προσαρμογή. Για να δούμε τώρα τι γίνεται με τις κρατικές δημόσιες υπηρεσίες. Θέλω και εδώ να σας διαβεβαιώσω ότι όπως και στη ΣΥΤΑ, όπως και σε όλες τις συμφωνίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πρόκειται να διαπραγματευτεί με τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να περιφρουρήσει τη δυνατότητα των κρατών μελών αλλά και τη Ένωση να αποφασίζουν για το πώς θα οργανώσουν αυτές τις κρατικέ υπηρεσίες. Ε, υπάρχουν κάποιε οριζόντιες επιφυλάξει και σε την περίπτωση όπως και πάντα. Οπότε και θα, ότι θα πρέπει το κράτος να αποφασίζει αν θα κάνει υπεργολαβίες, ε, αν θα ιδιωτικοποιήσει κλπ. Το θέμα είναι να συνεχίζει να υπάρχει αυτή η ελευθερία, να διαμορφώνονται οι πολιτικέ, να μπορεί να κάνει το outsourcing, αυτές τις εξωτερικές αναθέσεις τις υπερεκολαβίες και θα πρέπει να δούμε πώς θα προσαρμόσουμε αυτές τις επιφυλάξεις και να δούμε τι θέλουν τελικά τα κράτη-μέλη πέραν των ε, κινδύνων. Είναι τεχνικό το θέμα και είναι αλήθεια ότι θα πρέπει κανείς να επαγρυπνεί όταν ε, τέτοιες διατάξεις παίρνουν από διαπραγμάτευση. αλλά υπήρχαν ρήτρες διαφύλαξης ε, σε κάθε συμφωνία, πέραν το αν υπήρχε κάποιο είδους ε, θετική ε, απαρίθμηση ή αρνητική. Τώρα, να δούμε για τους εμπειρογνώμονες. Άμα θέλει μια, μια κυβέρνηση να ξαναγίνει κρατική μη υπηρεσία που είχε ανατεθεί σε ιδιώτη. Μπορεί αυτό να γίνει. Τι θα γίνει με το ISDS ως πώς αυτό. Το ISDS δεν θα έχει να κάνει με αυτό γιατί εφαρμόζεται σε πολύ περιορισμένο αριθμό περιπτώσεων που έχουμε κάποιο είδους δυσμενή διάκριση ή κάποιο είδους ε, ε, βλάβες σε κάποια εμπράγματα δικαιώματα. Άρα, μόνο όταν φύγεται η περιουσία ενός ε, ξένου επενδυτή θα έχουμε το ISDS. Τώρα, ε, έχουμε το δικαίωμα της νομοθεσίας, ε, έχουμε άλλες βασικές αρχές ε, για την ανάπτυξη, διάφορα οριζόντια θέματα τα οποία αναφέρει η κυρία Χάρκιν. Αυτά όλα να ισχύσουν, λέει, και αυτά είναι πολύ σημαντικά. Οπότε, θα πρέπει και αυτό να το δούμε σε σχέση με την με το, το αν θα περιληφθεί εδώ πέρα η επίλυση των διαφορών για τέτοια ζητήματα. Τώρα, για να σας πω για κάτι που με απασχολεί ιδιαίτερα όσον αφορά δηλαδή, τα εργασιακά δικαιώματα. Σε κάθε ε, εμπορική ε, εταιρεία έχουμε διατάξεις ώστε να μην κατέβει ο, ο πύχης και έχουμε και μια τέτοια ρήτρα διαφύλαξης εδώ, όπως θέλετε και εσείς. Πάντως εγώ θα σα έλεγα ότι μια τέτοια εμπορική συμφωνία δεν είναι δυνατόν να περιστεί μόνο στο κοινωνικό ντάμπινγκ γιατί εδώ έχουμε μια πραγματική ευκαιρία να αλλάξουμε τον κόσμο, να τον αλλάξουμε λιγουλάκι. Γιατί μιλάμε για σημαντική δημοκρατία, μιλάμε για μεγάλο εταίρο εμπορικό, ακόμη και έχουμε τις διαφορές μας. Οπότε ε, έχουμε τις δεσμεύσεις με τον ILO και αυτό θα διαμορφώσει και το εμπόριο και τα εργασιακά δικαιώματα παγκοσμίω ένας από τους τομείς που συζητούμε είναι το αν θα υπάρχουν ε, διατάξεις για την ασφάλεια. Δεν είχαμε παλαιότερα τέτοιες συμφωνίες. Να συμφωνήσουμε σε ένα τέτοιο φιλόδοξο άρθρο για την ασφάλεια στον χώρο της εργασίας. Ε, βεβαίως. Και εδώ πέρα η αρχή της διαφύλαξης είναι κάτι σημαντικό. Τώρα, για ο ILO. έχει, έχει μια μελέτη και συνεργαζόμαστε πάρα πολύ με τον ΑΕΛΟ πάνω σε αυτό και είπαμε ότι υπάρχουν κάποιες διατάξεις στη συμφωνία μας που είναι άμεσα εκτελεστές και γι' αυτό και ε, θα είναι αυτές οι διατάξεις, οι μηχανισμοί δηλαδή την επίλυση του διαφορών θα είναι το τελευταίο το οποίο θα συζητήσουμε στις διαπραγματεύσεις. Και τώρα, εν κατακλείδη να σας πω κάτι για τις σε στάσεις όσον αφορά την εμπλοκή της κοινωνίας των πολιτών. Είναι πολύ σημαντικό. Και είπαμε να υπάρξει διαρθρωμένος διάλογος με τους Αμερικανούς για την κοινωνία των πολιτών και έτσι να προχωρήσουμε για την εφαρμοστική συμφωνία και να έχουμε εδώ πέρα προσώπους της κοινωνίας και βέβαια συνδικαλιστές. Ε, Ευχαριστούμε. Ο κύριος Ρούντι Ντελαρίου από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Θέλετε να προσθέσετε κάτι? Όχι? Ε, εντάξει. Ευχαριστούμε. Τη Γενική Διεύθυνση Εμπορίου πάντως. Κύριε Χάρκιν, σε δύο λεπτά σίγουρα μπορείτε να ολοκληρώσετε αυτό το θέμα. Εντάξει, τι να κάνω στα δύο λεπτά. Πρώτα απ' όλα, ευχαριστώ πολύ όλους τους συναδέρφους για τα σχόλιά τους. Τους άκουσα προσεκτικά. Βλέπω ότι υπάρχει μια θετική διάθεση για τις δυνατότητες που έχουμε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για αυτά που μας είπε και που ήταν και ιδίω στη χθεσινή διάσκεψη. Πολύ βοήθησε αυτό, τουλάχιστον εγώ το βρήκα πολύ χρήσιμο. Ένα σχόλιο. Ακούω ότι στις διαπραγματεύσεις πρέπει να κρατήσουμε τη σκληρή θέση και ότι πρέπει να δούμε πιο πολύ την κοινωνική ευθύνη. Ναι, άκουσα όμως και τον κύριο Πυρίνσκι, ο οποίος είπε ότι πρέπει να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε με τις επενδύσεις και την απασχόληση και όχι να σκεφτόμαστε ότι θα αλλάξουμε με τη συμφωνία αυτή τον κόσμο. Ε, εγώ νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε λίγο και από τα δύο. Ευχαριστώ. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ προθεσμία τροπολογιών 6 Μαρτίου, αύριο δηλαδή το μεσημέρι, και η συζήτηση των τροπολογιών 24 Μαρτίου και η έγκριξη την 1η Απριλίου. Θέλω να προσθέσω ότι οι τροπολογίες θα πρέπει να περιλαμβάνονται μέσα στις ε, αρμοδιότητες της Επιτροπής Απασχόλησης. Αν έχετε γενικότερες τροπολογίες θα πρέπει να τις καταθέσετε στην Επιτροπή ΙΝΤΑ και η προθεσμία για αυτό είναι 26 Μαρτίου. Σας ευχαριστώ λοιπόν για την τόσο ενδιαφέρουσα συζήτηση και πάμε τώρα στο σημείο 7 της ημέρας διάταξης επένδυση για την απασχόληση και την ανάπτυξη προώθηση οικονομικής, κοινωνικής και εδαφικής συνοχής στην Ευρώπη και δίνω το λόγο στην κυρία Γιάσλοβιέσκα. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι, η γνωμοδότηση αυτή προέρχεται από την Επιτροπή μας και είναι η συνεισφορά μας για τη συζήτηση που έχει να κάνει με το, την έκτη έκθεση του Ταμείου Συνοχής της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Κομισιόν έχει αξιολογήσει την αποτελεσματικότητα και αποδοτικότητα της πολιτικής συνοχής στο διάστημα 2007-2012. Δυστυχώς η οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση έχει μειώσει την απόδοση της πολιτικής συνοχής. Σε πολλές περιοχές χάρη στα διορθωτικά ταμεία διατηρήθηκαν οι επενδύσεις και οι θέσεις απασχόλησης, αλλά συνολικά υπήρξε σημαντική αύξηση της ανεργίας, ιδίως της ανεργίας των νέων. Υπήρξε επίσης αύξηση στην ένδια σε πολλές περιφέρειες της Ευρώπης και άνοδος του κοινωνικού αποκλεισμού. Επίσης, μετά το 2007 οι επενδύσεις έχουν μειωθεί κατά 15%. Χωρίς λοιπόν τη δράση των διαφορετικών πόρων, αυτή η μείωση θα ήταν ακόμα μεγαλύτερη. Θα μπορούσε να φτάσει και το 50% ακόμα. Η πολιτική συνοχή λοιπόν παραμένει μια σημαντική πολιτική επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία μπορεί να καταπραίνει τα αρνητικά στοιχεία της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης. Για να το κάνει αυτό όμως θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε επωφελώς αυτή την πολιτική. Λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν και περιορισμοί στο μέγεθος, στο μήκος της γνωμοδότησης. Εγώ τόνισα τα θέματα των επενδύσεων, της απασχόλησης, τη λειτουργία του Κοινωνικού Ταμείου και την απορροφησή της και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ας ανα αναλάβω αυτά τα στοιχεία. Πρώτα η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Χάρη στο Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης το 2007 με 2012 δημιουργήθηκαν 6.000 νέες θέσεις εργασία. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο έδωσε απασχόληση στο ίδιο χρονικό διάστημα σε 5,7 εκατομμύρια άνεργους. Δυστυχώς παραμένουν άλλα 24 εκατομμύρια ανέρχων στην Ευρωπαϊκή Ένωση και πολλοί από αυτούς είναι πια μακροχρόνια άνεργοι. Το Ταμείο Συνοχής λοιπόν θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πιο κατεπήγον πρόβλημα που είναι η έλλειψη οικονομικής μεγέθυνσης και απασχόλησης. <clears throat> θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι το Ταμείο αυτό χρησιμοποιείται για να διατηρήσει τις θέσεις εργασίας που υπάρχουν ήδη και να δημιουργήσει νέες θέσεις εργασίας. Δεύτερον, το θέμα της ανεργίας των νέων. Η ανεργία των νέων εξακολουθεί να είναι ένα σοβαρό πρόβλημα πέραν αυτών που έχουν γίνει η ανεργία των νέων πολλές φορές οδηγεί σε μόνιμη ένδια και κοινωνικό αποκλεισμό. Η πρωτοβουλία για την απασχόληση των νέων δεν έχει τύχει πλήρους εκμετάλλευσης από τα κράτη-μέλη. Ελπίζω ότι το 1 δισεκατομμύριο ευρώ που έχει ε, προσθεωριστεί για αυτό το στόχο θα βελτιώσει και εκεί την κατάσταση. Τρίτον, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και η απορρόφησή του. παρά το υψηλό επίπεδο ανεργίας εξακολουθούν να υπάρχουν ακόμα 2 εκατομμύρια κενέ θέσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση γιατί δεν έχουμε τα άτομα με τα απαραίτητα προσόντα και τι δεξιότητε που χρειάζονται. Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο θα πρέπει να προωθήσει περισσότερη κατάρτιση και παιδεία και επανακατάρτιση σε ορισμένου τομεί έχει ένα κεφαλαιόδη ρόλο. Θα πρέπει να δούμε όμως πώς θα χρησιμοποιήσουμε καλύτερα τα, τα, τα κονδύλια του Ταμείου και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Αυτό είναι μια νέα πρωτοβουλία μετά από μια δεκαετία σχεδόν λιτότητος και παγιοποίησης και σταθεροποίησης των δημοσιονομικών θα πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα τις επενδύσεις και την υποστήριξη των επενδύσεων. Εμείς θα πρέπει να υποστηρίξουμε στο εγχείρημα αυτό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την πρόταση για το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, διότι μαζί με τα διαφορετικά ταμεία αυτό μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό εργαλείο επενδύσεων για την Ευρωπαϊκή Ένωση που θα μπορούσε δυνητικά να δημιουργήσει 1,3 εκατομμύρια νέε θέσει εργασία και αυτά και προσβλέπω στα σχόλια των συναδέλφων. Ευχαριστώ, θα δώσω τώρα το λόγο στους σκιώδεις. Καταρχήν την Εύα Καϊλή που είναι αναπληρωματικό μέλος. Uh, Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ την εισηγήτρια για την εξαιρετική της δουλειά στο σχέδιο αυτό γνωμοδότησης. Πρέπει να πω επίσης ότι είμαστε πολύ ικανοποιημένοι που αναφέρεται το θέμα της ανεπάρκειας των κονδυλίων για την απασχόληση. Η θέση της ομάδας μας, όπως γνωρίζετε, είναι ότι πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο προς αυτή την κατεύθυνση, ιδιαίτερα για την απασχόληση ποιότητας. Τονίζουμε το ποιότητα για νέους κυρίως. Συνεπώς δεν μιλάμε γενικά για την δημιουργία απασχόλησης, μιλάμε για απασχόληση που θα καλύψει τις ανάγκες του εργατικού δυναμικού και βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα. Εκπροσωπούμε τους πολίτες μιας χώρας που έχει τα μεγαλύτερα ποσοστά ανεργίας των νέων. Στην Ελλάδα σχεδόν 50% των νέων είναι άνεργοι. Είμαστε ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένοι σε αυτό το ζήτημα και χαίρομαι που συμπεριλαμβάνεται στη δεύτερη παράγραφο του σχεδίου γνωμοδότησης. Όμως θέλουμε να προσθέσουμε και κάποια άλλα σημεία που πιστεύουμε ότι είναι αναγκαία και θα μπορούσαμε να τα συμφωνήσουμε όλοι. Όταν λέμε αντιμετώπιση της ανεργίας πρέπει να λάβουμε υπόψη μας τη διάσταση του φύλου. Όλε οι στατιστικέ δείχνουν ότι οι γυναίκε αγωνίζονται πολύ περισσότερο να έχουν μια μόνιμη θέση απασχόληση και η θέση του στην αγορά εργασία είναι πιο επισφαλή από την εκείνη των ανδρών. Επίση, πλήττονται περισσότερο από την οικονομική κρίση. Υπάρχει και διαφορά στις αμοιβέ που εξακολουθεί να υπάρχει σε πολλέ ευρωπαϊκέ χώρε. Το ίδιο ισχύει και για διάφορες μειονότητες σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες που έχουν λιγότερες ευκαιρίες στην εκπαίδευση, την κατάρτιση και την απασχόληση. Ένα άλλο θέμα είναι ότι πρέπει να έχουμε προδιαγραφές ποιότητας στην ε, κατάρτιση που προσφέρουμε. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούμε σαν άλλο την κρίση και να μην κάνουμε τίποτα γι' αυτό. Επειδή όταν μιλάμε για τις χώρες της Νότιας Ευρώπης, η αγορά εργασίας εκεί έχει πληγεί όλος ιδιαίτερος. Ένας ελάχιστος μισός σε αυτές τις χώρες θα μπορούσε να είναι ένα ζωτική σημασία μέτρο. Πρέπει επίσης να ερευνήσουμε και τις επιπτώσεις των μέτρων λιτότητας σε διάφορες ευρωπαϊκές αγορές απασχόλησης και τι δυνατότητες δημοσιονομικές υπάρχουν για να αμβληθεί και το φαινόμενο της κυκλικής ανεργίας. Αυτό δηλαδή που χρειαζόμαστε είναι προοπτικές ανάπτυξης για όλους. Εννοούμε ανάπτυξη που να μειώνει την ανεργία, μια που η ανάπτυξη και η απασχόληση δεν έχουν γραμμική σχέση απαραίτητα. Τα όσα προτείνει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικικών Επενδύσεων είναι βέβαια σημαντικά για να πετύχουμε αυτό το στόχο. Το ρόλο του λοιπόν πρέπει να τον τονίσουμε. Επενδύσεις, ναι, που να δημιουργούν απασχόληση όμως, όχι επενδύσεις χωρίς απασχόληση και μακρόχρονα μάλιστα, μακροπρόθεσμα. Γιατί όταν δεν υπάρχει πια αυτό το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στατικών Επενδύσεων, πρέπει η κατάσταση να είναι τέτοια που να συνεχίζουν να δημιουργούνται θέσεις απασχόλησης. Θέλουμε και τον ρόλο των νέων τεχνολογιών και των τεχνολογιών πληροφορικής για τη δημιουργία περισσότερων θέσεων απασχόλησης, κυρίως της νέας γενιάς και γυναικών. Γιατί και εδώ παίζει το θέμα της ισότητας των φύλων. Οι νέες τεχνολογίες μπορούν να βοηθήσουν με δημιουργία τέτοιων θέσεων απασχόλησης που να είναι πιο ευέλικτες όσον αφορά το ωράριο. Η τεχνολογία λοιπόν είναι ένα εργαλείο που πρέπει να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά προς αυτή την κατεύθυνση. Γιατί μείωση της ανεργίας με την ψηφιακή τεχνολογία και τον Horizon 2020. Τέλος, η αρμόδια επί της ουσίας είναι η Επιτροπή Περιφερειακών Υποθέσεων. Η σύγκληση στην Ευρώπη λοιπόν είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο. Ένα από τα αποτελέσματα της κρίσης δυστυχώς ήταν η διάλυση των περιφερειακών δομών. Συνεπώς, τροπολογίες μας θα έχουν να κάνουν με αυτές που σας ανέφερα. Ευχαριστώ και πάλι για το σχέδιο γνωμοδότησης. Thank you. And now give the... Εμείς ευχαριστούμε. Να δώσουμε το λόγο σε άλλο ένα νέο αναπληρωτή, τον Αμάλ Μπασίρα από το ECR. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Σας ευχαριστούμε ε, και για το καλωσόρισμά σας την τελευταία φορά. Και εγώ προσδοκώ να συνεργαστώ πάρα πολύ καλά με τους αδέλφους. Να ευχαριστήσω την εισηγήτρια. Πάρα πολύ σωστά τα όσα λέει και εστιάζει την προσοχή της στη δημιουργία θέσεων απασχόληση. Για να ρωτήσετε κάποιον ο οποίο είχε μικρομεσαία επιχείρηση όπω εγώ, ε, στο μέτρο μέρος ζωής μου, από πρώτο χέρι γνωρίζω το πόσο σημαντικέ είναι οι ΜΜΕ σε δημιουργία θέσεων απασχόληση και πόσο σημαντικέ για την ανάπτυξη. Νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι ο ρόλος των ΜΜΕ αποτυπώνεται στο κείμενο. Έχω υποβάλει σχετικές τροπολογίες. Επίσης, συμφωνώ ότι δυστυχώς οι ενωσιακοί πόροι δεν χρησιμοποιούνται όσο αποτελεσματικά θα έπρεπε και άρα θα πρέπει να εστιάσουμε προσοχή μας στην αποτελεσματικότητα αλλά και στην πιο εύστοχη νομοθεσία ούτως ώστε να εξασφαλιστεί ότι θα πηγαίνουμε προς μια χάραξη πολιτικής που φέρνει αποτελέσματα. Συνάδελφοι, ως μέλος της ECR, ε ε, για μένα είναι ξεκάθαρο ότι η πολιτική της συνοχής δεν θα πρέπει να οδηγεί σε επιδότηση μη βιώσιμων επιχειρήσεων. Πάντως, <clears throat> αν θέλουμε να δημιουργηθούν θέσεις απασχόλησης και ανάπτυξη θα πρέπει να προσέξουμε το πώς θα δημιουργήσουμε το κατάλληλο επιχειρηματικό περιβάλλον, ούτω ώστε να ε, ε, εκμεταλλευτούμε τις δυνατότητες των βιώσιμων ΜΜΕ, γιατί αυτές είναι η της οικονομίας. Και σας ευχαριστώ. Πρόεδρος. Σας ευχαριστώ. η κυρία Τάνια Γκονσάλες Πένιας από την ΚΟΕ. Ευχαριστώ πολύ την ε, εισηγήτρια για το έργο της. Σύμφωνα σε πολλές πτυχές ότι παραδείγματος χάρη ήταν μεγάλη η επίπτωση σε αρνητικό επίπεδο της μείωσης των δημοσίων επενδύσεων για την ανάπτυξη και την απασχόληση. Σύμφωνα ότι τα Ταμείο Συνοχής είναι πολύ σημαντικό για τις επενδύσεις και επομένως θα πρέπει να ξανασκεφτούμε λιγάκι την στρατηγική Ευρώπη 2020 γιατί όπως πηγαίνουμε δεν θα επιτύχουμε τους στόχους της 75% απασχολησιμότητας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα πρέπει λοιπόν να συγκεντρώσουμε τις προσπάθειες μας για να γίνει, γενικό, για να γίνει, στο, πραγματικότητα αυτός ο στόχος. Γενικά τα κονδύλια που έχουν να κάνουν με την απασχόληση και ιδίως για τις χώρες του Νότου όπου είναι πάρα πολύ ψηλό το επίπεδο ανεργία, είναι απαράδεκτο υψηλό όπως συμβαίνει στη δική μου χώρα, που η ανεργία των νέων έχει ξεπεράσει και το 50% είναι απαραίτητο να εστιάσουν εκεί οι προσπάθειε, αλλά συγχρόνως θα πρέπει να σκεφτούμε ότι δεν αρκεί να δίνουμε κονδύλια και μόνο. Δεν πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μονάχα τα χρήματα, αλλά πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε σωστά για να δημιουργήσουμε θέσει απασχόληση και μάλιστα θέσει απασχόληση που να έχουν κάποια ποινότητα ποιότητα. Λέει οι εισηγήτρια πρέπει να χρησιμοποιηθούν πιο γρήγορα τα διαθέσιμα κονδύλια για την απασχόληση των νέων. Αυτό είναι ένα παράδειγμα έλλειψης <coughs> προγράμματος. Ξεκινά αυτό το πρόγραμμα με μια λανθασμένη αντιμετώπιση για την ανεργία των νέων. Θεωρεί ότι το πρόβλημα είναι η απασχολησιμότητα των νέων, το πόσο δύσκολο είναι οι νέοι να έχουν μία απασχόληση, θεωρεί ότι δεν έχουν αρκετά, ε, αρκετά μεγάλη ευελιξία, δεν έχουν την απαραίτητη ικανότητα να βρούνε μια θέση εργασίας. Αλλά στην Ισπανία έχουμε προγράμματα ε, επιχειρήσεων όπως η McDonald's που ωφελούνται από αυτό το πρόγραμμα. Η απασχόληση στη McDonald's είναι ακριβώς ένα παράδειγμα που δεν δίνει εργασία ποιότητος, αλλά κάνει ακριβώ το αντίθετο. Είναι μια φάμπρικα η οποία φτιάνει επισφαλείς θέσεις εργασίας. Θα πρέπει λοιπόν να εστιάσουμε στην ε, πραγματική απασχόληση ποιότητος και όχι στην επισφαλή και περιστασιακή εργασία. Όταν το Παρτίδο Ποπουλά στη χώρα μου λέει ότι δημιουργεί θέσει απασχόληση, η πραγματικότητα είναι ότι όλε αυτέ τι θέσει απασχόληση που δημιουργήθηκαν στο 2014 είναι κατά 90% Επισφαλή θέση εργασία. Αυτό είναι λοιπόν μια δυναμική η οποία όχι μόνο χάσει στην Ισπανία αλλά και σε όλη την Ευρώπη ε, αντικαθιστά τη μόνιμη απασχόληση, την αξιοπρεπή απασχόληση με επισφαλή και προσωρινή εργασία. Και αυτό υποβαθμίζει τις συνθήκες εργασίας και εδώ θα πρέπει εμείς να σκεφτούμε περισσότερο για το πώς θα χρησιμοποιήσουμε αυτά τα κονδύλια με έναν τρόπο ο οποίος θα δημιουργήσει πραγματικές θέσεις εργασίας και δεν θα οδηγήσει μονάχα σε επισφαλείς εργασίες. Πρέπει να βιομηχανοποιήσουμε και πάλι την Ευρώπη, πρέπει να έχουμε διατήρηση των επιχειρήσεων στην Ευρώπη και να πρέπει να δώσουμε οικονομικές ευκαιρίες. Η Τζιν Λάμπερτ. Ευχαριστώ. Ε, για λόγω της Μόνικα να σας μιλήσω που είναι ισχυώδης εισηγήτρια. Θα ήθελα να ευχαριστήσει η Μόνικα την εισηγήτρια για το έργο της και επίσης ε, να πούμε ότι πρόκειται για αξιόλογη έκθεση και θα είναι αφετηρία για περαιτέρω προβληματισμό και δείχνει πόσο σημαντική είναι η πολιτική της συνοχής, ιδίως τις ώρες της ε, κρίσης ακριβώς, όπως και κατέληξε και έκθεση για την συνοχή. Αλλά θα πρέπει να ενδυναμωθεί γενικά η πολιτική τη συνοχή, ιδίως για κοινωνικές υποθέσεις και βεβαίω ο σκοπός δεν είναι μόνο να αντιμετωπίσουμε την ανεργία, αλλά επίσης να αντιμετωπίσουμε και τον κοινωνικό αποκλεισμό. Αυτό θα πρέπει να το τονίσουμε. Επίσης, και να ενσωματώσουμε εδώ τους στόχους της Ένωσης για το 2020. Όχι μόνο για την απασχόληση, όλους τους στόχους. Όπως είπαμε για την ισότητα των ε, φύλων, για το κλίμα, για τη φτώχεια. Τώρα μια επίκριση γενικού χαρακτήρα όσον αφορά το χρηματοδοτικό μέσο, ότι δεν υπάρχει εδώ πέρα κάποια δέσμευση υποχρεωτική σε σχέση με τον στόχο της ε, δαφικής ε, συνοχής. πρέπει να γίνει εδώ αυτή η σύνθεση, γιατί έχουμε τη μελέτη του ILO που λέει ότι όταν έχουμε επενδύσει σε περιφέρειες με την περισσότερη ε, ε, ανεργία, ε, τότε θα πρέπει να έχουμε κάποια αυθεντικά μέτρα για την αγορά εργασίας, όχι μόνο κυρώσεις. Και τότε οφείλεται η απασχόληση από ε, την πολιτική αυτή. Τώρα, εκεί που λέμε για δημιουργία θέσεων απασχόληση να τονίσουμε την σημασία των ΜΜΕ και σε σχέση με τους στόχους του 2020. Αυτά για μας είναι πολύ σημαντικά. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε, λέει Πρόεδρος. Σοφία Ριμπέιρο. Ευχαριστώ πολύ. Και εγώ θέλω να συγχαρώ την εισηγήτρια για το έργο που έχει φέρει σε πέρα. Είναι απαραίτητο να λάβουμε υπόψη την ανάγκη της αξιοπρεπούς εργασίας και του, της αντιμετώπισης του κοινωνικού αποκλεισμού. Αυτό αφορά περισσότερο τις πιο φτωχές περιοχές οι οποίες έχουν μεγάλες δυνατότητες ανάπτυξης. για μένα είναι απαραίτητο να έχουμε μια βιώσιμη ανάπτυξη και αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρξει μια τροποποίηση του παραδείγματος των ταμείων συνοχής. Δεν θα πρέπει να υπάρξει μια κεντρική αντιμετώπιση για όλα αυτά τα θέματα. Θα πρέπει όμως να συμπεριλάβουμε και κοινωνικούς ε, στόχους στην εφαρμογή των ταμείων αυτών και να μπορέσουμε να επιτύχουμε <clears throat> βιώσιμες κοινωνικές συνδίκες. Πρέπει λοιπόν να έχουμε μια σωστή επιλογή των επιλεξίμων σχεδίων για τα θέματα αυτά. Θα πρέπει λοιπόν να υπάρξει ένα μοντέλο επενδυτικό το οποίο θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει και την άποψη των κοινωνικών εταίρων, των ε, τοπικών αρχών της κοινωνίας των πολιτών και γι' αυτό θα πρέπει η πρόταση της Κομισιόν να συμπεριλάβει και αυτή την πτυχή ε, θεσμοποιήσει σε ένα ευρωπαϊκό κώδικα συμπεριφοράς. Εγώ θέλω να δω πώς η Κομισιόν θέλει να εξασφαλίσει την ε, κοινωνική ενσωμάτωση. Εγώ πιστεύω ότι δεν λαμβάνει υπόψη τις συλλογικές συμβάσεις στο πρόγραμμα της Κομισιόν και επίσης δεν λαμβάνει υπόψη όλα τα θέματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση και την ε, ε, κοινωνική ε, δικαιοσύνη. Θα πρέπει λοιπόν τα 315 δισεκατομμύρια να έχουν στόχους οι οποίοι θα πραγματικά λειτουργήσουν υπέρ της μείωσης των κοινωνικών, κοινωνικών, οικονομικών και περιφερειακών ε, ανισοτήτων. Είναι απαραίτητο λοιπόν να υπάρξουν συνοδευτικά μέτρα για τα λειτουργικά προγράμματα στο Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να εμπλακεί πλήρως σε αυτή τη διαδικασία. Θα πρέπει να υπάρχουν επίσης και κανόνες σαφείς για την αξιολόγηση των προγραμμάτων που θα πρέπει να ε, έχουν αποφασιστεί τώρα και να μην φτάσουμε το 2017 όταν γίνεται η ενδιάμεση αξιολόγηση και να δούμε ότι υπάρχουν κράτη-μέλη τα οποία δεν έχουν πετύχει τους στόχους και δεν έχουν σωστή αξιολόγηση. Δεν πρέπει να παραβιαστεί η αρχή της επικορικότητας, αλλά θα πρέπει να υπάρξει μόνιμη εποπτεία της εφαρμογής αυτών των ταμείων και έλεγχος των κοινωνικών αποτελεσμάτων που προκύπτουν, αλλιώς θα δημιουργήσουμε ανισομέρειες σε κοινωνικό επίπεδο και μεγαλύτερες διαφορές μεταξύ κρατών μελών και περιοχών και ιδίως σε αυτές που έχουν μεγαλύτερη δυνατότητα να παίξουν το ρόλο τους σε κοινωνικό επίπεδο. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό λοιπόν αυτό το στοιχείο γιατί προέρχομαι από μια περιφερειακή περιοχή της Αζόρες που έχουν πολλά μειονεκτήματα λόγω της περιφερειακότητάς τους, δυσκολίες πρόσβασης στην ευρωπαϊκή αγορά λόγω του χαρακτήρα του νησιωτικού και περιφερειακού. Γι' αυτό πρέπει να δώσουμε την πρέπουσα προσοχή στους δείκτες αυτούς οι οποίοι έχουν κοινωνικό χαρακτήρα και να παρακολουθούμε μόνιμα αυτά τα οποία γίνονται στον κοινωνικό τομέα όταν εφαρμόζονται τα ταμεία αυτά. Αλλιώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα μπορέσει να έχει την συνένεση των Ευρωπαίων πολιτών. Ευχαριστούμε κύριε Στόμας Μαν. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω και την Δανούτα. Είναι η δεύτερη έκθεση που αντιμετωπίζουμε σήμερα. Το σημαντικότερο επιχείρημα είναι θέλουμε να διατηρήσουμε την κοινωνική συνοχή και να υποστηρίξουμε και την εδαφική συνοχή. Πρέπει να δούμε και τις περιοχές της περιφέρειας ότι και αυτές μπορούν να επωφεληθούν και να δώσουμε κίνητρα στους ανθρώπους να μπορέσουν να δημιουργήσουν θέσεις εργασίας σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις, να δώσουμε τους ανθρώπους να είναι πιο ανταγωνιστικοί και να έχουν νέα προϊόντα. Υπάρχουν πολλές οργανώσεις ε, ε μικρομεσαίων επιχειρήσεων που μπορούν να συμβάλλουν σε κάτι τέτοιο. Τα ταμεία συνοχής λοιπόν θα πρέπει να δράσουν, πολλές φορές αντιμετωπίζονται με επικριτικό τρόπο σε ορισμένα κράτη. Δεν μπορούν να κάνουν τα πάντα και χωρίς αυτά είναι πάρα πολλά πράγματα τα οποία δεν θα γίνουν. Τα κράτη-μέλη δεν έχουν τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα αυτά ένδυας που αναδύονται. Είναι απαραίτητο να δώσουμε τη δυνατότητα να έχουμε και δημιουργία νέων επιχειρήσεων οι οποίες αναλαμβάνουν υψηλότερους κινδύνους και εδώ υπάρχουν μέθοδοι όπως η μικροχρηματοδότηση. Θα πρέπει να εστιάσουμε, να βοηθήσουμε αυτούς οι οποίοι έχουν ένα νέο προϊόν αλλά δεν ξέρουν πώς θα μπορέσουν να βγουν στην αγορά. Αυτό λοιπόν θα πρέπει να υποστηρίξουμε γιατί έτσι δημιουργούνται θέσει εργασία. Δεν έχουμε βέβαια καμία εγγύηση της ε, ε, αηφορίας αλλά θα πρέπει να έχουμε και κάποια εστίαση σε νέες πρωτοβουλίες οι οποίες αναλαμβάνουν κάποιο κίνδυνο. Γιατί δεν έχει προχωρήσει η πρωτοβουλία για τους νέους. Σε πολλά κράτη-μέλη δεν είναι σαφές πώς θα γίνει αυτή η διαχείριση των κονδυλίων. Υπάρχουν εσωτερικές διαμάχες στην, στις δημόσιες διοικήσεις για το πώς θα γίνει αυτό με συγκεκριμένο τρόπο. Λοιπόν, θα πρέπει να κάνουμε συγκεκριμένα μέτρα για να μπορέσουμε να αντιμετωπίσουμε την αργία των νέων, γιατί αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό τομέα για τον οποίο πρέπει να εργαστούμε. Ανέφερε η συνάδελφος από την Ισπανία πόσο δύσκολη είναι η κατάσταση. Εγώ θέλω να τονίσω ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα με την ε, εφαρμογή του προγράμματος για τους νέους. Σιγά σιγά τώρα στην Ισπανία ξεκινάει το θέμα της δυτής ε, κατάρτισης. Αυτό είναι ένα καινούριο στοιχείο το οποίο θα μπορέσει να λύσει πολλά προβλήματα. Δεν πρέπει λοιπόν η εκπαίδευση να οδηγεί σε δεξιότητες οι οποίες δεν είναι χρήσιμες. Θα πρέπει να έχουμε μια νέα επανεξισορρόπηση της παιδείας και αυτό είναι κάτι το οποίο ελπίζω ότι θα μπορέσει να στεφθεί υπό επιτυχία στην Ισπανία. Δεν πρόκειται να τα καταφέρουμε όλα αυτά μέσα σε ένα εξάμεινο ή σε ένα χρόνο. Θα πρέπει όμως να προχωρήσουμε σε μακροπρόθεσμο επίπεδο και να έχουμε συγκεκριμένα προγράμματα τα οποία δεν αφορούν μονάχα την, ε, ε τη δημιουργία μελετών αλλά τη συγκεκριμένη εφαρμογή. Δεν θέλουμε λοιπόν να αποτύχουν σε αυτό το κατημέρι θέλουμε να δημιουργήσουν την απαραίτητη ευρωπαϊκή προσθέμενη αξία. Ευχαριστούμε. Η κυρία Σαντόροβα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ και την εισηγήτρια βέβαια. Θα ήθελα να ασχοληθώ με το θέμα της μέτρησης, της εκτίμησης των προγραμμάτων. Ο μόνος τρόπος με τον οποίο μπορούμε να υποστηρίξουμε τέτοιου είδους επενδύσεις είναι αν γνωρίζουμε ότι πράγματι θα λειτουργήσουν, ότι πράγματι θα δώσουν αποτελέσματα. Μιλάμε για τεράστια ποσά. Η Επιτροπή Γυναικών θα εξετάσει και αυτή το θέμα από πλευρά της ανεργίας των γυναικών και την επανένταξη των μητέρων στην αγορά εργασίας. Θα ήθελα επίσης να ρωτήσω κάτι και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μια στιγμή, διακόπτη πρόεδρος. Είσαστε πάρα πολύ κοντά στο μικρόφωνο και δεν ακούγεστε καλά. Συγγνώμη, λέει η ομιλήτρια. Έχω την εξή ερώτηση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με εκπλήσει η μεγάλη αύξηση 72% στην χρηματοδότηση μεταρρυθμίσεων δημοσίων υπηρεσιών. Είμαστε σε μια κατάσταση όπου μέχρι το 2013 αυτός ήταν ένας τομέας που επίσης είχε υποφεληθεί από υψηλή χρηματοδότηση. Η στήριξη αυτή ήταν, είχε αποφασιστεί πριν το 2013 και συνεχίστηκε και μετά με μεγαλύτερα ακόμα ποσά. Μπορεί να εξηγήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατά πόσο τα ποσά αυτά συνοδεύτηκαν και με ποιοτική αύξηση. Ωραία, τώρα το λόγο έχει η συγγήτρια. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω όλους τους ευρωβουλευτές για τις απόψεις τους και τα σχόλιά τους. Φυσικά και θα έχω υπόψη μου τα σχόλιά σας αυτά και περιμένω να δω και τις τροπολογίες σας. Τώρα για να απαντήσω στην κυρία Καϊλή. Πρέπει να πω ότι έχω κάποιες αμφιβολίες και θα εξηγήσω ποιες είναι αυτές και γιατί. Η κυρία Καϊλή μας είπε ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των χωρών μελών όσον αφορά τις αμοιβέ, τους μισθούς. Οι έρευνες όμως δείχνουν ότι στις περισσότερες περιπτώσεις η μείωση των αμοιβών στα πλαίσια της κρίσης δεν είχε ένα τέτοιο αποτέλεσμα. Δεν υπήρξαν επενδύσεις, είναι αλήθεια, και αυτό επιδίνωσε γενικά την κατάσταση. Επίσης η έρευνα δείχνει ότι οι επιχειρήσεις ή οι επιχειρηματίες δεν συμμετέχουν στην κατάρτιση λέμε ότι πρέπει να έχουμε βασική κατάρτιση για τους εργαζόμενους, για τους εργάτες, αλλά δεν φροντίζουμε από την άλλη μεριά οι επιχειρήσεις και οι επιχειρηματίες να περάσουν και αυτοί από κάποια κατάρτιση, γιατί αλλάζει ο κόσμος. Γι' αυτό και λέω ότι έχω κάποιες αμφιβολίες. Ίσως πρέπει να το συζητήσουμε περισσότερο και ίσως πρέπει να συμπεριλάβουμε κάτι τέτοιο έτσι ώστε να υπάρξει αύξηση στην παραγωγικότητα των εργαζομένων. Κάτι το οποίο θα οδηγήσει με τη σειρά του σε υψηλότερους μισθούς. Σας ευχαριστώ πάντως για τις παρατηρήσεις και τα σχολιά σας και προσβλέπω σε συνεργασία. Ευχαριστούμε κυρία Η προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών είναι η 10η Μαρτίου στις 12 το μεσημέρι. Θα εγκριθεί στην Επιτροπή μας στις 16 Απριλίου η γνωμοδότηση αυτή και η Ρέτζη θα ψηφίσει 4 με 5 Μαΐου. Ωραία. Και φτάνουμε στο τελευταίο σημείο που έχουμε για σήμερα στην ημερήσια διάταξη, που είναι οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση είναι η πρώτη ανταλλαγή απόψεων που έχουμε επί της νομοθετικής πρότασης Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εγκρίθηκε στις 2 Μαρτίου. Οι κατευθυντήριες γραμμές αναθεωρούνται για πρώτη φορά μετά το 2010 και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμμετέχει στη διαδικασία διαβούλευσης. Αρχίζουμε λοιπόν προσκαλώντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Και έχουμε τον κύριο Γιώργεν Γιούτε από την Γενική Διεύθυνση Απασχόλησης. Παρακαλώ, έχετε το λόγο πρώτα η Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Στην αρχή της εβδομάδας, πράγματι, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε ένα νέο πακέτο κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση Και αυτές τις κατευθυντικές γραμμές ήρθα να σας παρουσιάσω σήμερα. Φυσικά και έχουν άμεση σχέση με τις ευρύτερες πολιτικές μας. Αλλά έχουμε δύο νομικά μέσα, πιο συγκεκριμένα, ε, με τα οποία έχει πιο σημαντικό ρόλο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Από πού ξεκινάμε. Οι κατευθύνσεις γραμμές για την απασχόληση εγκρίθηκαν καταρχήν με τις ευρύτερες κατευθύνσεις γραμμές πολιτικής ως πακέτο το 2010. Είχαμε τη στρατηγική 2020 που αποφάσισε ότι οι ολοκληρωμένες αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα παραμείνουν μέχρι το 2014. Για να στηρίξουν τις, τα επιτεύγματα μια εφιούς ε, ανάπτυξης με τη συμμετοχή όλων που βασίζεται στον οικονομικό συντονισμό. Οι κατευθυντήριες γραμμές μιλούν για την κατεύθυνση του συντονισμού των πολιτικών των χωρών μελών και αποτελεί και τη βάση για τις ειδικέ συστάσεις των χωρών έτσι όπως καθορίζονται στην ε, διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και εγκρίνονται από το Συμβούλιο Μάιο και Ιούνιο. Τι αλλάζει. Με την έγκριση των νέων κατευθυντηρίων γραμμών από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, η Επιτροπή επομίζεται την κληρονομιά της κρίσης και την πολιτική της για βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση την ε, κάνει συγκεκριμένες προτάσεις, συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές που αντικατοπτρίζουν μια νέα προσέγγιση στην εκπόνηση οικονομικής πολιτικής, ενισχύοντας την επενδύσεις, προθώντας την ανάπτυξη με την εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων. Έχουμε συγκεκριμένους προσανατολισμούς για την ενίσχυση των επενδύσεων και για τις διαστατικές μεταρρυθμίσεις. Επίσης, καταργούμε τους φραγμούς στην ανάπτυξη και την απασχόληση σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και βελτιώνουμε την βιωσιμότητα και το φιλικό περιβάλλον για τη, τα δημοσιονομικά των χωρών μελών. Επιπλέον, στην περίπτωση των κατευθυντηρίων γραμμών για την απασχόληση, αυτό σημαίνει ότι καλύπτουν και διαφορετικές αλλαγές στον τομέα της απασχόλησης. Και αυτό το πετυχαίνουμε με τέσσερα πράγματα. Δίνουμε όθηση στη ζήτηση για απασχόληση, ενισχύουμε την αγορά εργασίας και προσόντα και δεξιοτεχνίες των εργαζομένων, όπως επίσης και την λειτουργία της αγοράς. Ας αρχίσουμε από την αρχή την ενίσχυση της ζήτησης για απασχόληση. Με τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, με τη φορολόγηση στην εργασία και με καθορισμό αποδοχών. Δεν θέλουμε να υπάρχει μεγαλύτερο βάρος, μεγαλύτερο εργασιακό κόστος. Ο δεύτερος τομέας είναι η προσφορά απασχόλησης. Εδώ συμμετέχουμε με συστάσεις και συμβουλές σε επίπεδο εκπαίδευσης και επαγγελματικής κατάρτισης και αντιμετωπίζουμε και την ανεργία των νέων, καθώς επίσης και τη μακροχρόνια ανεργία. Όσον αφορά τη συμμετοχή τώρα και τα επίπεδα δεξιοτεχνίας, είναι και αυτό ένα θέμα που περιλαμβάνουμε, καθώς επίσης και ε, να βοηθήσουμε τις διαφορετικές αδυναμίες που υπάρχουν για να πάψουν να υπάρχουν βέβαια. Επίσης, ενισχύουμε την λειτουργία των αγορών εργασίας, μειώνοντας τον κατακαιρματισμό των αγορών εργασίας, βελτιώνοντας τις πολιτικές για το ενεργό δυναμικό και την κινητικότητα των εργαζομένων. Θέλουμε ευελιξία και προστασία. Και φυσικά καλύτερα στοχευμένα μέτρα για την αγορά εργασίας και στήριξη στην κινητικότητα των εργαζομένων. Και το τελευταίο έχει να κάνει με την ε, δικαιοσύνη, με την καταπολέμηση της ένδιας και της ίσες ευκαιρίες. Εδώ η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θέλει να προχωρήσει σε εξυγχρονισμό των κοινωνικών ε, συστημάτων, κοινωνικής ασφάλισης δηλαδή είτε πρόκειται για ανέργους, είτε πρόκειται για συνταξιούχους, είτε πρόκειται για άτομα που χρήζουν περίθαλψης. Θέλουμε υπηρεσίες οι οποίες να διευκολύνουν τη συμμετοχή όλων στην αγορά εργασίας. Με την πρόταση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής συζητάμε τις κατευθυντήριες γραμμές πια. Κατά το παρελθόν, οι ανταλλαγές που είχαμε, ιδιαίτερα με τους ευρωβουλευτές, ήταν πολύ καρποφόρες και ο Γενικό μου Διευθυντής, γενικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσβλέπουν σε αυτό το διάλογο με στόχο να κατελήξουμε σε κατευθυντήριες γραμμές για όλες τις χώρες μέλη και να διασφαλίσουμε και την πρόοδο. Ελπίζουμε, ελπίζουμε να έχουμε τις συστάσεις αυτές τον Ιούνιο, να εγκριθούν δηλαδή τον Ιούνιο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας και εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προσβλέπω στα αρχικά σας σχόλια. Ευχαριστώ. Θα δώσω τώρα το λόγο στην Λάουρα Αγγί, την εισηγήτρια. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την ε, εισήγησή της. Θα εστιάσουμε την προσοχή μας για αυτά τα τέσσερα στοιχεία, τέσσερα τέσσερις άξονες όπου μας τα εξήγησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να πω και τις παρατηρήσεις μου. Ε, μιλούμε τώρα για κάποια φορολογική πίεση και ότι θέλουμε να μετακυλιστεί από την εργασία ε, σε άλλου είδους φορολογικές επιβαρύνσεις. Θέλουμε ομογενοποίηση ε, της φορολογίας, διότι μιλούμε για κάποια φαινόμενα τα οποία τώρα έχουν καθορίσει την κρίση. Και αυτό γίνεται γιατί δεν υπάρχει ακριβώς αυτή η ομοιογένεια στην ευρωπαϊκή φορολογία. Οπότε θα πρέπει να δούμε ότι θα αποφύγουμε να κάνουμε τέτοια μέτρα, ας πούμε, την, με την κατάσταση και επίσης θα καταπολεμήσουμε και την ανεργία. Για να δούμε τώρα τις ε, διαρθωτικές μεταρρυθμίσεις. Και επίσης την ε, δημιουργική λογοδοσία. Αυτά τα οποία ζητούνται από τα κράτη-μέλη είναι ακριβώς αυτό το να υπάρχει περισσότερη δημοσιονομική πειθαρχία. Πρόκειται για κάποια μέτρα τα οποία επιβάλλονται και πρόκειται για κάποιες διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις ε, που κατατείνουν στην λιτότητα χωρίς να βοηθούν στην απασχόληση. Δεν θα πρέπει να ξεχνούμε ότι η κρίση που πάρα πολλοί επιμένουν να θεωρούν ότι είναι κάτι το οποίο αφορά τον νότο της Ευρώπης και μόνο τον νότο δημιουργεί τα ασύμετρα σοκ και αργά ή γρήγορα αυτό θα είναι ένα κύμα που θα πλήξει όλες τις χώρες της Ένωσης γιατί τώρα έχουμε τα προβλήματα της απασχόλησης σε κάποιες χώρες αλλά θα πρέπει να θυμόμαστε ότι η απόλυτη φτώχεια έχει χτυπήσει πολύ περισσότερες χώρες και αυτά τα σύμμετρα σοκ χτυπάνε περισσότερες χώρες εκεί όπου μπορούμε να έχουμε κάποια αντιμετώπιση αποτελεσματική και να υπάρχει έλεγχο σε και για το χρέος. Όλα αυτό θα έπρεπε να τύχει βοήθειας για να μπορέσουμε να λύσουμε το ζήτημα της απασχόλησης. Γιατί λέμε εδώ πέρα για πρόληψη της ανεργίας, μα έχουμε σαφείς ενδείξεις και θα πρέπει να οργαστούμε σε αυτό το μέτωπο για να αντιμετωπίσουμε την ανεργία. Να μην μιλάμε για απασχόληση αν πρώτα δεν λύσουμε το πρόβλημα της ανεργίας. Επίσης βλέπω με ικανοποίησή μου ότι μιλούμε για τους ε, ανέργους, για τους ανέργους, τους ανέργους νέους ε, γιατί μιλούμε για τους ε, μακροπρόθεσμα άνεργους. Είναι εκείνοι οι οποίοι δεν μπορούν να επανενταχθούν στην αγορά εργασίας. Μιλούμε για εκατομμύρια Ευρωπαίων μεταξύ 40 και 50 ετών, οι οποίοι βρίσκονται εκτός αγοράς εργασίας και οι οποίοι δεν έχουν καθόλου την ευκαιρία να ξαναμπούν στην αγορά εργασίας και δεν μπορούν επομένως να προστατευτούν από κάποιο κοινωνικό αποτελεσματικό δίκτυο. Δεν έχουν δουλειά. Επίσης θα πρέπει να υπάρξει κοινωνική πρόνοια και προστασία με τρόπο όσο γίνεται πιο κοινό, πιο ομοιογενή. Μιλούμε για την επικουρικότητα και την αλληλεγγύη στην Ευρώπη. Οπότε και είναι σημαντικό να ξεκινήσουμε από το πώς θα το αποδείξουμε ότι υπάρχει αυτή η αλληλεγγύη και είναι αποτελεσματική. Λέμε επίσης για κάποιους ε, μισθούς που θα συνδέονται με την παραγωγικότητα. Αλλά θα πρέπει να βοηθηθεί η παραγωγικότητα, να υπάρξουν κάποια κίνητρα και να υπάρξουν αποτελεσματικές επενδύσεις ε, που να αφορούν τις μη, έψιλων, ε, τις νεοφυείς startup για τους νέους με τις καινοτόμες ιδέες και να λέμε ότι θα πρέπει να υπάρχει κάποια αναλογία μεταξύ μισθού και παραγωγικότητας ε, αυτό μου φαίνεται σαν ιδέα αρκετά περιοριστικό. Επίσης αναφέρεται η κινητικότητα. Σήμερα η κινητικότητα περνάει από κάποια, κάποιο περιορισμό γιατί θα πρέπει η κινητικότητα να είναι εθελούσια, εκούσια, να μην είναι υποχρέωση η εργασία γιατί ο κόσμος θα πρέπει να δουλεύει με αξιοπρέπεια πρώτα πρώτα και αν εγώ ως ελεύθερος πολίτης αποφασίσω να ψάξω μια ευκαιρία σε άλλη χώρα ε, τότε ε, το κάνω αυτό εκεί που θεωρώ ότι υπάρχουν περισσότερες ευκαιρίες. Αν εγώ είμαι οικογενειάρχης και είμαι υποχρεωμένος να αφήσω την οικογένειά μου και να υποχρεούμε να μεταβώ σε άλλη χώρα, αυτό δεν πάει να πει κινητικότητα. Επίσης αναφέρονται κάποιες ε, μορφές υποστήριξης, κάποιο είδους δέσμευση που αναλαμβάνει η Επιτροπή, η Ευρωπαϊκή Ένωση και κάτι το οποίο εμείς το υποσχόμαστε στους πολίτες που εκπροσωπούμε για να προστατεύσουμε ε, κάποια κοινωνικά πρότυπα τα οποία να είναι αξιοπρεπή γιατί ε, είναι αλήθεια ότι υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη φτώχεια. Είναι ενσυχητικό αυτό είναι ντροπή και όμως δεν έχουμε αρκετά στοιχεία για αυτή την φτώχεια, την απόλυτη φτώχεια. Οπότε δεν μπορεί κανείς να αρνηθεί την ύπαρξη του φαινομένου γιατί υπάρχουν κάποιες ευρωπαϊκές χώρες εκεί όπου υπάρχει πείνα και πάρα πολλοί πλήσονται εκεί από την πείνα. Άρα θα πρέπει και εδώ να είμαστε αποτελεσματικοί και να μην κάνουμε το σφάλμα το να μην αφήσουμε να ακουστεί η φωνή των πολιτών. Είναι δυνατόν να καταπιούν οι Ευρωπαίοι κάποιες άστοχες αποφάσεις. Εγώ νομίζω ότι θα πρέπει να αναλάβουμε αυτή μας την προσπάθεια εδώ, μέσω θεσμικών οργάνων, μέσω των όσων έχει υποσχεθεί το Κοινοβούλιο στους πολίτες. Άρα άνοιγμα και συνεργασία ούτως ώστε να απασχίσουμε να βρούμε τη λύση για αυτό το πρόβλημα που ε, σήμερα όλο ένα και παραξύνεται. Παρά το ότι υποτίθεται ότι αυτό έχει πλήξει λίγες χώρες, αυτές δηλαδή του Νότου. Θεωρώ ότι αργά γρήγορα αυτό πρόκειται να πάει σε όλη την Ευρώπη. Ευχαριστώ κύριε Μπαχ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να είμαι σύντομος. Θέλω να ευχαριστήσω ιδιαίτερα την Κομισιόν για την παρουσίασή της. Νομίζω ότι έχει συλλέξει τα ουσιαστικότερα στοιχεία. Η, τα σημεία έμφαση της Κομισιόν είναι οι επενδύσεις, οι διαφορετικέ αλλαγές και μια υπεύθυνη δημοσιονομική πολιτική και όλα αυτά θα υποστηρίξουν τον στόχο μιας πιο κοινωνικά δίκαιης Ευρώπης και δημιουργίας θέσεων απασχόλησης. Πρέπει όμως και τα κράτη-μέλη να κληθούν να παίξουν το δικό τους ρόλο σε εθνικό επίπεδο για να βοηθήσουν αυτό το εγχείρημα. Και πιστεύω το πιο σημαντικό είναι <clears throat> να μην χάσουμε και από τα μάτια μας τους στόχους της Ευρώπης 2020 θα πρέπει να εξασφαλίσουμε την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης, να εξασφαλίσουμε την ε, περιεκτική κοινωνία και να συμβάλλουμε στην κοινωνική Ευρώπη. Δυστυχώς, αν κοιτάξει κανείς τα, τι έχει γίνει τα τελευταία πέντε χρόνια, σε πολλά επίπεδα έχουμε απολέσει αυτούς τους στόχους και αν δεν επιτευχθούν αυτή η στόχη το 2020, ιδίω σε ό,τι αφορά την ένδια, την κοινωνική, τον κοινωνικό αποκλεισμό και την ε, ανεργία, θα είναι αυτό λυπηρό, αλλά εάν τα κράτη-μέλη συμπληρώσουν αυτές τις προσπάθειες με δικές τους ενέργειες, τότε έχουμε καλές ελπίδες να μπορέσουμε <laughs> μέσα στα επόμενα πέντε χρόνια να προχωρήσουμε προς την επίτευξη των στόχων αυτών, ώστε να τους επιτύχουμε. Χαίρομαι πάρα πολύ για την συνεργασία και με την συγκήτρια έχει πει πάρα πολλά και στη δική της ε, ε, παρουσίαση για τα οποία μπορούμε να σκεφτούμε όλοι και να προσπαθήσουμε να βρούμε κοινέ λύσεις. Και ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστώ. Η Μαρία Ροντρίγκης. Ευχαριστώ πολύ. Η ομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών θεωρεί ότι αυτή η επικαιροποίηση των κατευθυντήριων γραμμών ότι είναι πάρα πολύ σημαντική. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε κατά τη δική μας άποψη είναι να βελτιώσουμε το συντονισμό των κρατών μελών με κοινούς στόχους και επίσης να βελτιώσουμε τη δημοκρατική νομιμοποίηση και αυτό αφορά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Θεωρούμε ότι αυτή η επικαιροποίηση ήταν απαραίτητη. γιατί αυτά τα οποία υπολογίζαμε να συμβούν το 2010 έχουν ξεπεραστεί από την νέα κατάσταση που έχουμε. Γι' αυτό η Κομισιόν πολύ ορθά θέλει να ε, αναθεωρήσει τις κατευθύνες γραμμές για να μπορέσει να τις προσαρμόσει στην τωρινή ανησυχητική κοινωνική και οικονομική κρίση. Η Ευρώπη, οι στόχοι της Ευρώπης 2020 για την απασχόληση και την καταπολέμηση της ένδυας δεν έχουν επιτευχθεί κάθε άλλο. Υποχωρούμε σε ό,τι αφορά την επίτευξη αυτών των στόχων. Για όλους αυτούς τους στόχους εμείς χαιρετίζουμε την προσπάθεια να υπάρξει επικαιροποίηση των κατευθυντηριών γραμμών. Θεωρούμε ότι οι κατευθυντήριες γραμμές για την απασχόληση μπορούν να βελτιωθούν και είναι βελτιωμένες φυσικά αυτές που παρουσιάζονται σε σχέση με τις προηγούμενες. Θέλω να κάνουμε όμως μερικά σχόλια για να μπορέσουμε να ξεπεράσουμε τα προβλήματα που έχουμε στον κοινωνικό τομέα και τον τομέα της απασχόλησης αλλά και τις ανισότητες χρειαζόμαστε μια νέα επανεξισορρόπηση των κατευθυντήριων γραμμών όχι μόνο στον τομέα της απασχόλησης αλλά γενικά στον οικονομικό τομέα. Θα πρέπει να μιλήσουμε για τις επενδύσεις και αυτό φυσικά γίνεται αλλά θα πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι οι επενδύσεις συνδέονται με τις απαραίτητες μεταρρυθμίσεις σε όλες τις κατευθυντήριες γραμμές για να ληφθεί υπόψη δυνατότητα επενδύσεων θα πρέπει να τονιστούν αυτά στις κατευθυντήρες γραμμές. Ένα δεύτερο στοιχείο. Στο νέο μείγμα πολιτικών το οποίο προτείνεται από την Κομισιόν θα πρέπει να τονίσουμε ιδιαίτερα και τον ρόλο της ζήτησης Πρέπει να αντιμετωπίσουμε φυσικά την πλευρά προσφοράς με περαιτέρω μεταρρυθμίσεις και επενδύσεις. Πρέπει να αυξήσουμε όμως και την ζήτηση στο εσωτερικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τη ζήτηση για την εργασία. Ξέρω ότι λέτε ότι αυτό πρέπει να είναι η πρώτη κατευθυντήρια γραμμή και αυτό είναι θετικό. Θέλω να κάνω και ορισμένα σχόλια για τις συγκεκριμένες προτάσεις. Για την πρώτη κατευθυντήρια γραμμή για την ζήτηση του στον χώρο εργασίας. Αναφέραμε το ρόλο του ελάχιστου μισθού και αυτό είναι σημαντικό για να μειώσουμε την ένδια ιδίω την ένδυα των εργαζομένων, αλλά εκεί πρέπει να λάβουμε υπόψη και το ρόλο της ανταγωνιστικότητας. Δεν μπορούμε να δεχτούμε όμως να υπάρξει μια μείωση των, του εργασιακού κόστους ως την κύρια μέθοδο βελτίωσης της ανταγωνιστικότητας. Οι λύσεις εσωτερικής υποτίμησης που έχουν λάβει η χώρα σε πολλά κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης τα τελευταία χρόνια δεν είναι αποδεκτές. Δεύτερον, για την κατευθείαν γραμμή που αφορά την πλευρά της προσφοράς, την υπαριθμών 6, σε ό,τι αφορά την ανεργία των νέων. Φυσικά τα προγράμματα εγγύησεων για τους νέους έχουν σημασία. Να υπογραμμίσουμε όμως ότι το κύριο πρόβλημα έχουμε είναι η δημιουργία θέσεων απασχόλησης. Για την κατευθυντήρια γραμμή 7. Ναι. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε τον κατακαιρματισμό, αλλά με τέτοιο τρόπο ώστε να μην υπάρχει μία, ένας φαύλος κύκλος προς τα κάτω σε ό,τι αφορά την ποιότητα της απασχόλησης. Πρέπει να βελτιώσουμε και την ε, κινητικότητα, αλλά πρέπει να αποφύγουμε την υποχρεωτική μετακίνηση και την διαρροή εγκεφάλων που λαμβάνει χώρα ήδη σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Και το τελευταίο μου σχόλιο είναι ότι ακόμα και αν είμαστε η Επιτροπή Απασχόλησης θα πρέπει να λάβουμε υπόψη και το έργο των άλλων συναδελφών μας στην Επιτροπή Οικονομικών Θεμάτων γιατί οι οικονομικές κατευθυντήρες γραμμές περιλαμβάνουν και πάρα πολλά στοιχεία τα οποία άπτονται της απασχόλησης της αγοράς εργασίας και των μεταρρυθμίσεων στον τομέα αυτό. Πρέπει λοιπόν και οι οικονομικές και οι ε, κατευθυντές γραμμές απασχόλησης να αντιμετωπιστούν ως συνδεδεμένες. Αυτό σημαίνει πρέπει να βελτιώσουμε και τη συνεργασία μας με τους συνάδελφους της Συναδέλφους Επιτροπής Οικονομικών Θεμάτων. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε. Η Ρενάτα Βέμπερ έχει τώρα το λόγο. Άλντε, ευχαριστώ. Έχοντας ακούσει τους συναδέρφους που πήραν το λόγο πριν από μένα, αντιλαμβάνομαι ότι θα είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα διαδικασία διαπραγμάτευσης. Έχω την αίσθηση ότι δεν συμφωνούμε με μερικά από τα οποία υπόθηκαν ήδη. Ευχαριστώ και εγώ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την παρουσίασή της. Κατά τη γνώμη μου πρόκειται για τίτλους των κατευθυντηρίων γραμμών, απλώς. Γιατί ο διάβολος κρύβεται στη λεπτομέρεια, όπως ξέρουμε. Και εγώ θα ήθελα να καταλάβω πώς κάποια από τα πράγματα τα οποία τόσο ωραία μας παρουσίασε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πώς θα ερμηνευτούν στην πράξη, σε συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές που θα τεθούν σε εφαρμογή σε 28 διαφορετικές χώρες μέλη με τέτοιο τρόπο ώστε να φέρουν ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα. Αλλά φαντάζομαι ότι θα ξαναβρεθούμε κατά τη διάρκεια των διαπραγματεύσεων και ότι θα κατανοήσουμε έτσι καλύτερα τις λεπτομέρειες. Ε, δεν αμφισβητείτε το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι πολίτες περιμένουν από την Ευρωπαϊκή Ένωση κάτι πιο συγκεκριμένο. Θέλουν απασχόληση, να συνεχίσουν να έχουν δουλειά και να έχουν δουλειά ποιότητας. Μέχρι τώρα όμως έχουμε αποτύχει να αντιμετωπίσουμε την κρίση. Υπάρχει απογοήτευση λοιπόν, απογοήτευση απόλυτα κατανοητή. Mm. Όμως, έχουμε πολλές νομοθετικές διατάξεις στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχουμε και 28 διαφορετικά συστήματα. Και ακριβώς εδώ είναι που δυσκολεύομαι να κατανοήσω στην πράξη πώς θα έχουμε όχι εναρμόνιση, αλλά κάτι, εν πάση περιπτώσει, που να φέρνει τα ίδια αποτελέσματα σε όλες τις χώρες μέλη. Ελπίζω ότι η συγγήτρια ιδεολογικά θα καταλήξει σε κάτι συγκεκριμένο και ελπίζω να μπορέσουμε να συνεργαστούμε μαζί μας πάνω στις κατευθυντήριες αυτές γραμμές, ακόμα και αν το Κοινοβούλιο έχει σε βουλευτικό καθαρά ρόλο. Στο τέλος της διαδικασίας θα δούμε τι τελικά από αυτά που θα έχουμε πει θα λάβει υπόψη του το Συμβούλιο και τι όχι. Πρόεδρο, ευχαριστούμε πολύ. Η Τατιάνα Στάνοκα τώρα. Ευχαριστώ πολύ. Πρόεδρε, μια που δεν έχουμε και χρόνο, θα είμαι σύντομη. Θα ήθελα και εγώ πιο συγκεκριμένες προτάσεις και όχι αντιφατικές μεταξύ τους. Γιατί ορισμένες είναι αντιφατικές με κάποιες άλλες, ακόμα και αν βρίσκονται στην ίδια παράγραφο κατευθυντήριων γραμμών. Για παράδειγμα, για τις επιχειρήσεις, για τη μεταφορά του εργασιακού κόστους κτλ. Εμείς ως πράσινοι θέλουμε να εκφράσουμε την απογοήτευσή μας όσον αφορά τη δημιουργία πράσινων θέσεων απασχόλησης. Εξαφανίστηκε αυτό ή δεν μπήκε ποτέ. Φυσικά είναι πολύ δύσκολο να συνδυάσουμε τα πράγματα μια που προχώμαστε από διαφορετικές πολιτικές πλατφόρμες. Πάντως Είπε και η Ρενάτε ότι αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα, ότι θέλουμε πιο συγκεκριμένες κατευθυντήριες γραμμές. Ε, θα συνεχίσουμε την προσπάθεια και προσβλέπω και εγώ σε συνεργασία με την εισηγήτρια. Και θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να καταλήξουμε σε ένα καλό κείμενο. Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η Λάουρα Αγγε για να ολοκληρώσουμε τη συζήτηση αυτή. Έχετε το λόγο. Βέβαια και επαναλαμβάνω ότι είμαι διαθέσιμη να συζητήσω και να αναζητηθεί όπου είναι δυνατόν μια κοινή θέση και κάποιες συγκεκριμένες κοινέ λύσεις. Ε, εάν είναι δυνατόν να βοηθήσουμε να λυθεί το πρόβλημα της απόλυτης φτώχειας και της ανεργίας. Είναι πραγματικά προβλήματα τα οποία έχουν πλήξει την Ευρώπη μας και αυτό πλέον είναι κάτι το οποίο ε, παντού ακούγεται οπότε και θα πρέπει κάποια στιγμή να καταβληθεί μια προσπάθεια και θα πρέπει όμως να προσγειωθούμε στην πραγματικότητα των ε, προαστίων των πόλεων μας γιατί πραγματικά ε, ο κόσμος τον νιώθει στο πετσί του δεν είναι λαϊκισμός αυτό δεν είναι δημαγωγία εγώ ε, δούλευα μέχρι τον Μάιο σε κάποια εταιρεία και είδα εκεί από κοντά τι γίνεται όσον αφορά αυτούς που, που χάνουν τη δουλειά τους και ποιες είναι ακριβώς οι συνέπειες. Οπότε και εγώ ζητώ απαντήσεις πραγματικές από την Ευρώπη, από την Κομισιόν, από το Συμβούλιο, γιατί γνωρίζω την πραγματικότητα και εμείς από το κίνημα των πέντε αστέρων ε, πραγματικά θεωρούμε ότι θέλουμε να περάσει μέσα από αυτή την υπόθεση που συζητούμε τώρα η γνώμη των ε, πολιτών όλων εκείνων των πολιτών, των, τους οποίους τους εκπροσωπούμε. Μιλώ για την πραγματικότητα από την οποία προέρχομαι, γιατί γνωρίζω τα, πραγματικά προβλήματα του κόσμου. Γιατί αλλιώς δημιουργείται μια ε, αποξένωση μεταξύ εκείνων και ημών. Εγώ όμως ε, προέρχομαι από τέτοιου είδους κόσμο, από τον κόσμο που έχει αυτά τα προβλήματα και αυτό θέλω να σας μεταφέρω εδώ και θα, θα ήθελα παρακαλώ να βοηθήσουμε αυτόν τον κόσμο και να τον αφουγκραστούμε. Πρόεδρος. Ευχαριστώ. Νομίζω ότι ο καθένας έχει εμπειρία από τη δική του πραγματικότητα και όντως ε, πολλοί από μας ε, έχουμε δοκιμάσει τη σκληρότητα ε, του κόσμου Οπότε νομίζω ότι ε, η καλή συζήτηση μπορεί να οδηγήσει σε καλές αποφάσεις συνήθως, όχι πάντα. Το να δούμε το χρονοδιάγραμμα για αυτές τις ε, κατευθυντήριες συζήτηση του σχεδίου κειμένου στις 16 Τετάρτου. Προθεσμία τροπολογιών 22 Τετάρτου το μεσημέρι και κατόπιν ψήφιση στην Επιτροπή 16 Ιουνίου. Πέραν αυτών τώρα σας υπενθυμίζω ότι η επόμενη συνεδρίαση θα είναι στις 24 Μαρτίου. Αλλά εκεί θα είναι τα πράγματα πιο δύσκολα γιατί θα έχουμε και πρωινή και απογευματινή συνεδρίαση μέχρι 6.30 το απόγευμα. Οπότε προσαρμοστείτε, προσαρμοστείτε και κανονίστε τα του ταξιδιού σας. Άρα τα λέμε τότε, 24 Μαρτίου. Σας ευχαριστώ για μια τόσο ωραία συνεδρίαση. Τόσα ενδιαφέροντα. Και ελπίζω να αχθούμε σε πολύ εύστοχες αποφάσεις.